Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, συνεδρίαση. Θα συζητήσουμε την έκθεση τη κυρία Θεοχάρου και του κυρίου Γκαμπού. αιτήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Και αμέσω δίνω το λόγο την κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλουμε η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούγεται δυνατά σε μια εποχή κατά την οποία η πολυμερή συνεργασία για την ευημερία των ανθρώπων και για το καλό του πλανήτη τόσο στο πλαίσιο των δράσεων για την κλιματική αλλαγή όσο και για την αλληλεγγύη και την ειρήνη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη ως εκ τούτου είναι σημαντικό να συνεχίσουμε την πρακτική της ετήσιας έκθεσης στρατηγικής σχετικά με την εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη και για να εκπροσωπείται το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κάθε χρόνο στο υψηλού επίπεδου πολιτικό φόρουμ σήμερα η έκθεση στρατηγικής είναι ακόμη πιο επίκαιρη δεδομένου ότι η επιτροπή ετοιμάζει την κοινή συγκεφαλαιωτική έκθεση την οποία αναμένουμε σύντομα σχετικά με τη στήριξη της ευρωπαϊκής ένωσης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά την εφαρμογή της ατζέντα του 2030 με την συμβολή και των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης. Είμαστε πεπισμένοι ότι απαιτείται η προσέγγιση πραγματικά πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με ενεργό εμπλοκή του κοινού της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα σε ευρεία βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη. η στενή παρακολούθηση η αναλογική υποχρέωση λογοδοσίας και οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί επανεξέτασης που θα αξιολογούν την επιτευχθήσα πρόοδο είναι ουσιαστικής σημασίας για την βελτίωση των εθνικών στρατηγικών και την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων σε όλα τα επίπεδα η έκθεσή μα σκοπεύει να συμβάλει στην προετοιμασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη μια συνολική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2030 προς εφαρμογή των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη και για την βελτίωση τη ενσωμάτωσή του στι πολιτικέ και του μηχανισμού διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Μια στρατηγική με αναπτυξιακό χαρακτήρα με βάση την παιδεία την εξειδίκευση επαγγελματιών και την δημιουργία βασικών υποδομών μια τέτοια ευρεία κλίμακα ευρωπαϊκή πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση των πολιτικών ελλημάτων και σε εκτίμηση της απόσταση προς τους στόχους. πρέπει να καθορίζει σαφεί και διακριτές στοχεύσει, δείκτε και δράσεις που απαιτούνται για βελτίωση του πολιτικού συντονισμού και της πολιτική συνοχή για βιώσιμη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προ τον σκοπό αυτό καλούμε την επιτροπή να προβεί σε μια ει βάθο ανάλυση της ανισότητας και ανυπάρκειας των υφισταμένων πολιτικών προκειμένου να εντοπίσει κρίσιμους τομείς σε επίπεδο συνεργειών και ασυνεπιών. Κύριε Επίτροπε, βασικά θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας που θα εφαρμοστούν μέχρι το 2030 όσον αφορά πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις στατιστικές και συλλογή αναλυτικών στοιχείων διακυβέρνηση και βέλτιστες πρακτικές με στόχο την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την επιτυχία της ατζέντα 2030 ή δυνατόν πριν από το τέλος του. 2019 το γεγονό ότι πολλά κράτη μέλη και κράτη εταίροι πέραν τη ευρωπαϊκή ένωση έχουν καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε για τον σχεδιασμό μηχανισμών και στρατηγικών για την επιτυχή εφαρμογή των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη και την ενσωμάτωσή του στι πολιτικέ και στην διακυβέρνησή του είναι ένα πολύ πολύ θετικό βήμα. Εν τούτης, πρέπει να κάνουμε και άλλε βελτιώσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε τι τρίτε χώρε να ακολουθήσουν ανάλογε πρακτικέ θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου λέγοντα ότι η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να είναι παγκόσμιο πρωτοπόρο στην εφαρμογή τη ατζέντα 2030 και των στόχων για την αηφόρο ανάπτυξη σε συνεργασία με τα κράτη μέλη τη. ο στόχο μα πρέπει να είναι πάντα σταθερό η κατάκτηση τη βιώσιμη ανάπτυξη και η ευρύτερη ευημερία όλων χωρί διακρίσει χωρί ουραγού χωρί να μένει κανεί πίσω. σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και δίνω το λόγο στον κύριο Γκαμπούς. Ευχαριστώ πολύ κύρια Πρόεδρε. <clears throat> Κύριε Αντιπρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνεισηγήτριά μου, την κυρία Θεοχάρουσα και τους κοιόδης συζητητές από την Επιτροπή Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την κατανόηση και την ε, συνεργασία τους. Αυτό οδήγησε στο να καταλήξουμε σε συμφωνία για ένα θέμα πολύ σημαντικό για όλους μας, όπως είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Συζητήσαμε την αλλαγή του κλίματος και ακριβώς η δράση για το κλίμα είναι ένας από τους στόχους που θα αναθεωρηθούν το καλοκαίρι στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου των Ηνωμένων Εθνών. Οι νέε γενιέ Ευρωπαίων απαιτούν από εμά συγκεκριμένε δράσει και η ευθύνη μα είναι να ανταποκριθούν με στα αιτήματά του και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να του εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πρέπει να του εξηγήσουμε την ευρωπαϊκή επιτυχία που ήταν η COP21 με την πρώτη διεθνή συμφωνία για περιβαλλοντική ουδετερότητα. Πρέπει να του εξηγήσουμε στο πλαίσιο τη θητεία Γιούγκερ και με τον Επίτροπο Αρία Κανιέτε ε, και οι δύο από το ΕΛΚΑ και οι δύο από τη δική μου πολιτική ομάδα και με τη φιλοδοξία του Κοινοβουλίου προχωρήσαμε περισσότερο από ποτέ στον αγώνα για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Εγκρίναμε τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, αναθεωρήσαμε τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και ε, για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, για τον κοινό κανονισμό για το ηλεκτρικό ρεύμα, καταπολέμηση τη ενεργειακή στόχια. Είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε. Έχουμε τον κανονισμό για τι εκπομπέ, για τα εθνικά όρια, για τι οριακέ τιμέ. Έχουμε τι νέε εκτελεστικέ και κατεξοδότηση πράξει και από την Κομισιόνα ε, για το co-design. Για τον καθαρό αέρα έχουμε κανονισμό. Για τα πλαστικά μια χρήση έχουμε οδηγία. Τελικά έχουμε σπείρει του πόρου ε, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σπείρει την επανάσταση επανάσταση την ενεργειακή για τον 21ο αιώνα και δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε κανέναν. Σίγουρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη η κατάσταση του περιβάλλοντος. Ούτε μετριάζεται η κλιματική αλλαγή βάζοντας φωτογραφίες στο Instagram. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε ε, να προχωρούμε έχοντας ε, την επίγνωση ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και σε θέματα έρευνα ε, και ανάπτυξης για να επιτύχουμε τους στόχους μας που πρέπει να είναι όλο και πιο φιλόδοξοι. Αν υπάρχει όμως μεταγκατάσταση της βιομηχανίας δεν θα μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι ούτε από κοινωνική ούτε από οικονομική ούτε από υπερβολοντικής πλευράς. Θα πρέπει λοιπόν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης να τους θεωρήσουμε ευκαιρία. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ναι, όμως έχοντας τα πόδια στο έδαφος, πατώντας γερά όντα προσγειωμένοι, να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, να ε, καταργήσουμε ανισότητε εντό Ένωση, να καθιερώσουμε δίκαιου μισθού που θα επιτρέπουν στου εργαζόμενου να ζουν μια αξιοπρεπή ζωή και να προοδεύουν. Θέλουμε επίση του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη να του χρησιμοποιήσουμε όχι για να δημιουργήσουμε νέε δομέ, αλλά για να βελτιώσουμε τι ήδη υφιστάμενε. Το να έχουμε αστιφύλακα για, τις, ε, για του στόχου ε, δεν θα πετύχουμε κάτι καινούριο αλλαγή νοοτροπία θέλουμε, βελτίωση των μέσων αναδιανομή του πλούτου. Θέλουμε εμβάθυνση και ενίσχυση της κοινωνική οικονομίας της αγοράς Θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία ε, ώστε να υπάρχουν εισφορέ. Θέλουμε επιχειρήσει που θα έχουν την έδρα του στην Ευρώπη και όχι αλλού. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία υψηλή προστιθέμενη αξία και να μετασχηματίσουμε την οικονομία μα για να μην μείνουμε αγκυλωμένοι στο ε, παρελθόν. Όπω έλεγε και ο Ιούλιο Βέρν, δεν θέλει ο πλανήτη νέε υπήρου, ε, αλλά θέλει νέου άντρε, νέε γυναίκε. Σα ευχαριστώ. Merci beaucoup, monsieur. Κύριε Timmermans, ε, η σειρά σα να παρέμβετε σε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την ετήσιατική έκθεση του Κοινοβουλίου για τη στρατηγική για την επίτευξη του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι λεπτομερή στατή έκθεση και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί όσον αφορά την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030 και να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη θα προσανατολίσουν τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Η έκθεση είναι επίκαιρη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει τι εκλογέ που επίκυνται. Η προετοιμασία του στρατηγικού θεματολογίου για το 2019-2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμικέ προτεραιότητε για τον επόμενο κύκλο πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω διαφαίνονται στον ορίζοντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη, θέλει να πετύχει τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέλουμε να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους κατά τη διάρκεια του επομένου κύκλου πολιτικής για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που αναλάβαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο ε, προβληματισμού για τη βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 για να εμπνεύσει τη συζήτηση. Επιτάπητος έχουμε θέσει τρία ενδεικτικά σενάρια για να καθοδηγηθούν συζητήσει και πώς η εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξη μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα στην Ευρώπη και να γίνει ο σωστός των ρόλων μεταξύ ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ανώσεω και κρατών μελών. Να υπογραμμίσω κάτι, ότι αυτά τα σενάρια όλα βασίζονται επί της κοινή υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι χρειαζόμαστε ε, προσπάθεια μεγάλη στην Ευρώπη για να έχουμε βιώσιμο μέλλον και θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μέχρι το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και πέρα από αυτή την ημερομηνία. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το ερώτημα είμαστε θύματα της αλλαγή ή θα ενστερνιστούμε και θα την αγκαλιάσουμε την αλλαγή, θα την καθοδηγήσουμε. Ξεκινάμε με διάγνωση της καταστάσεως και αντιμετώπιση της πραγματικότητας και ότι θα δεχτούμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα δεν θα μπορούν να μας ανησυχούν και να μας φοβίζουν, να μας εμπνέουν, να δράσουμε τάχιστα, με αποφασιστικότητα. Λοιπόν, οι βασικοί στόχοι βιωσιμότητας για την Ευρώπη και για άλλε ε, αναπτυγμένε περιοχέ του κόσμου είναι να βρούμε τον τρόπο να αυξήσουμε την ευημερία μα και να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωή μα τον καλό, χωρί να καταστρέψουμε του φυσικού βιότοπου και να ξεπεράσουμε τα όρια του πλανήτη. Ένα μόνο πλανήτη έχουμε. Για να πετύχουμε λοιπόν ανταπόκριση σωστή τη πρόκληση, από γραμμική σε κυκλική οικονομία πρέπει να πάμε. Και θα πρέπει το σύστημα τροφίμων να είναι βιώσιμο και θα πρέπει να είναι πράσινη η ενέργειά μα, η κινητικότητα και τα κτίρια. Για να γίνει αυτό, πρέπει όλε τι πολιτικέ μα να εφαρμόσουμε, όλα τα εργαλεία μα προ την επίτευξη των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παιδεία, ε, έρευνα, καινοτομία, επιστήμε, η ψηφιοποίηση, επίση η χρηματοδότηση, η φορολόγηση, η τιμολόγηση, και υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και εμπορευματική πολιτική προφανώ. Και οποιαδήποτε μετάβαση πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαια και να μην μένει κανένα πίσω. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα χωρί κοινωνική βιωσιμότητα. Και για να είμαστε αυτοί που είμαστε στην Ευρώπη, όλε οι δράσει θα πρέπει να σέβονται πλήρω το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώ και το να καλύπτονται όλοι, να συμπεριλαμβάνονται όλοι και να έχουμε στοιχεία με τα οποία, στα οποία βασιζόμαστε. Α προχωρήσουμε τώρα με πεποίθηση, με αισιοδοξία η Ευρώπη είναι το καλύτερο μέρο στον κόσμο που μπορεί να ηγηθεί ε, για τι μεταβατήσει αυτή τη ε, βιώσιμης. Έχουμε τη δεξιότητα, τα μυαλά, τον κόσμο είναι η καλύτερα στεδεμένη ήπειρο και η βιωσιμότητα έχει βαθιέ ρίζε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Του επόμενου μήνε θα πρέπει να καταλήξουμε συμφωνία σχετικά με το πώ και τι πρέπει να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω την επόμενο κύκλο πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέταξε έκθεση, όπου ευνοεί το πρώτο σενάριο που παρουσιάστηκε στο έγγραφο προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει γενική στρατηγική των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη που θα καθοδηγούν τι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη και αυτά θα πρέπει να αποφασίσουν. Αυτό θα βοηθήσει την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαράξει πορεία σαφή για την ανάπτυξη ενό μια πλήρου στρατηγική στην εφαρμογή των στόχων βιομηχανικού ανάπτυξη. Μια στρατηγική που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είπα στην αρχή τη εβδομάδα στο, άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ότι και στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την εργασία μα, οι στόχοι τη βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι το τέλειο πλαίσιο για το πώ θα κατανείμουμε τι εργασίε και τα καθήκοντα και θα ασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τα σωστά βήματα προ μια βιώσιμη ανάπτυξη, βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη. Η συλλογική συνεισφορά για, όσον αφορά την πλατφόρμα, την πολυεπίπεδη που ασχολήθηκε με την επιχειρήση στην Ευρώπη μέχρι τη ζωή των πουλιών, δείχνει σαφώ ότι περιμένουν οι λαοί μα μια φιλόδοξη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη αυτή. Και θέλω να κλείσω λέγοντα Ας μην το μετατρέψουμε σε μια διαμάχη αριστεράς και δεξιάς. Είναι ένα θέμα που είναι σημαντικό για όλο το πολιτικό φάσμα στο Κοινοβούλιο και πάντα έτσι αισθανόμουν ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για αυτό το λόγο από το Κοινοβούλιο για τους στόχους αυτούς και πιστεύω ένθερμα σε αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν την εκπροσώπηση των ομάδων με τον κύριο Πέτερλε που έχει το λόγο για ένα λεπτό εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω έμφαση στο λεπτό που έχω στην υγεία, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υγεία. Και οι δύο συνεισηγητές, ένας από τον οποίων ε, φυσικός, έχουν συζητήσει το μάλλον οι γιατρός, ε, έχουν συζητήσει το ζήτημα της ε, υγείας. βέβαια η υγεία είναι μια διάσταση η οποία καλύπτει πολλούς τομείς ε, της ζωής μας. Είναι τα πράγματα αρκετά ανησυχητικά εξού και θα πρέπει διάφορες στρατηγικές, ε, τομεακές ε, να ενταχθούν σε μια γενικότερη στρατηγική που θα είναι το, ο βασικός μοχλός. Αν έχουμε περισσότερους καρκινοπαθείς διαβητικούς και άλλους στον πλανήτη μας, πώς θα πετύχουμε τους στόχους. Οι στατιστικές είναι γνωστές, θα ήθελα πιο μεγαλύτερη φιλοδοξία για όλους. Ευχαριστούμε εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, κυρία Σλάιν, δύο λεπτά. Συνάδελφοι, υπάρχει μεγάλη αντίφαση μεταξύ τη αίθουσα αυτή που είμαστε ελάχιστοι και στι πλατείε στην Ευρώπη όλοι, όπου αύριο χιλιάδε νέοι θα κατέβουν στου δρόμου για να διαμαρτυρηθούν, για να προσελκύσουν την προσεχή μα ε, για το κλίμα και κατά της αλλαγή του κλίματος ε, που απειλούν το μέλλον μας και κατά των ανισοτήτων που εξακολουθούν να έχουν καταστροφική συνέπεια όσον αφορά την συνοχή και την ευημερία τη ευρωπαϊκή κοινωνία. Και εκείνοι κατάλαβαν ότι η μάχη για τη δικαιοσύνη την περιβαλλοντική γίνεται μαζί με εκείνη για την κοινωνική δικαιοσύνη. Και σε αυτή την αίθουσα και η πολιτική πρέπει να είμαστε στο ύψο τη Γκρέτα Τούμπερ και των άλλων νέων, στο ύψο αυτών. Θα τι χρειάζεται για να εφαρμόσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030. Τρία πράγματα που δεν βλέπω. Χρειάζεται θάρρος, πολιτική βούληση και επαρκή πόρη. Θα χρειαζόταν ένα μεγάλο Green New Deal επενδύσεων για να καταφέρουμε να συνοδεύσουμε την οικολογική μετάβαση που είναι απαραίτητη για την οικονομία μας. Και δεν είναι μόνο θέμα να διασώσουμε τον πλανήτη, αλλά και να δημιουργήσουμε απασχόληση ποιοτική και ποσοτική, διότι τα δύο πράγματα θα πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Λοιπόν, από όταν είμαστε στη Νέα Υόρκη για την έγκριση του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, εμεί ζητούσαμε και ζητούμε και με την έκθεση σημερινή επιτέλους να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική εφαρμογή των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ κρατών μελών και με επαρκή ε, παρακολούθηση για την επίτευξη των στόχων. Με το έγγραφο προβληματισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε την ευκαιρία να κάνει ένα βήμα προόδου αναφερόμενη σε αυτού του είδους την κατεύθυνση και περιοριζόμενη να παρουσιάσει τρία σενάρια σαν να ήταν ίσα τα ενδεχόμενα. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσουμε τι προσπάθειε. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πρέπει επιτέλου να έχουμε τη στρατηγική και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθοδηγήσει την υλοποίηση των στόχων σε παγκόσμιο επίπεδο και να δείξει συνοχή όσον αφορά τι πολιτικέ τη εσωτερικέ και εξωτερικέ. Ξεκινώντα από τον προπολογισμό, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και από το οικονομικό εξάμεινο. Έχουμε τεράστια ευθύνη έναντι των νέων που αύριο και αυτού του μένε έχουν βγει στι πλατείε και δεν μπορούμε να υπολοιπούμεθα αυτή τη αντίδραση. Ευχαριστώ. Εν ονόματι των σοσιαλιστών, ο κύριος Ότς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να βασίζεται σε μία βασική αρχή. Πρέπει να βελτιώνουν το επίπεδο ζωής των κοινωνιών και τώρα και στο μέλλον και όχι να μεγιστοποιούν τα έσοδα για τους λίγους. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα είναι ουραγός. Θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και ε, στα θέματα της οικολογίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν κερδοφορία. Θα πρέπει να ε, προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Ισορροπία λοιπόν, ενδυνάμωση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η καλή διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η επιχειρηματικότητα, η γεωργία, η περιβαλλοντική προστασία και καλύτερη προστασία της υγείας, ισορροπημένη ε, διαχείριση των αποβλήτων, μείωση της φτώχειας και της ανεργίας, όλα αυτά είναι τα βασικά στοιχεία είναι συγκοινωνούνται δοχεία η υγεία των ανθρώπων και η ευημερία τους με την ισορροπία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βεκάπερα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη καθορίστηκαν πριν από τέσσερα χρόνια και έχουν γίνει πολλά για την επίτευξή του, αλλά ακόμη απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν και δεν μπορώ λίγα παραδείγματα να σας δώσω. Πολύ λίγα έχουν φτάσει στο στόχο του 0,7% αναπτυξιακής βοήθειας. Δεύτερον, ε, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι σε καλή σειρά κατάταξης όσον αφορά ε, ε, τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων και οι ανισότητες έχουν αυξηθεί, δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι θα πρέπει να κατανοήσουμε το πόσο καθολική είναι η στόχη των βιώσιμης ανάπτυξης. Χρειάζεται συνοχή της πολιτικής σε όλους τους τομείς. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να μεταβούμε σε κλιματική ουδετερότητα, γιατί όλα αυτά ε, παίζουν ένα ρόλο κλειδί για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη η Επιτροπή έχει καθυστερήσει όσον αφορά μια στρατηγική που πρέπει να δημιουργηθεί για να επιτευχθούν όλα αυτά. Και το έγγραφο προβληματισμού που μας έχει δώσει η Επιτροπή πρέπει να το επικροτήσουμε. Χρειαζόμαστε να πάρουμε την πρώτο καθεδρία σε όλα αυτά. Έχει αρχίσει η συζήτηση και για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε καινούργια επιτροπή, καινούργιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη μα του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη σε όλα τα επόμενα προγράμματα. Ελπίζω το Μάιο ε, στην διάσκεψη κορυφή να ληφθούν τα κατάλληλα, οι κατάλληλε αποφάσει για το μέλλον τη Ευρώπη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους εισηγητές για αυτή την έκθεση για την ετήσια στρατηγική έκθεση. Πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει για την ε, διάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2019 τονίζονται στο κείμενο οι προσπάθειες, οι μεγαλύτερες προσπάθειες που απαιτούνται και από τα κράτη-μέλη και από την Επιτροπή. Στο πλαίσιο τη στρατηγική μα για το 2030 θα πρέπει όλε οι ευρωπαϊκέ στρατηγικές να κινητοποιηθούν και να υπάρχει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση ε, στη διακυβέρνηση σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030. Δεν αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τα εφιστάμενα εργαλεία και του εφιστάμενου δείκτε. Χρειαζόμαστε μια αλλαγή μοντέλου. Χρειάζεται ε, στόχοι και κατευθύνες γραμμέ, να μπουν σε όλε τι πολιτικέ με συνεπεί δείκτε και σημεία σύγκριση και ένα πλαίσιο παρακολούθηση όλες ε, οι αποφάσεις ε, για τα έσοδα και οτιδήποτε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα και αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν για να τα επιτύχουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Χάζεκαμπ εκ μέρου τη Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε η κοινωνία, η οικονομία, <clears throat> το καταναλωτικά μοντέλα πρέπει να αλλάξουν αν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο πλανήτη στο μέλλον. Και είναι θετικό που έχουμε συμφωνίες σε ό,τι αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, στο πλαίσιο του ΙΕ, αλλά πρέπει να περάσουμε τα λόγια στις πράξεις. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή, δεν υπάρχει ε, πλανήτης Β. Έχουμε χιλιάδες νέους που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Αντί να πάνε σχολείο, ε, πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα. Και έχουμε τις γεωργικές ε, πολιτικές που αν παραμείνουν παραδοσιακές θα δημιουργήσουν πρόβλημα και στην ε, βιοπικιλότητα και στην ασφάλεια των τροφίμων. Βλέπουμε επίσης ε, και τι συμβαίνει με το ζωικό κεφάλαιο, με τις διάφορες ζωνόσους, άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τα παραδοσιακά μοντέλα, δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα αν ο ίδιος δεν αλλάξει. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε νοοτροπία, θα πρέπει να παράγουμε λιγότερο κρέας και να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας μεταξύ άλλων. Οι καταστροφικές πολιτικές της Ένωσης πρέπει να αλλάξουν άρδιν τώρα. Εξού και θεωρώ πως θα πρέπει να καταργηθεί και η Ευρωπαϊκή Γεωργική Επιδότηση, για επιδοτήσεις γενικώ του χέρια 1,5 λεπτό από την ομάδα ENF. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για βιωσιμότητα εδώ στο Κοινοβούλιο, πάντα εξετάζουμε την περιβαλλοντική διάσταση. Θέλω να αναφερθώ στη βιωσιμότητα της κοινωνίας και του πολιτισμού. Διότι αυτά είναι τα στοιχεία που δέχονται πιέσεις έξωθεν λόγω μετανάστευσης, κυρίως από τις Ισλαμικές χώρες που δεν μοιράζονται τον πολιτισμό μας και δεν θέλουν να προσαρμοστούν, που έχουν τη δική τους κουλτούρα, που θεωρούν ότι είναι ανώτεροι και οποίοι είναι εχθρικοί προς το δικό μας πολιτισμό και εκ των ένδων. Τα αριστερά κόμματα, τα οποία πάντα μιλάνε για πολιτισμό και για ταυτότητα και θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά σαν το κλειδί κατανόησης των κοινωνιών μας. Αλλά ο πολιτισμός και η κοινωνία μας είναι στο επίκεντρο του θέματος. Αν υπονομευθούν, τότε όλος ο οργανισμός θα πρόκειται τελικά να μαραθεί και να χαθεί. Μιλάμε για βιωσιμότητα, αλλά ας μιλήσουμε για τον πολιτισμό και την κοινωνία, διότι πρέπει και αυτά να είναι βιώσιμα. Η συνέχιση ύπαρξης του τρόπου ε, ζωής του δυτικού, η επιβίωση των δυτικών κοινωνιών. Και αυτό αφορά τη βιωσιμότητα ε, που εδράζεται επί της ε, ιουδοχριστιανικής ρίζας, που είναι κάτι γνωστό για μας και θα πρέπει να διατηρηθεί. Ο κ. Σόνικ έχει το λόγο για ένα λεπτό η έκθεση είναι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου, η πρώτη έκθεση που υποβάλλεται στα πλαίσια του ΟΗΕ που αφορά την ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Πέρα από τον ε, τις προαιρετικές εθνικές εκθέσεις. Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας μόνο μέσω ολιστικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις στρατηγικές στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, καθώς και στους μηχανισμούς διαχείρισης, σύμφωνα με το σενάριο παριθμό 1 που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο προβληματισμού του Ιανουαρίου. Γι' αυτό είναι σημαντικότατο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση κενών όσον αφορά τις πολιτικές στρατηγικές και την υλοποίηση αυτών και να διαπιστώσει τους τομείς όπου ακόμα δεν επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταλή για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαστε παραμονή μια ακόμη πορεία ε, κατά τη κλιματική αλλαγή και στη Μάλτα, τη χώρα μου. Οι ε, σπουδαστέ κινητοποιούνται, αλλά δεν είναι μόνο η νέα γενιά που κινητοποιείται. Αφορά ε, και το μέλλον μα, αλλά όλου μα και το παρόν όλων μα. Ε, η θερμοκρασία θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 1,5 βαθμού μέχρι το 2030, αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα. Η αύξηση κατά 1,5 βαθμού τη θερμοκρασία θα οδηγήσει σε αύξηση τη στάθμη τη της θάλασσας κατά 3 με 4 μέτρα. Θα πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε αυτό τι σημαίνει για τις παράκτες περιοχές, για τους ανθρώπους που ζουν σε νησιωτικές περιοχές όπως στη χώρα μου, δίπλα στη θάλασσα ή για ε, χώρες ε, που είναι χαμηλή, χαμηλό, το υψόμετρο. Πρέπει να το σκεφτούμε. Έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, βιομηχανία 4.0 που μας λένε ότι είναι για την ε, ψηφιοποίηση, τον αυτοματισμό. Εγώ όμως, ε, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω, θα πρέπει να είναι για τις οικολογικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και τώρα είναι η στιγμή να αλλάξουμε ε, παράδειγμα, να κάνουμε στροφή. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι οι οικονομίες μας να ανθίσουν, να αναπτύξουν. Το παραδοσιακό μοντέλο ε, δημιουργεί προβλήματα. Ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι προτεραιότητα για αυτό το μοντέλο. Πρέπει όμως να έχουμε φιλοδοξία ε, και να θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο, να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο σε ό,τι κάνουμε, ώστε να έχουμε ένα εξασφαλισμένο μέλλον για τους νέους μας, για τις οικονομίες μας. Θετικός μετασχηματισμός που πρέπει να ξεκινήσει από τις χώρες, αλλά να πάρει ε, και δόθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εκπαίδευση, την ασφαλή των τροφίμων, την καταπολέμηση της και Και στι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη ε, αυτό ακριβώ ε, αποσκοπούν να πετύχουν ε, περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. Να είναι εξασφαλισμένε για το μέλλον. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, θα πρέπει να παραμείνουμε σε αυτό το ρυθμό ώστε να έχουμε εξασφαλισμένο μέλλον για τις κοινωνίες μας. 1,5 λεπτό τώρα ο κύριος Γερμπράντη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω για τα ευγενικά του λόγια τον Επίτροπο. Πολύ ωραία λόγια πράγματι. Αλλά με τα ωραία λόγια δεν ε, φτάνουμε και απαραίτητο στα έργα, αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Δύο πράγματα για να είναι ξεκάθαρα αυτά που θέλω να πω. Στόχοι 14 και 15 η ζωή κάτω από το νερό και η ζωή ε, στη ξηρά. Έχουμε τη στρατηγική για την βιοπικιλότητα. Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε έναν υδροφόρο ορίζοντα υγιή. Αν δεν εφαρμοστεί η στρατηγική από την Κομισιόν, τίθεται σε κίνδυνο η ζωή στον πλανήτη. Τους στόχους όμως που τους έχουμε και εμείς οι ίδιοι διατυπώσει στη δατική για τη βιοπικιλότητα είναι σαφές ότι δεν θα τους εφαρμόσουμε γιατί έχουμε προθεσμία δύο ετών. Έχουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Λένε όλοι οι δείκτες είναι στο κόκκινο. Πολλές μελέτες επίσης ε, κάνουν λόγο για εξαφάνιση εντόμων. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τι κάνει η Κομισιόν, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και ακόμη χειρότερα ό,τι έχει να κάνει με τα οικολογικά ζητήματα τα παρακάμπτουν, τα αποφεύγουν. Θα εξαντληθεί το φυσικό κεφάλαιο. Τι θα κάνει η Κομισιόν, αυτό είναι το ερώτημά μου. Τι θα κάνετε, θα σκάψετε ακόμη περισσότερο τον ε, τάφο μας ή θα αντιδράσετε. Η κυρία Χάουτελα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο προβληματισμού τη Επιτροπή δείχνει ότι οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να διαπνέουν όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε στρατηγικές βιωσιμότητας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα παραδοτέα για το 2030, τα οποία θα έχουν και χρονικού ε, περιορισμού. Η πολιτική θα πρέπει να ε, ε, λαμβάνεται ε, με διαφορετικό τρόπο μέσα σε όλες τις πολιτικές και για όλα τα θέματα και θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσανατολίζεται προς την επίτευξη των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης όλοι οι τομεί τη πολιτική από την γεωργία μέχρι τη βιομηχανία, από τι μεταφορέ μέχρι την απασχόληση και όλοι οι ενδιάμεσοι τομεί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και να συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεσή του δείχνει ότι θέλουμε να το επιτύχουμε, να έχουμε δηλαδή νέου τρόπου θέσπιση πολιτική. και θέλουμε να συμμετέχουμε στο ανώτατο, στο φόρουμ, ε, στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επίπεδου και είναι σημαντικό να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να εξετάσουμε με τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο κ. Τίμερμανς που ανέφερε την υπεύθυνη συμπεριφορά επιχειρήσεων που θα είναι σημείο κλειδί. Κύριε Χάουτελα, δέχεστε να απαντήσετε σε μια ερώτηση του κυρίου Στιουαρτ. Παρακαλώ, ναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Χάουταλα τι κάνει η ίδια προσωπικά τώρα για να βοηθήσει το περιβάλλον. Ε, από τι παρετήστε. Και δεν μιλώ για επιδοτήσεις στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή στους λαμπτήρες LED. Αλλά τι κάνετε, δεν οδηγείτε αυτοκίνητο, δεν χρησιμοποιείτε αεροπλάνο, δεν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, δεν τρώτε κρέας, δεν έχετε κατοικίδια. Από τι έχετε παρετηθεί, κάτι που να σας κοστίζει προσωπικά. Καταπληκτική ερώτηση, ερώτηση, λέει η κυρία Χάουτελα. Μπορώ να σας πω, ναι μου, ότι το 1974 συνίδρυσα ένα χορτοφαγικό εστιατόριο και την ίδια γραμμή έχω ακολουθήσει σε όλη μου τη ζωή. Η κυρία Σάντσεφ Καλντεντέ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Σεπτέμβριο θα ε, γίνει η πρώτη συνάντηση των ε, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ε, για να εξολογηθεί πρόοδο του θεματολογίου 2030. Είναι τότε η στιγμή για να κλείσουν τα κενά στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Πολιτική συνέπεια για την ανάπτυξη πρέπει να είναι εμφανή σε όλου του τομεί, όλα τα επίπεδα. Όμω, ο ελέφαντα στο δωμάτιο λέγεται εμπορική πολιτική. Θα πρέπει οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη να έχουν μια εγκάρση διάσταση φύλου και θα πρέπει να είναι οι αρχέ που θα διέπουν την γεωργική, αλληλευτική, καταναλωτική μα πολιτική και φυσικά θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με του στόχου του θεματολογίου. Η πρόοδο μέχρι στιγμή είναι ανεπαρκή. Αυτό είναι σαφέ και το ίδιο θα συνεχίσει να ισχύει εάν αφήνουμε ταμπού ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα. Γιατί αντί να επενδύουμε δι ε, στη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, δεν μιλάμε για κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Παραδείγματο χάρη, έχουμε το στόχο τη ε, μηδενική πείνα. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε για την ε, κυριαρχία την διατροφική και να πάψει να υπάρχει κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια για τα τρόφιμα. Μιλάμε για τέλος στην φτώχεια. Πρέπει να πάψει ε, ο ακραίος πλούτος ταυτόχρονα. Όταν μιλάμε για υγεία και ευημερία θα πρέπει να διορθωθούμε τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση της υγείας και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θέλουμε το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης. Πρέπει όμως να αναζητήσουμε την ισορροπία γιατί είναι πεπερασμένος ο, πόρη του πλανήτη πρέπει λοιπόν παρότι είναι σεξι να μιλάμε για διάσωση των καταπιεσμένων, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που τους καταπιέζουν αρχικά και να τους βάλουμε ε, αντίσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το θεματολόγιο του 2030 βασίζεται στη δημοκρατία, τη συμμετοχή, τη διακυβέρνηση, σωστή κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, βιωσιμότητα και σεβασμό του κράτου δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό Ευρωπαϊκή Ενώση των κρατών μελών και σε όλο τον κόσμο. Το θεματολόγιο του 2030 είναι ζωτική σημασία για να πετύχουμε καλύτερη ευημερία για όλου και να δίκαιο κόσμο και να μην αφήνουμε κανέναν πίσω. Και είναι τέσσερι κεντρικοί πυλώνε βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και διακυβέρνηση, πρέπει να εφαρμοστούν. Λοιπόν, οι συνθήκε, οι δίκε για μια οικονομία με χαμηλό άνθρακα που θα καλύπτει όλου είναι σημαντικό κομμάτι αυτού. Καλωσορίζω αυτή την έκθεση που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μια φιλόδοξη στρατηγική για την εφαρμογή του θεματολογίου του 2030. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό επίση να τονίσουμε τη σημασία τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Και τέλο θέλω να πω ότι κάθε κράτο μέλο θα πρέπει να δεσμευθεί να δώσει 0,7% σαν αναπτυξιακή βοήθεια, κάτι που ζητήσαμε και χαίρομαι που το δικό μας κοινοβούλιο είπε ότι η Ιρλανδία θα το κάνει αυτό. Το είπε ο Λοιπόν, ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Γκραπίνη θα ξεκινήσει. Έχουμε τρεις που θέλουν να μιλήσουν. Ναι, εσείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Προέδρε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπη. Η σημερινή ανάλυση δείχνει ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κάνουμε μια δελεχή ανάλυση των πολιτικών που διαθέτουμε. Έχουμε αποτελέσματα ή όχι. Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των λαών. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών και αν πράγματι η οικονομική προσπάθεια και η δουλειά που κάνουμε στο Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν ε, οδηγήσει σε μια εκρίζωση της φτώχειας και σε καλύτερα εισοδήματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στη διαχείριση μία ανάλυση προϋποθέτει και διορθώσεις των πολιτικών αν αυτές δεν είναι σωστές. Γι' αυτό το 2030 πρέπει να δούμε ότι δεν είναι πολύ μακριά. Πρέπει συνεπώς να λάβουμε υπόψη τις απομακρυσμένες ζώνες και να λάβουμε υπόψη επικουρικότητα και αναλογικότητα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε καλωσορίζουμε την έκθεση για την ε, εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι σημαντικό το ότι υπάρχει ετήσια έκθεση για να μπορούμε να παρακολουθούμε την πρόοδο και κυρίως να διαπιστώνουμε κατά πόσο οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί μπορούν πραγματικά να δρομολογηθούν και νομίζω ότι οι στόχοι όπως αναφέρθηκαν είναι σημαντικοί στηρίζονται κυρίως στην δημοκρατία στην αλληλεγγύη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το βασικό στοιχείο φυσικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρώτα απ' όλα είναι να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας γιατί είναι δυνατόν να έχουμε ανάπτυξη χωρίς θέσεις εργασίας. εμείς θέλουμε ανάπτυξη με θέσεις εργασίας και κυρίως πρέπει να γίνει η ανάπτυξη αυτή με τέτοιο τρόπο που να αξιοποιηθούν οι πόροι να αξιοποιηθούν οι πόροι για τους ίδιους τους λαούς ιδίως για τους λαούς του αναπτυσσόμενου κόσμου προκειμένου να χτυπηθεί η φτώχεια και να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν και οι μεταναστευτικές ροές από τον αναπτυσσόμενο κόσμο προς την ευρώπη και θα μπορέσει έτσι να εμπεδοθεί η δημοκρατία και στην ευρωπαϊκή ένωση και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. ευχαριστώ. Ε, ε, ε, και τέλο ο κ. Καπούτο, πρόεδρε βιωσιμότητα και μετάβαση προ την οικονομία με αντίκτυπο ουδέτερο για το κλίμα, κυκλικό και που καλύπτει όλου, είναι θεμελιώδη σημασία για να εγγυηθούμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μακροπρόθεσμα. Το θεματολόγιο 2030 μπορεί να μα κάνει να το πετύχουμε αυτό, καθορίζοντα φιλόδοξου στόχου παγκόσμιου ε, που θα είναι διασυνδεμένοι μεν με του δε. Όμω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καθορίσει μια παγκόσμια στρατηγική, γενική στρατηγική για την υλοποίηση του θεματολογίου του 2030, που συμπεριλαμβάνει στρατηγικού στόχου εσωτερικού και εξωτερικού Ευρωπαϊκή Ενώσεω με ε, χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030 και με στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, όπω το γενικό πλαίσιο που θα πρέπει να είναι για του προσανατολισμού που θα ακολουθήσουμε μετά το, που έχουν καθορίσει το 2017. Χρειάζονται μεγάλε προσπάθειε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κρατη Χρειάζομαστε μια στρατηγική γενική που είναι, διατρέχει όλες τις πολιτικές και είναι σε πολυεπίπεδη εφαρμογή διακυβέρνησης. Δεν αρκούν τα μέσα που έχουμε, χρειάζεται να αλλάξουμε και παράδειγμα και σενάριο, χρειάζεται ένα αποτελεσματικό ε, πλαίσιο εποπτείας. Το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να προσανατολίζεται περισσότερο προς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο δρόμος που έχουμε να κάνουμε δεν είναι απλός, αλλά θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε για τις νέες γενιές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομο κατστιά ήταν και ξανά προ εσά απευθυνόμαστε κύριε Τίμερμαν, και έχετε και πολλές ερωτήσεις να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώντα σε κάποια από τα σημεία που ελέγχθησαν, θέλω να πω ότι έχουμε μια τεράστια ευκαιρία για να κάνουμε ακριβώ αυτό που είπε τώρα ο κ. Καπούτο, δηλαδή να οργανώσουμε αυτή την αλλαγή μοντέλου. Όταν ε, μίλησα και στους Υπουργούς ε, Γενικών Υποθέσεων ε, αυτή την εβδομάδα, ένιωσα ότι όντως κάτι αλλάζει και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Κοινοβούλιο αυτό με την Νέα Επιτροπή θα έχουν μια τεράστια ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δραστηριότητες των επομένων πέντε ετών χρησιμοποιώντας τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Αρχίζει να υπάρχει και όλο και μεγαλύτερη συνένεση στα κράτη-μέλη προς κάτι τέτοιο. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση αυτοί που αρνούνται σε γενικές γραμμές την κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι σε διάφορες ε, τυχές του πολιτικού φάσματος που αρνούνται την κλιματική αλλαγή. Αυτοί που πιστεύουν ότι θα έπρεπε ε, να τρεφόμαστε με, με χορτάρι ε, πρέπει να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να περάσει αυτό το κλίμα εκφοβισμού. Πρέπει να έχουμε υψηλά επίπεδα ευημερίας χωρίς να χρησιμοποιούμε τον πλανήτη σαν να έχουμε και άλλους δύο ανταλλακτικού πλανήτες. Υπάρχει τρόπος να επιτύχουμε στην πολιτική μας αυτή. Το θέμα είναι ότι όσο περισσότερο περιμένουμε, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να ενστερνιστούν αυτή την ιδέα κοινωνίες μας είναι να μπει η κοινωνική ευθύνη στο προσκήνιο. Και συμφωνώ με τον κύριο Μαριά που είπε ότι θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι στο μέλλον έχουν βιώσιμες επιλογές με βιώσιμους και αξιοπρεπείς μισθούς και κοινωνική προστασία. Αν ε, νιώθουν ότι θα τους βάλουμε σε σπηλιές να τρώνε χορτάρι, δεν θα δώσουν την πολιτική υποστήριξη που χρειαζόμαστε για να κινηθούμε προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προς τον κύριο Γκέρμπραντι θέλω να πω ότι αν ε, πιστεύετε ότι αυτά που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλονται στη δική σας επιμονή, με τα χαράς να σας το παραχωρήσω. Η Σκακέλε είπε πρόσφατα σε κάποια συναντήση ότι η καλύτερη νομοθεσία οδήγησε σε μείωση των ε, προδιαγραφών. Νομίζω ότι η θέσπιση καλύτερη νομοθεσία μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε την άποψη των ε, Ευρωπαίων πολιτών δεν θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε ε, τους πολίτες αν δεν είχαμε τη διαβούλευση ε, για την οδηγία για τη φύση για να μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα τη φύση. Μας βοήθησε λοιπόν η θέσπιση καλύτερης νομοθεσίας και για την στρατηγική για το πλαστικό. Το ξέρει ο κύριος Γκεμπράντη, είναι μοναδική η στρατηγική μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κινούμεθα ε, με την ταχύτητα του φωτό για την κυκλική οικονομία. Και ο κύριος Κατάινεν έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και αυτό θα είναι προ όφελο όλων μα στο μέλλον. Όλοι οι φόβοι που υπάρχουν στην αρχή ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε χαμηλότερε προδιαγραφέ, σε χαμηλότερε φιλοδοξίε δεν ισχύουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινήθηκε προ τα μπρο ε, με μεγάλη ταχύτητα μάλιστα. Και τώρα, ε, άλλο ένα θέμα για την βιωσιμότητα. Τα πολιτικά κινήματα που προσπαθούν να περικόψουν τι τις πολιτιστικές ε, επιδοτήσεις, γιατί λένε ότι αυτά είναι για τις ελίτ, είναι τα ίδια κινήματα που μας ζητάνε να κρατήσουμε και να διατηρήσουμε ε, τον πολιτισμό, ε, που είναι υπέρ της πολιτιστικής βιωσιμότητας. Για μένα ο πολιτισμός δεν είναι ένα μέσο για να αποκλείσουμε κάποιους. Τα πολιτιστικά μας θέματα είναι αυτά που μας δίνουν περηφάνεια για αυτό που είμαστε, που αναπτύσσουν την περιέργειά μας για τους άλλους. Χωρίς την, το φιλοπερίεργο αυτό πνεύμα και την κριτική σκέψη δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και αυτοί που θέλουν να μας κάνουν εχμαλώτους ενός πολιτισμού και να φοβόμαστε τους άλλους πολιτισμούς, απλώς θα σκοτώσουν αυτό το φιλοπερίεργο πνεύμα και δεν θα μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στου συζήτητε, ξεκινώντα από την κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον επίτροπο τίμερμανς για την εμπνευσμένη πρωτομιλία του και για τις απαντήσεις καθώς επίσης και τον συνάδελφο καμπούς και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεισφορά τους θα συμφωνήσω ιδιαίτερα με τον κύριο πέτερλε ότι η υγεία είναι βασική παράμετρος της ανάπτυξης. δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς υποδομές υγείας και δεν μπορεί να υπάρξουν υποδομές υγείας χωρίς εκπαίδευση γιατρών μεών νοσηλευτών τεχνητών δασκάλων. η παιδεία συνεπώς είναι ο ισχυρότερος μοχλός για την ανάπτυξη νομίζω ότι πολλά από όσα έχουν λεχθεί από τους συναδέλφους είναι ενσωματωμένα στις προοπτικές αυτής της έκθεσης. εμείς θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς υπαναχωρήσεις και παλινοδίες. βασική βέβαια προϋπόθεση είναι η διάθεση του 0,7 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των κρατών μελών προς τον σκοπό αυτό. σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ Κύριε εσείς για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κομισιόν, θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου όσους έλεγαν το λόγο στη σημερινή συζήτηση θα ψηφίσουμε και στι 12 το μεσημέρι. Ελπίζω και η συζήτηση και η ψηφοφορία να μα εμψυχώσει, να μα δώσει περισσότερη ελπίδα για να έχουμε μια ουδέτερη εκπομπές κοινωνία. Αλλά το στόχο αυτό θα τον πετύχουμε εάν μα συνοδεύσουν και άλλοι φορεί. Αλλιώ δεν θα έχει και τόσο νόημα. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ηγετική θέση και είναι σε ηγετική θέση σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων του θεματολογίου 2030. Όμως ε, δεν σημαίνει ότι αν είμαστε γρήγοροι θα φτάσουμε πιο γρήγορα στο στόχο, όπως μας δείχνει και ο μύθος ε, της χελώνας και του λαγού. Ε, διότι πρέπει να του πετύχουμε πραγματικά του στόχου. Το είπε και χθε ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτε, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο που θα προκύψουν από τι επερχόμενε εκλογές θα είναι η υπεύθυνη, το είπατε και εσεί, κύριε Τίμερ, για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Για πολύ σημαντικές αναθεωρήσεις όπω τι οδηγίε πλαισίου για τα είδωτα που σχετίζεται με το στόχο 6 του θεματολογίου 2030. Δεν είναι όμω μόνο το έργο τη Κομισιόν ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και διακυβέρνηση πολυεπίπεδη, διότι είναι περιορισμένε οι αρμοδιότητε μα εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει να οργανώσουμε διάλογο και συμμετοχή του, του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου και η ε, εξωτερική πολιτική πρέπει επίσης να ε, κάνει το δικό ε, να παίξει το δικό της ρόλο. Πρέπει να ακούσουμε όλες τις φωνές και τις πιο ασθενείς και τις πιο μικρές, γιατί όλοι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την ένωση. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι κλειδί. Αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αίσθηση του ανήκει σε αυτό το ειρηνευτικό εγχείρημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να περάσουμε στο τι έχουμε κάνει στην Ευρώπη, όχι στο τι θα κάνουμε. Και ολοκληρώνοντας, ε, έχετε δίκιο κύριε Αντιπρόεδρε, δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς. Είναι ένα θέμα Ευρωπαίων ε, και είναι θέμα επιθυμίας να είμαστε ηγέτες. Και πραγματικά αυτό, γι' αυτό έχουμε εμείς την ευθύνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε η δεξιά. ειναι ενα θεμα ευρωπαιων και ειναι θεμα επιθυμιας να ειμαστε ηγέτε. και πραγματικα αυτο γι αυτο εχουμε εμεί την ευθυνη ευχαριστω προεδρος ευχαριστω εδω ολοκληρωθηκε η συζητηση και θα ψηφίσουμε αργότερα σήμερα. Η μερίσια διάταξη τώρα προβλέπει Ε, Προβλέπει τη συζήτηση τη έκθεση του κυρίου Φιέλνε σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων και θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Φιέλνε, συζητητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Το ελεύθερο εμπόριο είναι από του καλύτερου τρόπου για να βγουν από τη φτώχεια οι χώρε. Το αποδεικνύει αυτό με ακρίβεια ιστορία. Α πάρουμε την Ολλανδία, επί παραδείγματι αναπτύχθηκε όταν οι πολίτες της έγιναν ε, ελεύθεροι, είχαν ελεύθερο εμπόριο το 17ο αιώνα και στη χώρα μου στη Σουηδία ξεκίνησε 100 χρόνια ανάπτυξη τη δεκαετία του 18, που ξεκίνησε το 1870 όταν άνοιξε το εμπόριο. Και αυτά δεν είναι μόνο στο παρελθόν. Η Κορέα και τώρα η Κίνα δεν θα είχαν τη θέση που έχουν εάν δεν είχαν ε, ενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και περί αυτού πρόκειται το σύστημα γενικών προτιμήσεων. Το γενικό σύστημα λοιπόν αυτών προτιμήσεων θα έλεγα ότι είναι η κορονίδα τη εμπορική πολιτική Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Τη προσπαθεί να συσχετήσει τι φτωχέ χώρε με την παγκόσμια οικονομία και να τι βγάλει από την φτώχεια. Πολλέ χώρε στον κόσμο έχουν αυτού του είδου τα προγράμματα, αλλά εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το πρόγραμμά μα. Είναι άκρο γενναιόδωρο και δίνει αξία και περικοπές στις ταρίφες, συγγνώμη στους δασμούς που έχουν νόημα στους δικαιούχους και είναι πολύ γενναιόδοροι για τις πιο φτωχέ χώρες στον κόσμο με πρόσβαση χωρίς ποσοστό ή χωρίς δασμούς στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για όλα τα προϊόντα πλην όπλων. Το καλύτερο κομμάτι, το καλύτερο τμήμα του συστήματος γενικών προτιμήσεων είναι το GSP+. Το GSP χορηγεί και άλλες προτιμήσεις συμπληρωματικές στις χώρες εκείνες που κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια, που προσπαθούν να συμπεριφερθούν καλύτερα εφαρμόζοντας, κυρώνοντας και υλοποιώντας 27 διεθνείς συμβάσεις από θέματα διακυβέρνησης στο, περιβάλλον και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και αυτό είναι ένα εργαλείο για να δώσει περαιτέρω κινήτα στις χώρες, ούτως ώστε να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι βιώσιμος και θα ωφελεί όλους τους πολίτες. Είναι ένας τρόπος να εξασφαλίσουμε το ότι γίνεται σεβαστή η ορθή διακυβέρνηση. Τώρα φτάνουμε στα μέσα του προγράμματος και αρχίζουμε να βλέπουμε τι μπορεί να βελτιωθεί, τι θα έπρεπε να βελτιωθεί και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζει και η έκθεση. Καταρχάς, πρέπει να διευκολύνουμε τις δικαιούχες χώρες να μπορούν να έχουν ε, πηγές και από άλλες χώρες και θα πρέπει οι κανόνες προέλευσης να αλλάξουν για να φύγουμε από αυτό το μπέρδεμα που έχουμε τώρα. Ε, το πρόγραμμα αφορά τη διευκόλυνση των χωρών να ενταχθούν στα παγκόσμια συστήματα προσθήκης αξίας στα προϊόντα και όχι το αντίθετο. Δεύτερον, θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνουμε την επιτόπια παρακολούθηση και εδώ όλοι μπορούν να βοηθήσουν. Η κοινωνία των πολιτών, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, διάφοροι φορείς του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, πρεσβείες κλπ. Μετά θα πρέπει να εντάξουμε και τι υπηρεσίε στο Γενικό Σύστημα Προτιμήσεων, ώστε να μπορούν να έχουν ποικιλομορφία οι χώρε στην προσέγγιση του και να μπουν και σε αυτό το τομέα. Υπάρχει προηγούμενο με ε, τις υπηρεσίες ε, για την εξαίρεση υπηρεσιών για τι λιγότερο χώρες. Θα πρέπει να να θέσουμε σωστέ προτεραιότητες για να μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω την ανάπτυξη, αλλά υπάρχουν και κάποιε φωνέ που απειλούν αυτή την προσέγγιση. Καταρχά θα έλεγα υπάρχουν οι φωνέ εκείνε που θέλουν να επιβάλλουν πολλέ απαιτήσει στις δικαιούχε χώρε. Αν βάλουμε πολλέ απαιτήσει όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, προστασία περιβάλλοντο και επιβάλλουν σε αυτές τις χώρες αυτό, ίσω τελικά ε, να είναι επιβλαβέ για τι φτωχότερε. Δεν είναι Νορβηγία αυτέ οι χώρε. Αν ήταν Νορβηγία θα χρειαζόταν αυτό το εργαλείο. Είναι καλύτερο να είναι κάποιο λιγότερο φτωχό και καταπιεσμένο, παρά είναι ακόμα φτωχότερο και ακόμα περισσότερο καταπιεσμένο. Μετά έχουμε ένα άλλο παράδειγμα προστατευτισμού, το δεύτερο. Δηλαδή ότι φοβόμαστε τι αγωγέ από τι φτωχότερε χώρε και δυστυχώ η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει να θέσει δάσματα σε ρύζι από την Καμπότζη και το Μιανμάρ είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αντικατοπτρίζει φόβους αυτή η έκθεση και ελπίζω ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα εξετάσει το θέμα του νέου προγράμματος γενικών προτιμήσεων και δεν θα ακούσει ε, τις φωνές που θέλουν να, να απειλήσουν αυτό το σύστημα ε, που χρησιμοποιεί το εμπόριο για ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Κύριε Μίμητσα, έχετε το λόγο εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ε, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές ε, αξίζουν τις ευχαριστίες μας για το χρόνο που έχουν επενδύσει και για την προσοχή που έδωσαν στην έκθεση αυτή για την εφαρμογή του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων φτάνει σε μια στιγμή που αξιολογούμε τις επιπτώσεις ε, και την αποτελεσματικότητα του υφιστάμενου κανονισμού για τις γενικευμένες προτιμήσεις και τι βελτιώσεις μπορούμε να επιφέρουμε στο διάδοχο σχήμα. Από το 1971 έχουμε σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος στόχος, όπως τέθηκε στην αρχική ρήτρα του ΠΟΕ, ήταν να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να μειώσουν τη φτώχεια και να ενσωματωθούν στην παγκόσμια οικονομία. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετασχηματιστεί αρκετές φορές στο πέρασμα του χρόνου. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων έγινε το 2012 με τρει βασικούς στόχους. Πρώτον, να συνεισφέρουμε στην εξάλληψη της φτώχειας, αυξάνοντας τις εξαγωγές από τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό έγινε με σημαντική μείωση του αριθμού των δικαιούχων, εστιάζοντας τις προτιμήσεις στις περισσότερο ευάλωτες οικονομίες. Δεύτερον, να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και τη χρηστή διαχείριση και διακυβέρνηση με μεγαλύτερη ε, ορατότητα και ελκυστικότητα για το GSP+, ε, με συνδέοντάς το και με βασικές διεθνείς συμβάσεις για τα εργασιακά δικαιώματα, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστής διακυβέρνησης. Και βεβαίως και καλύτερη προστασία των οικονομικών ε, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο μηχανισμός διασφάλισης ε, φροντίζει να γίνει το σύστημα αυτό περισσότερο προσβάσιμο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Τώρα μετά από τα πρώτα χρόνια εφαρμογή αυτού του συστήματο, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνούν σε γενικέ γραμμέ με την αξιολόγηση ότι ο κανονισμό για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ε, επιτυγχάνει αποτελεσματικά του στόχου του. Οι ε, εξαγωγέ από τι πιο ευάλωτε οικονομίε έχουν αυξηθεί σημαντικά και αυτό μπορεί να συνεισφέρει στην εξάλληψη τη φτώχεια. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και ιδίω το GSP Plus ε, συνεισφέρει θετικά στην προώθηση των ε, εργασιακών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφωνούμε με την άποψή σας ότι η εμπορική πολιτική συμπεριλαμβανομένου και του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων, πρέπει να είναι κομμάτι του συστήματο των Ηνωμένων Εθνών ε, και θα πρέπει να είναι υπέρ των βασικών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε δημοκρατία, κράτο δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα. Η εμπορική πολιτική δεν μπορεί από μόνη τη να το κάνει αυτό, ούτε απομονωμένα φροντίζουμε με μεγάλη προσοχή να εξασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματος χάρη, διασφαλίζουμε το διάλογο για το GSP Plus ε, και το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις χώρες ε, δικαιούχους, ώστε να ενισχύει ο ένας διάλογος τον άλλον. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα να οθούμε προς μεγαλύτερη πρόοδο. Ε, της εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων παρατηρούμε πρόοδο σε όλες τις ε, χώρες δικαιούχους. Παραμένουν βέβαια αρκετά προβληματικά ζητήματα και θα συνεχίσουμε να προσέχουμε ε, πάρα πολύ τις ε, χώρες δικαιούχους μένοντας σε στενό διάλογο με αυτές. Θέλω να θίξω και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας και συγκεκριμένα τη διαφάνεια στην εμπορική πολιτική για την υλοποίηση του κανονισμού γενικευμένων προτιμήσεων κάνουμε σημαντική προσπάθεια να εξασφαλίσουμε δράσεις βιώσιμες και διαφανείς. Διαβουλευόμαστε με την κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις δικαιούχους χώρες και μάλιστα σε τακτική βάση. Πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα οποία έχουν να συνεισφέρουν, τα οποία αξιολογούμε με μεγάλη προσοχή. και προσπαθούμε ε, να λαμβάνουμε υπόψη τη θέση τους, ε, ακούγοντας ε, τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, ακόμη και αν πάντοτε δεν καταλήγουμε στα ίδια συμπεράσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τις ευθύνες της για θέματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι δράσει μα όσον αφορά την Καμπότζη και τη Μιανμάρ καταδεικνύουν αυτή τη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ω προ αυτό, συμφωνώ μαζί σα ότι η απόσυρση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων πρέπει να είναι η έσχατη λύση στην οποία θα καταφύγουμε. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, τώρα ξεκινάμε με ένα νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί όταν ε, ε, λήξει το εφιστάμενο σύστημα προτιμήσεων ε, τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Η γενική μας εκτίμηση είναι ότι λειτουργεί σωστά και από αυτό το σημείο φετηρία θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Η έκθεση και το ψήφισμά σα περιλαμβάνουν αρκετές προτάσεις τις οποίες θα εξετάσουμε με προσοχή. Το επόμενο άμεσο βήμα για τη μελλοντική μας πορεία είναι να κάνουμε μία αξιολόγηση επιπτώσεων ε, η οποία θα μας καθοδηγήσει για το έργο μας για το νέο κανονισμό GSP. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει και ευρία διαβούλευση με τους πολίτες και προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κύριος Μπράντο Μπενιφέη, εκ μέρους της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατίας δεν μπορεί να θεωρείται σαν κάτι δεδομένο. Πρέπει να ενισχύεται με κάθε διαθέσιμο μέσο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό προθητή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στον κόσμο. Οι εμπορικέ πολιτικέ θα πρέπει με τη σειρά του να εγγυώνται την υποστήριξη αυτών, την παγίωσή του. Μέσω του GSP Plus στι ευάλωτε χώρε επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγουν αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλει να σέβονται 27 ε, συμβάσει για, το, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και το εμπόριο. Είναι σημαντικό μοχλό για υποστήριξη τη δημοκρατία και βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι δικαιούχε χώρε. Σε κάποιε περιπτώσει όμω, παρά τι σοβαρέ παραβιάσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναστείλει την προτιμησιακή αντιμετώπιση. Άρα χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι διαδικασίε διαβούλευση και να υπάρχει εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση των δικαιούχων χωρών. Να καθορίζεται σαφώ ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του όλου συστήματο που, αν ξεπεραστούν, συνεπάγονται την αναστολή του, γενικού συστήματος, συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων. Ευχαριστώ εκφραστούν οι ομάδε. Με το ΕΛΚ ξεκινάμε τον κύριο Φίσα, που έχει, τον κύριο Φίσα που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες με τις πλέον ευάλωτες οικονομίες στον κόσμο. Όπως δείχνει και η έκθεση του συναδέλφου Φιέλνερ, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων έχει ε, φέρει οικονομικά ωφέλη σε αυτές τις χώρες. Ε, βοήθησε τις εξαγωγές του, βοήθησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύστημα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο για την προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καλή διακυβέρνηση, την προστασία του περιβάλλοντο ε, στι δικαιούχου χώρε. Δεν θα πρέπει όμω να ξεχνούμε πω σε ορισμένε περιπτώσει η αύξηση των εξαγωγών ε, δημιούργησε και ανεπιθύμητε παρενέργειε για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την κοινωνική ανάπτυξη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω Ω προ αυτό, πως οι εμπορικέ προτιμήσει θα πρέπει να συνοδεύονται με την τήρηση των διεθνών συμφωνιών και μεταρρυθμίσεων, ώστε τα προγράμματα του συστήματο γενικευμένου προτιμήσεων να μην συνοδεύονται από περιβαλλοντικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Ροντρίγε Πινιέρο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Εγώ υποστηρίζω στεναρά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο της εμπορικής πολιτικής για την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στη λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η κατάργηση δασμών στις χώρες αυτές με αντάλλαγμα την προστασία των εργασιακών περιβαλλοντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της χρηστή διακυβέρνησης φυσικά και οδήγησε σε καλύτερη απασχόληση και μας επέτρεψε να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα της παιδικής εκμετάλλευσης, της διαφθοράς Βοήθησε επίση στην καταπολέμηση τη φτώχεια. Δεν αρκούν όμω οι πρόοδοι αυτέ. Και δυστυχώ αυτό που βλέπουμε είναι σημαντική οπισθοδρόμηση σε ορισμένε εξ αυτών των χωρών. Έξω και είναι σημαντική η μεταρρύθμιση και χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που ο εισηγητή έδειξε ότι και όπω και ο Επίτροπο ότι θα δεχθούν ε, τι ε, τροπολογίε. Διότι πρέπει να θεωρήσουμε ότι έσχατη λύση είναι η άρση αυτών των προτιμήσεων, εάν δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν γίνονται σεβαστές οι δεσμεύσεις. Πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ε, υποστήριξη των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε σε λιγότερο προηγμένες χώρες που εκμεταλλεύονται ε, την χαμηλότερη προστασία περιβαλλοντική και ε, εργασιακή να δίνεται δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να εξάγουν με πολύ χαμηλότερους δασμούς τα προϊόντα τους ε, στις χώρες που εφαρμόζουν υψηλότερα πρότυπα. Πρέπει να βελτιώσουμε τη ρύθμιση, να εμβαθύνουμε σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί μεν, αλλά πρέπει να βελτιωθεί ως προς την εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν βλέπω τον ε, εκπρόσωπο των συντηρητικών, οπότε θα περάσουμε στην Άλντε και στην κυρία Σχάκη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συνάδελφοι, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων είναι ένα παράδειγμα του πώ χρησιμοποιούμε την οικονομική μα δύναμη, ούτω ώστε να ρίξουμε το βάρο μα και να επηρεάσουμε και να επιφέρουμε αλλαγέ για του φτωχού στι φτωχότερε χώρε. Και η έκθεση που εθετούμε σήμερα δείχνει πω το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ευνοεί του δικαιούχου μα, έχουν αυξήσει τι εξαγωγέ του πολύ σημαντικά προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω αυτού του είδου η προτιμησιακή πρόσβαση δεν πρέπει να θεωρείται σαν κάτι δεδομένο. Συνδέεται με σαφεί προποθέσει, παραδείγματο χάρη όσον αφορά τη βελτίωση τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Και μετά την συμπεριφορά του, την καταπιεστική του ηγέτη τη Καμπότζη του Χομσάν, η Επίτροπο η κυρία Μάλστρομ ξεκίνησε διαδικασία ούτω ώστε να αποσυρθούν τα δικαιώματα τη Καμπότζη στα πλαίσια του σχήματο Τα Πάντα Πλην Όπλων. Αυτή είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη κίνηση που θα πρέπει να στηρίξουν τα κράτη-μέλη και οι επίτροποι και η ύπατη εκπρόσωπο σε όλε τι ε, συναλλαγέ με την Καμπότζη. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε δευτερόλεπτο για να ξεκινήσουμε και άλλη διαδικασία για το Μιανμάρ διότι συνεχιζόνται οι δολοφονίε, συστηματικέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυλακίσει δημοσιογράφων και όλα αυτά δεν πρέπει να του δίνουν το δικαίωμα για εμπορικέ προτιμήσει. Ένα σύστημα το οποίο απολαμβάνει τώρα Μιανμάρ. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το σύστημα γενικευμένων προϊόντων με έναν καλό και οργανωμένο τρόπο και έτσι να μεγιστοποιούμε τον αντίκτυπο που έχουμε και την επιρροή στον κόσμο. Ευχαριστώ. Εν ε, της, των Πρασίνων, η κυρία Χάουτα, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το, το εργαλείο το, του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων μπορεί να εξασφαλίσει ε, το εμπόριο και την ανάπτυξη. Αλλά η αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού έχει αμφισβητηθεί διότι δεν βελτιώνει απαραίτητα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και δεν προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα απαραίτητα. Πιστεύω ότι η προσέγγιση ε, η ξεκάθαρη διαπόσυση όλων των δασμολογικών προτιμήσεων από μια χώρα δεν είναι κάτι αποτελεσματικό. Έχουμε τέτοιο παράδειγμα όπως το Μιανμάρ και την Καμπότζη. Και νομίζω ότι θα πρέπει οι επιλογές να αυξηθούν. Πιστεύω ότι αντί ε, θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο ορισμένου οικονομικού τομεί μέσα αυτού του εργαλείου, όχι γενικά την οικονομία, και να είναι στοχευμένε οι κυρώσει κατά των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή άλλες υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει να μπορούμε να βάζουμε εταιρείε ή εξαγωγή σε μαύρη λίστα που καταχρώνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβιάζουν τα ανθρωπίνα δικαιώματα. Επίτροπε, θα έχετε ένα σύστημα καταγγελιών για θύματα ε, που είναι, αυτούς που είναι θύματα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα πλαίσια του GSP+. Ο κύριος Σόλτσεν ονόματι της ΓΚΟΕ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε Φιέλνερ, μιλάμε για το ελεύθερο εμπόριο, μιλάμε για το ε, εμπόριο σύμφωνα με διοντολογικό ύφο και νομίζω ότι παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα θετική εικόνα. Πριν από πέντε χρόνια, στην προηγούμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων, παρά ισχυρή κριτική από τη δική μα πολιτική ομάδα και από την κοινωνία των πολιτών, διαγράφησαν από τον κατάλογο προτιμήσεων όλε οι χώρε που σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα είχαν επιτύχει κάποιο μεσαίο εισόδημα. Σήμερα μόνο 8 χώρε αποφελούνται από το GSP. Θα πρέπει το κριτήριο τη φτώχεια να το αντικαταστήσουμε με το κριτήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα πρέπει να δείξει ότι τη αποσύρει τη δασμολογική ελάφρυνση όταν υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στην περίπτωση της Καμπότζης και της Μιανμάρ θα πρέπει να ξεκινήσει να γίνει άμεσα αυτό και θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία για τις Φιλιππίνες. Το 2022 λύγει ο υφιστάμενος κανονισμός και η μεταρρύθμιση ζητάει από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή να λάβουν μέτρα για την εμπορική πολιτική μετά τις εκλογές άμεσα. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ε, ομάδα EFTD, η κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το εμπόριο για να βοηθήσουμε τι αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά θα πρέπει να προστατεύσουμε και τι ευρωπαϊκέ ευαισθησίε και να εμποδίσουμε να έχουμε νέα περίπτωση όπω το σχετικού ρυζιού. Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούνται οι φτωχέ χώρε σαν τεράστιε εκτάσει καλλιέργεια. Θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση και να, έχει, να, να αναπτυχθεί η βιομηχανία ε, και υπηρεσίε σε τοπικό επίπεδο. Χρειάζονται κοινωνικέ ρήτε. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε στι πολυεθνικέ, τι ευρωπαϊκέ, να μετακαθίστανται εκτό Ευρώπη για να παράγουν εκεί που εκμεταλλεύονται του εργαζόμενου για ελάχιστα ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό εγώ υποστηρίζω την ιδέα μέτρων διαφύλαξη όχι μόνο για τα γεωρικά προϊόντα ή τα βιομηχανικά, αλλά και για το σεβασμό των κοινωνικών και περιβαλλοντικών ε, ε, δικαιωμάτων θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι ρήτρε αυτέ διαφύλαξη να εφαρμόζονται άμεσα. Στην περίπτωση του ρυζιού χρειαστήκαμε πέντε χρόνια. Στο μέλλον πρέπει να είμαστε πολύ μα πολύ πιο γρήγοροι. Αλλιώ θα την πληρώσουν τελικά και οι Ευρωπαίοι συνέπειε. Για το ΕΝΕΦ, e η κυρία Ζανέτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 40 χρόνια τώρα δίνουμε αυτές τις προτιμήσεις στις θεσμολογικές αναπτυσσόμενες χώρες μετά τη διάσκεψη του ΛΟΜΕ για να ευκολύνουμε δήθεν την ανάπτυξή του, βοηθώντα να μπουν στο παγκόσμιο εμπόριο. Μετά τα 40 χρόνια έχουμε παταγώδη αποτυχία. Όλοι οι δείκτε ανάπτυξη δίνουν αποτελμάτιση και υπαναχώρηση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ο μηχανισμό τελικά προσπαθεί, υποτίθεται ότι προσπαθεί να συμμαζέψει αυτού που χρησιμοποιούν του εργαζόμενου σαν σκλάβου. Σε μια συνεδρίαση με την πρεσβεία τη Μπαγκλαντέ, με σχετικισμό, μας μετά μια πυρκαγιά που έγινε σε εργοστάσιο χημίας που είχαν δεκάδες ε, νεκροί είπαν ότι υπάρχουν παντού πυρκαγιές και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες μας είπαν. Σε χίλια εργοστάσια και αποθήκες χημικές στην πρωτεύουσα του Καπατέλς 850 κτίρια είναι παράνομα και δεν πληρούν προδιαγραφές και οι διευθυντές ε, μα κορυδεύουν οι ηγέτε αυτών των χωρών και δεν βλέπουν από το σύστημα ότι παρά μόνο σύστημα που μπορούν να απομυζήσουν χρήματα. Είναι απο, αναποτελεσματικό, δαπανηρό, καταστροφικό για άνδρες, γυναίκε και παιδιά και τα δικαιώματά του. Και κυρίω οικονομικά είναι παράλογο το σύστημα αυτό. Ολοκληρώσαμε τους, με του εκπροσώπου των ομάδων. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Το, γενικό, το σύστημα γενικών προτιμήσεων είναι ένα από τα τρία ε, σχήματα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προσφέρει στι αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι λογικό να ενθαρρύνει κανεί αναπτυσσόμενε χώρε να ενταχθούν στο παγκόσμιο εμπόριο. Πράγματι και εγώ ίδιο ε, ε, είχα ετοιμάσει μανιφέστο που μιλούσε για περάσπιση το εμπόριο αντί τη βοήθεια. Τα ωφέλη που απορρέουν από το εμπόριο πιθανότατα να διαρκέσουν πολύ περισσότερο από εκείνα που απορρέουν από μια ενίσχυα, από μια βοήθεια που χορηγείται. Όμω, και είναι ένα τεράστιο όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί αυτά τα συστήματα για να προωθήσει το δικό της πολιτικό θεματολόγιο. Δεν το λέω μόνο εγώ αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια, ο Επίτροπος για το Εμπόριο, ευρωβουλευτέ συνάδελφοι υπήρξαν σαφέστατοι από αυτού και πράγματι διαφανεί θα έλεγα ήταν υπερήφανοι όπως και ο Μεσάκερ νωρίτερα σε μια άριστη ομιλία. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, η Σρι Λάγκα ποτέ δεν ήταν πλούσια χώρα και υπέφερε πάρα πολύ από το τσουνάμι του 2004. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα μετά από αυτό απέσυρε το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν ε, από τη Σρι για καθαρά πολιτικούς λόγους. Με μία λέξη, αυτή η δράση ήταν μια δράση εκδικητική και δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τέλος, Λανσίνη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σύστημα γενικών προτιμήσεων ε, είναι μια μείωση τασμών για τις αναπτυσσόμενες χώρες, μια βοήθεια στην προσπάθεια να φτάσουν, να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτές τις χώρες. Υπάρχουν ελλείψεις όσον αφορά τη μηχανισμούς ε, για την προστασία του περιβάλλοντος, κυρίως στην παραγωγή και στη φαντουργία κυρίως σε αυτές τις χώρες. Πρέπει να, προγραμματι... να υπογραμμίσω ότι υπάρχουν και στρεβλώσεις στην αγορά από την αναγνώριση. Ε, ε, υπάρχει, μια, υπάρχει μια ρήτρα διαφύλαξης ε, όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Όπως και το είδαμε με το ρίζι του Μιανμάρ και της Καμπότζης, οπότε τις διαδικασίες κόστον Ιταλία ζημιές και πολλή δουλειά, πέντε χρόνια. Είναι πολύ περίπλοκες και ελάχιστε διαφανείς οι διαδικασίες που καταρτίζουν τον κατάλογο για τις χώρες που μπορούν να είναι δικαιούχες ε, μπορούν να υπάρχουν προσθήκε, αφαιρέ κλπ. Αν θέλει η Ευρώπη να βελτιώσει τι συνθήκε των εταίρων του που είναι κοντά και μακριά και να υποστηρίξει την ανάπτυξή του, χρειάζεται να κινηθεί συνεκτικά. Δεν μπορεί να επιβάλλει κανόνε όλο και πιο αυστηρού που είναι ει βάρο των επιχειρήσεών μα και να, ε, και να είναι ευνοϊκό για αυτούς που δεν σέβονται τα περιβαλλοντικά δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των εργαζομένων εκτός Ευρώπης. Κύριε Μαριά, είσαστε ο μόνος αγορητής του Catch the Eye. Έχετε το λόγο, κύριε Μαριά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων με τη μείωση δασμών προχώρησε προκειμένου υποτίθεται να στηριχθεί ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Όμως αυτό που είδαμε ήταν ότι κατά κύριο λόγο αξιοποιήθηκε από τις πολυεθνικές, οι οποίες με το outsourcing βρήκαν φτηνά εργατικά χέρια στον αναπτυσσόμενο κόσμο εκεί όπου δεν τηρείται καμία προδιαγραφή ούτε για την προστασία της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων ούτε για μισθούς ούτε βέβαια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. και αυτό που πρακτικά συμβαίνει είναι να υπάρχει ένα κοινωνικό ντάμπινγκ. ουσιαστικά παράγονται φτηνά προϊόντα μέσα στις αναπτυσσόμενες χώρες τα οποία εισάγονται χωρίς δασμούς στην ευρωπαϊκή ένωση και στους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι και ένας αθέμητος ανταγωνισμός. άρα επί του πρακτέου όλο αυτό το σύστημα αντί να βοηθήσει τους ίδιους τους εργαζομένους επί της ουσίας τους έχει μετατρέψει ακόμα σε πιο φτωχούς στις αναπτυσσόμενες χώρες και το μόνο που έχει κάνει είναι να αυξάνει τα κέρδη των πολυεθνικών εις βάρος και των εργαζομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατσιά. Ο κύριος Μίμητς, ο Επίτροπος, έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και την ε, συνεισφορά σας σε αυτή τη συζήτηση. Πράγματι παραμένουμε ε, προσιλωμένοι στο ότι η εμπορική πολιτική από κοινού μάλιστα ευρωπαϊκές πολιτικές ε, θα δώσει προτεραιότητα στον ε, σεβασμό των ε, θεμελιωδών οικομενικών αξιών. Και γι' αυτό και το σύστημα γενικευμένων Προτιμήσω ένα σημαντικό εργαλείο εμπορική πολιτική που έχει σχεδιαστεί για τι αναπτυσσόμενε χώρε, τι οποίε βοηθά ε, να έχουν περισσότερε εξαγωγέ. Ε, οι δικαιούχε χώρε ωφελήθηκαν γιατί πολύ μεγάλο αριθμό ε, υπηκών του βγήκε από τι συνθήκε τη φτώχεια. Έχει βοηθήσει επίση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μαζί με την ΕΕΔ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να έχει σταθερή ε, στάση απέναντι στο θέμα αυτό με τις δικαιούχες χώρους. Θα εξετάσουμε τις δυνατές βελτιώσεις στον κανονισμό και θα λάβουμε υπόψη πολλά από τα δικά σας αιτήματα και πολλές από τις δικές σας προτάσεις ώστε να συνεχιστεί το σύστημα αυτό γενικά με προθυμίσεων και να είναι μια δύναμη καλού. και σας ευχαριστούμε που δίνετε μεγάλη προτεραιότητα στο Ευρωκοινοβούλιο στην εμπορική πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Φιέλνερ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την πολύ καλή συζήτηση. Δύο βασικές τάσεις ε, βλέπω σε αυτή τη συζήτηση. Αφενός ε, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι δεν βλέπουμε την ανάπτυξη που θα θέλαμε και θα τους παρακαλούσα να διαβάσουν ε, τι στατιστικές. Αυτοί που μιλάνε για τελμάτωση, ότι δεν αναπτύσσονται οι φτωχότερε χώρες, διότι η ουσία είναι ότι ποτέ μα ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε τόσους λίγους ανθρώπους που να ζουν σε απόλυτη ένδυα, σε απόλυτη φτώχεια. και αυτό ε, το χρωστούν ε, στην ε, ένταξή του στην παγκόσμια οικονομία. Δεύτερος τομέας, πάνω στον οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή, είναι τι κάνουμε με όσους δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει. Κάποιοι εδώ δίνουν την εντύπωση ότι δεν κάνουμε τίποτε. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα η Σρι Λάνκα είναι ένα παράδειγμα που η χώρα αυτή, αν δεν συμπεριφερθεί σωστά, χάνει τι προτιμήσει τη Και με τη Μιανμάρ κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει όμω να έχουμε κατά νου το εξή. Όταν εκδιώκεται μια χώρα από το σύστημα, το σύστημα πάβει πλέον αποδίδει. Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι βλέπουμε αλλά και τι δεν βλέπουμε. Στην ιστορία, στα βιβλία της ιστορίας διαβάζουμε αυτά που έχουν συμβεί, αλλά δεν βλέπουμε αυτά που δεν συνέβησαν λόγω πιέσεων, λόγω διαλόγου, λόγω και του εργαλείου αυτών προκειμένου. Εγώ λοιπόν θα έλεγα ότι ε, θα βελτιώσουμε ε, τη βιωτικό επίπεδο και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παραμένοντας το σύστημα, αφήνοντας τις χώρες στο σύστημα, γιατί αν τους διώξουμε χάνεται αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό ζητώ από τους συναδέλφους να είμαστε σκληροί, κατηγορηματικοί και αυστηροί απέναντι στην παρακολούθηση, αλλά να μην τιμωρήσουμε τους ήδη καταπιεσμένους, κάνοντάς τους ακόμα πιο φτωχούς και ε, εκδιώχνοντάς τους από το σύστημα. Πρώτα πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε κάθε διάταξη του και δυνατότητα μας δίνει ο κανονισμό για να πιέσουμε προς μια καλύτερη εφαρμογή. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε στη συνέχεια. Περνάμε ε, στη ε, συζήτηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρχίζουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν και την κυρία Χάουταλα που είναι μία από τις συντάκτριες. Κυρία Χάουταλα. Mettez votre micro, <laughs> um, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με την επιδεινούμενη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προτύπων της δημοκρατίας στο Καζακστάν. Είναι μια χώρα, βλέπετε, που έχει υπογράψει διευρυμένη συμφωνία σύμπραξη και εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένα ευρύ πλαίσιο για τον ενισχυμένο πολιτικό διάλογο ε, και σίγουρα το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες και αρχές της οικονομίας της αγοράς και βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα πολιτικών διώξεων, πολιτικοί κρατούμενοι, βασανιστήρια στις φυλακές και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράσουμε όσον αφορά την επιδείνωση της καταστάσεως. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κατάσταση των ακτιβιστών των συνδικάτων. Αναφέρω δύο ονόματα. Στο κοινό μας ψήφισμα αναφέρονται. Νούρμπα Κουσοβάιφ και Αμίν Ελοίζνοφ που απελευθερώθηκαν με εγγύηση τον Μάιο του 2018 άρα του τους απαγορεύεται στηριότητα η συνδικαλιστική. Αυτό είναι δυνατόν με μια χώρα που έχει διευρυμένη αυτή η συμφωνία ε, εταιρική σχέση. Ο κύριος Μάκερ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το θέμα αυτό ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Το 2015 ε, ολοκληρώσαμε την ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με το Καζακστάν, όπου σημαντικά κεφάλαια είναι αυτά που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Όμως ε, πολλές φορές ε, ε, έχουμε μαρτυρίες από πολίτες του Καζακστάν που καταγγέλουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει εκφοβισμός, βασανιστήρια, παράνομες κρατήσεις το καθεστώς Ναζερβάγεφ έχει περιστήλει τα δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ατόμων που έχουν διωχθεί ή συλληφθεί. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν ε, ε, επισκεφθήκαμε το Κοινοβούλιο του Καζακστάν ε, όχι, ως αντιπροσωπεία στο Καζακστάν, δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς, γιατί δεν τους επέτρεπαν την πρόσβαση. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας, λέει η Πρόεδρος. Ο Σόλτ, Σόλτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ένα από τα βασικά διδάγματα ε, της ε, πτώσης ε, της σοσιαλιστικής, του σοσιαλιστικού αθεστώτος πριν από 30 χρόνια. Για να εγγυηθούμε τα δικαιώματα χρειαζόμαστε το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Αυτό είναι το κυρίαρχο, διότι η δημοκρατία και η δυνατότητα συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία ανάπτυξη κοινωνία θα πρέπει παντού να έχουν το προβάδισμα. Γι' αυτό είναι λυπηρό που τα τελευταία χρόνια η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στο Καζακστάν έχει επιδεινωθεί ιδίως γιατί υπάρχει νομοθεσία σχετικά με τον εξτρεμισμό που χρησιμοποιείται για την δίωξη των πολιτικών αντιπάλων. Έχουμε αρκετές μαρτυρίες που δείχνουν ε, ότι ε, οι πολίτες ε, θέλουν ένα πιο δημοκρατικό τρόπο διακυβέρνησης της κοινωνίας τους και νομίζω ότι θα πρέπει να καταδικάζουμε κάθε τέτοια δράση ε, πολιτικά κινούμενη από το καθεστώς. Κύριο Κλίντ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, το Καζακστάν έγινε ανεξάρτητο κράτο. Οι πολίτες της χώρας αυτής ε, θεώρησαν ότι αυτή η εξέλιξη θα του οδηγούσε σε μια δημοκρατική χώρα μετά από πολλά χρόνια αυταρχικού καθεστώτος. Ε, ελπίζαν ότι θα έχουν ένα κράτο δικαίου, ότι θα έχουν οικονομία τη αγορά και όλοι οι πολίτε θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθερα και να ε, εργάζονται με αξιοπρέπεια. Δυστυχώ αυτέ ε, οι ελπίδε δεν ευωδόθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο σημαντικότερο εμπορικό εταίρος. Έχουμε τη Συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία από το Δεκέμβριο του 2015, όπου τονίζεται μετεπιτάσεω η σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου. Δυστυχώ, πάνω από τρία χρόνια μετά από αυτή τη συμφωνία, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και μάλιστα σε μερικέ περιπτώσει έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Αθώοι φυλακίζονται, βασανιστήρια πολιτών δεν έχουν την δυνατότητα ελευθερία τη έκφραση, διώξει ε, απλών πολιτών και γι' αυτό θα πρέπει ε, διακομματικά να ψηφίσουμε όλοι ε, αυτό το ψήφισμα για να καλέσουμε την κυβέρνηση του Καζακστάν να κάνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκόμες, ένα λεπτό. Ε, είχαμε λοιπόν στην αποστολή στο Ιράν είχαμε συζητήσει για το καθεστώς Ερμπάιεφ ε, που γίνει μια προσωπικότητα που ζητεί σε ένα κλεπτοκρατορικό σύστημα που έχει δημιουργήσει και αυταρχικό. Και στην αντιπροσωπή αυτά Αλμάτι η αστυνομία του Καζακστάν ε, συνέλαβε ανθρώπους που ήρθαν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και ζητούμε να απελευθερωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν από το καθεστώς οι αντιπολιτευόμενοι, οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το απαιτούμε στο ψήφισμα, απαιτούμε όλοι να απελευθερωθούν, όπως ο Μοκτάζ Κεντάιφ, που ε, έχασε την όρασή έχασε την χώρασή του που όλοι αυτοί που απειλούνται και όλοι αυτοί που διαδηλώνουν που απειλούνται από το καθεστώς. Την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος Αρκάιεφ Επίσης θα παρέμβει, θα μιλήσει, θα πρέπει να τον πιέσουμε να, κάνει μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να συνεχίσει ε, να συνεχίσουμε να συναλλασσόμεθα με τέτοιους δεινοσαύρους που δεν έχουν θέση σε μια τέτοια ε, χώρα. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα τριμερής διάλογος. Ε, θα έπρεπε η Ρόζα του να είναι εδώ, την αντικαθιστώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο. Έχουμε 16 στάσεις για τις οποίες δεν μπορώ βέβαια να αναφερθώ ε, διεξοδικά. Θα αναφερθώ σε σημαντικότερες από αυτές. Ζητεί το ψήφισμα από την κυβέρνηση του Καζακστάν να εφαρμόσει τα όσα ζήτησε ο ειδικό ε, εκπρόσωπος του ΟΗΕ να σταματήσει δηλαδή τις αυθαίρετες προσαγωγές, στην καταστολή ε, και τις προσαγωγές και κράτησαν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να επαναφέρει ε, τον νόμο για την ελευθεροτυπία καταργώντας τις αλλαγές ε, που επέβαλε. Έχουμε και το 174 ε, του ποινικού κώδικα που μιλάει για την παρότρινση σε κοινωνική ιδιαίτερη και το οποίο χρησιμοποιείται με καταχρηστικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Συντροχεύση. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο η κυρία Τζούλι Βόρντερ. Παρακαλώ. Για τα τελευταία πέντε χρόνια Έχω επαφή με την κοινότητα των πολιτών του Καζαχστάν. Στέκομαι αλληλέγγυα με του πρέσβει ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διώκονται. Και έχω εξοικειωθεί με την πολύ ζωφερή κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. πολύ συνανισχυτικέ ε, περιπτώσει. Αυλοβάφηση του Ζεμάγεφ καταδικάστηκε σε τρία χρόνια επειδή online ε, κριτήκαρε την κυβέρνηση και η γυναίκα του, Άγγελα Παντάγεβα, με τέσσερα παιδιά διώκεται για το ίδιο θέμα. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη που το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε δεν αναφέρει το δικό της όνομα. Εκκρεμεί η υπόθεσή της ακόμη. Ε, και είναι το ίδιο σημαντική με τις υπόλοιπε ε, διεθνεί παρατηρητές που παρακολουθούν τέτοιες ε, υποθέσεις απελάβνονται χωρίς καμία αιτιολογία από τις αρχές όπως έγινε στο Λάιν Μαλαβολοσίμα Βαλέρη Λαφτουσέγκο είναι θύματα δικαστές επίσης ο πρόεδρος του δικαστηρίου της ΑΚΤΑ τιμωρούνται αν δεν ακολουθούν τις εντολές και άλλοι όπως ο Αζέντα Μπεσεφ καταδικάζονται σε φυλάκιση όπως ο που καταδικάζονται σε 8 και 7 χρόνια ε, ε, στον αγώνα καταπολέμησης της ε, των ακραίων εκδηλώσεων και του εξτρεμισμού. Όλοι αυτοί πρέπει να δικαιωθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Το λόγο τώρα έχει για ένα λεπτό από τη FTD ο Νίθαν Γκίλ. Ακούστε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ειδική εντολή, έχει ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Πρέπει να είναι ένας φάρος για το Καζακστάν και άλλους. Ε, και Έχουμε τους εκλεγμένους γραφειοκράτες όμως να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Ε, δεν μπορούμε να υποβαθμίζουμε τους ε, ε, ανθρώπους στο Καζαστάν. Έχουμε όμως σημαντικά ζητήματα. Έχουμε τις εκλογές, τις πέτρικες ε, στην Ουκρανία, την, ε, τα θέματα ασφαλείας και πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλες τις χώρες που έχουν συμφωνίες σύνδεση με την Ένωση και ενδεχομένω προσχωρήσουν. Αξιόπιστες πηγές από το Human Rights Watch μιλούν για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν λοιπόν έχουμε το News One και το Channel 112 που ε, ασκούν πίεση πριν από εκλογές, ε, τι να κάνει κανείς, πώς ε, μπορούμε να έχουμε δίκες εκλογές. Εγώ θέλω την ελευθεροτυπία για την Ουκρανία να την υποστηρίξουμε. Έχω ένα ψήφισμα, το υπέγραψα 43, όμως η γραφειοκρατία του το καταπολέμησε και θα το καταθέσουμε στο Στρασβούργο την επόμενη φορά. Ελπίζω αυτό να μην ξανασυμβεί. Εμείς θέλουμε παντού παντού ελευθερία τύπου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου με τον κύριο Χωσή Γνάσιο Φαρία. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Καζακστάν ήταν μία από τις πρώτες χώρες της Κεντρικής Ασίας που έγινε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, του ΟΗΕ, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δικών του πολιτών. Οι πολίτες του Καζακστάν βλέπουν ότι δεν έχουν την ελευθερία του συνέχεστε. Η κοινότητα των ε, ΛΟΑΔΜ και οι αντιφρονούντες διώκονται, ε, υφίστανται βασανιστήρια και βίες ε, συμπεριφορές. Ε, διώκονται οι συνδικαλιστές. Βλέπουμε επίσης ότι ε, οι μετανάστες έχουν πολλούς περιορισμούς, οι θρησκευτικέ ελευθερίες περιορίζονται, μειονότητες διώκονται διαρκώς και είναι αντικείμενο κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της συνεργασίας πρέπει να οθήσει τις αρχές ε, του Καζακστάν ως μέλη της διάσκεψης της Βενετίας να ε, τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και να ζητήσει από την κυβέρνηση της Αστάνα να απελευθερώσει τους όλο και περισσότερους ε, φυλακισμένους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Κύριε Επίτροπε Μίμητσα, Νομίζω ότι είναι μια πολύ δική περίπτωση αυτή ε, που συζητούμε σήμερα, δηλαδή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζαχστάν, έχοντα υπόψη ότι την χάνει προνομιακή ε, σχέση. Έχουμε σημαντική εταιρική σχέση τη Ένωση με το Πακιστάν που τον κάνει γίγαντα ε, στην περιοχή του. Όμω υπήρξε μεγάλη οπισθοδρόμηση ε, δημοκρατική στη χώρα. Ε, μα θυμίζει η εποχή Σοβιτικής Ένωση, η δράση του Προέδρου διώκει του ε, πολιτικού του αντιπάλους Ανασαρμπάγεφ. Έχουμε τον Μουχτάρ Ζαγιέφ, το, ο οποίος έγινε και αντικείμενο ιδιαίτερη προσοχή από τι ειδικέ Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τον ΟΗΕΝ Γέννη. Υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις όπως αυτό του Μουχτάρ ε, που πραγματικά ε, είναι ξόφθαλμη παραβίαση των δικαιωμάτων, βασανίζεται, έχει φυλακιστεί εδώ και καιρό. Η Επιτροπή όμως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, του ΟΗΕ έχει εκφραστεί ξεκάθαρα και πρέπει και εμείς να το στηρίξουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριος Μαριάς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα προστασίας δημοκρατικών δικαιωμάτων στο καζακστάν. οι χώρες αυτές οι οποίες ε, κατάφεραν ή ήθελαν εν πάση περιπτώσει έφυγαν από τον σοβιετικό εναγκαλισμό δεν πέρασαν όμως δυστυχώς στη δημοκρατία. δεν στήριξαν ε, την δημιουργία μιας κοινωνίας των πολιτών ένα χώρο όπου πραγματικά να λειτουργούν τα δημοκρατικά δικαιώματα. από την άλλη πλευρά όμως και η δύση θόπευσε αυτές τις χώρες και τη στόπευσε διότι είχε οικονομικά συμφέροντα διότι εκεί βρήκαν μια μεγάλη ευκαιρία οι πολυεθνικές της ευρώπης αλλά και της αμερικής να κάνουν επενδύσεις να εκμεταλλευτούν τις πλούτοπαραγωγικές πηγές και φυσικά να βγάλουν υπερκέρδη. στη βάση αυτή λοιπόν παρέμειναν τα καθεστώτα δεν έγιναν δημοκρατικές αλλαγές και τώρα έρχονται όλοι να διαμαρτύρονται. αυτή είναι η πραγματικότητα όταν κανείς κοιτάζει μόνο όπως κάνουν οι πολυεθνικές το να κερδίζουν χωρίς να ενδιαφέρονται φυσικά για την ανάπτυξη της δημοκρατίας. εμείς στηριζόμαστε και θέλουμε να στηρίξουμε τη δημοκρατία γι' αυτό στηρίζουμε και το συγκεκριμένο ψήφισμα. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Το Καζακστάν δεν είναι μόνο από τι πιο μεγάλες χώρες στον κόσμο, αλλά και από τι πλούσιες από πλευράς πολιτιστικής ιστορίας και παραδόσεων. Και σίγουρα η συνύπαρξη των διαφόρων κοινοτοτήτων, εθνοτικών και θρησκευτικών καταστούν υπόδειγμα αυτή την χώρα. Μπορούμε να μάθουμε. όμω σήμερα αυτή η ποικιλομορφία και ο πλούτο ο πολιτισμικό απειλούνται από παλαιοχρονικού απειρχαιωμένου κανόνε που στρέφονται εναντίον εκείνου που σκέφτεται φορετικά από την κυβέρνηση. Όλοι και πιο πολλοί ακτιβιστέ και μένει των ΛΟΑΔΜ και δημοσιογράφοι και μέλη των συνδικάτων στοχεύονται χωρί καμία δικαιολογία. Έχουμε τη μαρτυρία του 2016. Χίλια άτομα συνελήφθησαν μόνο διότι συμμετείχαν στη διαδήλωση ειρηνικά. Βιοπραγίε. Στι 10 Μαου που πέρασαν κατά ομάδα διαδηλωτών την ευκαιρία της επίσκεψης μια της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σκεφτούμε τον Αρντάκα ένα, μια μπλόκερ που είναι σε ψυχιατρική κλινική διότι παρακίνησε τη διαφωνία μέσω των αναρτήσεων βάσει του άρθρου 174 του άρθρου του ποινικού κώδικα που ακόμα δεν έχει μεταρρυθμιστεί. Λοιπόν, ο σε τι εξυπηρετεί να έχουμε συμφωνία συνεργασία ενισχυμένη και εταιρική σχέση όταν παραβιάζεται η δημοκρατία, ο σεβασμός της ελευθερίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κέλλη έχει το λόγο. Και Σον Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτό το ψήφισμα αφορά την εισηγητή κατάσταση αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και τη δημοκρατία στο Καζακστάν. Ο νέο ποινικό κώδικα έχει ε, κάνει πιο σοβαρού του ε, νόμου ε, που είναι κατά των ακτιβιστών, των υπολογισμένων και των δημοσιογράφων. Η ελευθερία έκφραση έχει περιοριστεί και πολλοί έχουν φυλακιστεί επί μακρόν χρονικό διάστημα, έχουν βασανιστεί, έχουν υποστεί κακομεταχείριση, ψυχολογική πίεση και βασανισμό. Η χρησιμοποίηση των κοινωνικών δικτύων ελέγχεται και περιορίζεται από τι αρχέ και οι χρήστε των κοινωνικών δικτύων καταδικάζονται σε φυλάκιση για τι σκεφτικέ πεπιθήσει που που χρησιμοποιούνται σαν ε, πρόσχημα θρησκευτικέ πεπιθήσει για φυλακισμό. Καλούμε το Καζακστάν να αλλάξει την νομοθεσία του και κυρίω τα άρθρα που, ποινικοποιούν ε, κάποιες πράξεις που έχουν πολιτικά κίνητα τελικά η, η τιμωρία τους και θα πρέπει να κάνει τι δύο στις στο Καζακστάν για να μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελειώσαμε τα μέλη και ο Επίτροπος ο κύριο Μίμητσα θα παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καζακστάν. Όπως ξέρετε, η συνεργασία, η συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καζακστάν έχει κυρωθεί από 25 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Καζακστάν ένα στέρεο πλαίσιο για να προωθήσουμε τη συνεργασία μας. Η πλήρης κύρωση θα μας δώσει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας και στα ανθρώπινα δικαιώματα, βασιζόμενοι επί του τακτικού ε, διαλόγου που λαμβάνει η χώρα με το Καζακστάν, ο διάλογος περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα πλαίσια της Υποπιτροπής Εσωτερικών και Δικαιοσύνης συζητήσαμε μεταξύ άλλων τη σημασία ανεξάρτητου δικαστικού τομέα και νομοθετικών εξουσιών που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα ε, του συνταγματικού μηχανισμού ελέγχου καθώς και μηδενική ανοχή όσον αφορά τα βασανιστήρια και θα εξασφαλίζουμε την ανεξάρτητη εποπτεία των διαφόρων ε, σοφρονιστικών ε, ιδρυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε ανησυχία σχετικά με, τη, με τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και του συναθρίζεστε. Παραμένει σημαντικό για το Καζακστάν να συνεχίσει να κάνει βήματα, ούτως ώστε να προωθήσει ένα περιβάλλον κατάλληλο για την κοινωνία των πολιτών, για τους προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τους ε, νομικούς, τα μέλη των συνδικάτων, τους δημοσιογράφους. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ ε, τις εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα του Καζακστάν, όπω και σχετικά με επικαιροποιημένο νόμο για τα συνδικάτα και το κατά πόσο συνάδει με τι συμβάσει του Διεθνούς Γραφείου εργασία και με τα πρότυπα τα διεθνή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντί τι έχουν για την κοινωνία των πολιτών οι νόμοι για τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ. Η Επιτροπή συνεργασία με το Καζακστάν τη Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον Ιανουάριο ότι η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχέ του Καζακστάν θα συνέχιζαν συζήτηση επί ανησυχιών που εξεφράστησαν και αυτό κάνουμε. Το κράτο δικαίου θα παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στήριξη που παρέχει στο Καζακστάν μέσω του προγράμματο για το κράτο δικαίου για την Κεντρική Ασία που θα ξεκινήσει το 2019. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, στο τέλος της συζητήσεως θα υπευλήθησαν κάποιες τροπολογίες του πράσινου στο ECR, GUE, ALDE, Σοσιαλιστές Δημοκράτες και ΕΛΚ. Η συζήτηση περατούτε, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ιράν. Η κυρία το θέμα των πρασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε έξι συντάκτες ε, του εγγράφου. Θα ξεκινήσουμε με παρεμβάσεις των συντακτών του εγγράφου. Καταρχάς, ε, συνάδελφος Μποντίν Βαλέρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το καθεστώς το Ιράν δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ξέρουμε, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία της θρησκείας την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, ε, δεν συμμορφώνεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Στο Ιράν μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς πολύ βαριές κατηγορίες. 273 άνθρωποι εκτελέστηκαν το 2018, κινδυνεύουν ιδιαίτερα οι γυναίκες, υπάρχουν αποσπάσματα ταινιών, εικόνων, που δείχνουν ότι ε, ε, έχουν ε, έχουν βάλει πάνω σε ξύλα τα χιτζάπ της, ε, τα καλύμα τη κεφαλής και τα ανεμίζουν. Αλλά πολλέ από αυτέ διαμαρτυρήθηκαν, φυλακίστηκαν. 112 ακτιβίστριες ε, συνελήφθησαν και πολλέ βασανίστηκαν. Και αυτές ήταν επικεφαλής των κινημάτων που υπερασπιζόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών και θα πρέπει να προασπίσουμε τις γυναίκες αυτές. Δεν μπορούμε να σιωπούμε όταν συμβαίνουν αυτά. Η, Σιωτούντε, η Ασφάν Σιωτούντε καταδικάστηκε σε 33 χρόνια κάθυρξη και 168 ε, μαστιγώματα. Και αν συμπεριλάβετε όλα αυτά που έχει περάσει ήδη, 38 χρόνια ακόμα έχει να περάσει στη φυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, η κυρία Κορνέλια ένστε έχει το λόγο. Το 2013 γνώρισα την Ασρίν του στην Τεχεράνη με τον Γιαφάρ Παναγή και οι δύο βραβεία Ζαχάροφ του 2012. Την είχαν απελευθερώσει τότε και μετά από τον Ιούνιο του 2018 ξαναείνε στη φυλακή όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλακή για 148 μαστιγώματα. Είναι σκάνδαλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί είναι ε, ε, άνθρωποι που ξέρουμε ότι αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ζητάμε την απελευθέρωση της Σοτουντέ και όχι μόνο της Σοτουντέ αλλά και άλλων που είναι ακτιβιστές για το περιβάλλον, που κατεβαίνουν στους δρόμους για κοινωνικά θέματα, για ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα για λόγους εθνοτικούς ή θρησκευτικού, δημοσιογράφους. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα θέτουμε συνεχώς χωρίς να χαμηλώνουμε την ένταση της διαμαρτυρίας μας. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλιμακώνονται και σε αυτή την κατάσταση μια διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ιράν πιστεύω ότι είναι σκανδαλώδες να δημιουργηθεί, σκανδαλώδες ε, και μας ντροπιάζει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Έρνστ. Η Μαρία Τεσάκη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο δίνουμε βραβείο Ζαχάροφ και το χορηγήσαμε στην ε, Νασρίν Σοτουντέ, η οποία συνέχισε να εργάζεται με τεράστιο θάρρος για να υπερασπίζεται απλούς πολίτες του Ιράν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ε, εξαιρετικά πολλές περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδίω ήταν δικηγόρος πολλών γυναικών που διαμαρτύρονταν ε, κατά της, του υποχρεωτικού χιτζάμπ, κατά την αφορούν υποχρεωτικά κάλυμα κεφαλής και είναι υπερβολικά παράλογη η καταδίκη της σε 38 χρόνια φυλακής και 148 μαστιγώματα. Είναι, ανθρώπ, είναι απάνθρωπο, είναι απαράδεκτο και η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη, θα πρέπει να μιλήσει δημόσια και να ζητήσει, όπως και εμείς, την άμεση απελευθέρωση της Νασρίν Σοτουντέ. Πιστεύω ότι η αιμονή με τις ε, ε, με την αναζρένηση του η αιμονή των ε, δικαστικών αρχών ε, και των θρησκευτικών αρχών που προσπαθούν ε, να σιγάσουν τη φωνή της αναζρένησης του είναι απαράδεκτη και χρειάζεται να την υποστηρίξουμε απερίφραστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Καν. Κύριε Πρόεδρε, οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, συλλαμβάνονται καθημερινά. Συλλαμβάνονται γιατί διαδηλώνουν για τα δικαιώματα των εργατών, για τα περιβαλλοντικά πρότυπα, κατά τη θανατική ποινή. Η Ιρανική κυβέρνηση στρέφεται κατά δημοσιογράφων του BBC και των οικογενειών του. Παραμένουν φυλακισμένοι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ακολουθούνται οι σωστέ δικαστικέ και δικονομικέ διαδικασίε δόθηκε μια μακρά καταδίκη στην Αθρήν Σοτουντέ, σε αυτή τη γενναία γυναίκα που υπερασπίζεται άλλε γενναίε γυναίκες οι οποίες βγάζουν το κάλυμα τη κεφαλή του. Πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ο περιορισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να ζητήσουμε την απελευθέρωση της νερίνσα του και όλων των άλλων ε, που ε, καταδικάστηκαν ε, με άδικη δίκη και βρίσκονται στη φυλακή άδικα. Δεν μπορούν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο υπόλοιπο κόσμο να παρακολουθεί. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε του Ιρανού που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενο ομιλητή ο Τσάρλ Τάνοκ για ε, Γνωρίζουμε το αποτριαπιαστικό ρεκόρ ε, των ε, εκτελέσεων και των διώξεων, δημοσιογράφοι, παρασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και όλοι όσοι ειρηνικά διαμαρτύρονται κατά της απάνθρωπης κυβέρνησης διώκονται και έτσι καταρρύπτονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία έκφρασης όπως και η θρησκευτική ελευθερία. Το δείχνει αυτό η δίωξη χριστιανών, μπαχάης και άλλων μειονοτήτων. Τους τελευταίους μήνες είδαμε να εντείνονται οι εκστρατείες ε, ε, εφόδων ε, σε τεμένοι χριστιανοί συλλαμβάνονται μόνο και μόνο επειδή ασκούν τη λατρεία της εσκέως. Επίσης τα δικαιώματα των γυναικών περικόπτονται και το 1839 γυναίκες συνελήφθησαν επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά της υποχρεωτικής μαντήλας 273 εκτελέσεις είχαμε το 18, αλλά η αναθεώρηση του νόμου για τα ναρκωτικά ε, δεν φαίνεται ότι έχει επηρεάσει και τόσο τα πράγματα. Ε, ουσιαστικά ο κόσμος δεν μπορεί να ζει καλά. Απομονωμένος λόγω της απομόνωσης από τη διεθνή κοινότητα παίνεται. Ε, πάρα πολύ μικρή ήταν η αλλαγή που έχουμε μέχρι σήμερα διαπιστώσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, του μου είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράν είναι μια από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ε, που εξασφαλίζει για τους ε, πολίτες. Τον δεύτερο πέρυσι στη σειρά σε ό,τι αφορά τις εκτελέσεις, 273 στον αριθμό. Και μπορεί κανείς να προσθέσει πολλές ε, περιπτώσεις που μιλούν για αυτοκτονία κάποιου κρατούμενου. Πέρυσι επίσης δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Ιράν διαμαρτυρήθηκαν για την αύξηση της του κόστου ζωής, ε, για ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ε, να δαπανώνται πολλά χρήματα για βαλιστικούς πυράβλους, ενώ η χώρα πεινάει. Και ίσο του δικαίου σύζυγός του έχουν καταδικαστεί λόγω του ότι μίλησαν κατά της μαντήλας. Φαρέτ, ήδη 9 χρόνια στη φυλακή. Εμείς ζητούμε από την κυβέρνηση του Ιράν να απελευθερώσει άνευ όρων όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, αντιρρησίες συνείδησης, περισπιστές των δικαιωμάτων δημοσιογράφους και λοιπούς. Ναι, για μια ακόμη φορά απευθύνουμε έκκληση. Ζητούμε, παρακαλούμε τις Ιρανικές αρχές να αλλάξουν, να συμπεριφερθούν σωστά. Θα αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Δεν μπορεί το καθεστώς να ζήσει αν δεν υπάρχει βελτίωση κατάστασης. Ζητούμε από την είπατε εκπρόσωπο να απαιτήσει τον σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι αυτό διακόπτεται. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλα, αλλά πρέπει να σας διακόψουμε. Τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Κρίστιαν Ντανπρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η καταδίκη της βραβευτής σας με το βραβείο Ζαχάροφ ε, έχει οδηγήσει σε κατακραυγή στη δημοσία ε, κοινή γνώμη και πραγματικά η καταδίκη της είναι φρικτή και δείχνει ότι η Ιρανική κυβέρνηση προχωρά σε πολύ μεγάλη καταστολή. Είχαμε μία ε, ακρόαση πρόσφατα ε, στην Υποπιτροπή Ντρουά για οκτώ ε, ακτιβιστές για θέματα περιβαλλοντικά που είναι κρατούμενοι στο Ιράν ε, και αναφέρεται και στο ψήφισμα. Εγώ το έχω πει και θα επιμείνω ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πραγματικά πρέπει να είναι στο επίκεντρο ε, των σχέσεων μας με το Ιράν και ελπίζω ο Επίτροπος Μίμητσα να το διαβάσει στην ε, εκπρόσωπο ήθελα να επιμείνω και στο ότι ζητήσαμε να σταλεί ad hoc, αντιπροσωπεία στο Ιράν και ελπίζω αυτό να γίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Φλέκενστάιν δεν έχει έρθει στη θέση του 2.47, οπότε το λόγο θα δώσουμε τώρα στον Bas Μπέλντερ από το ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 40 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν μας έθεσε ενώπιον παραλόγων ερωτημάτων. Φερρυπίν, πού βρίσκεται η, η, απειλή κατά η ασφάλειας από εκείνους τους ανθρώπους που διαβάζουν τη βίβλο ή, το Κοράνι. Αναφέρονται στα λόγια του Θεού. Όμως ένας παπάς και γυναίκα του καταδικάστηκαν σε δεκαετή φυλάκιση που διάβαζαν τη βίβλο. Και είδαμε επιδεινούμενη κατάσταση όσον αφορά τις διώξεις των χριστιανών. Και θα πρέπει να το λέμε αυτό θα πρέπει να καταδικάζουμε το γεγονό. Εγώ με στο, ζω στο Appledorn στην Ολλανδία και έχουμε περσική εκκλησία όπου μπορούν να πηγαίνουν εκεί πιστοί χωρίς κανένα πρόβλημα. Και δεν σέβονται τους μουλάδες πλέον οι άνθρωποι στο, στο Ιράν. Δεν θα πρέπει να υποστηρίζουμε το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν πλέον, αλλά τους απλούς πολίτες του Ιράν που αγαπούν την ειρήνη, όπως η Νασαντίν Σουτουντέ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τέτινα έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια, δίκες. Αυτό είναι το Ιράν σήμερα, όπως το ξέρουμε. Είναι παριθμός ένα χώρα όσον αφορά τις εκτελέσεις κατά κεφαλή. Συγκλονιστικό το 2015 977 εκτελέστηκα, 2016 567, 2017 507, 2018 273. Ακόμα και νέοι και γυναίκες εκτελούνται πολύ συχνά δημόσια. Με, ε, τους κρεμούν από γερανό οικοδομών. Έχουμε την Αστρίν Σουταντέ, που είναι Ιρανή νομικός και υπερασπίζεται τους διοκόμενους. Πέρα από τη μακρά φυλάκιση, έχει καταδικαστεί και σε 148 μαστιγώματα. Ξέρουμε, ε, έχει πάρει το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, και θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου για εκείνου που καταδικάστηκαν και είναι φυλακισμένοι και είναι ανώνυμοι. Προσπαθούμε να κατανομάσουμε κάποιου από αυτού στο ψήφισμά μα. Α πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Το καθεστώς στην Τεχεράνη είναι ένα ποινικό, ένα εγκληματικό καθεστώς. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στέτινα. Ο κύριο Άννα Βέστιγκεν έχει το λόγο. Στο Ιράν είναι μια τρομοκρατική χώρα που προωθεί την τρομοκρατία στην Ευρώπη, προωθεί την τρομοκρατία στην περιοχή του, στην ευρύτερη αλλά είναι ένα κράτος που ασκεί τρομοκρατία κατά του λαού του. Και περιβαλλοντικοί ακτιβιστές και εκείνοι που προσπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θρησκευτικέ μειονότητες και απλοί άνθρωποι που επικρίνουν το καθεστώς διώκονται. Το Ιράν δυστυχώς είναι μία από τις χώρες του κόσμου όπου έχει την πρώτη θέση στον κατάλογο των χωρών που καταστρέφουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν πούμε ότι έχουμε μια εξωτερική πολιτική βάση αξιών, αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη όταν ε, συνομιλούμε με το Ιράν. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάστηκε υπερβολικά επί συμφωνίας με το Ιράν όσον αφορά τις πυρηνικές, ε, την πυρηνική συμφωνία. Φαίνεται η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή δέχεται τον τρόμο που σπέρνει το Ιράν. Ας χρησιμοποιήσουμε τις κυρώσεις σαν αποτελεσματικό όπλο κατά του Ιράν, κυρίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Κατσουδιάη. Ο κύριος Ποσπίσελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση αυτή και χαίρομαι που κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί πριν από λίγους μήνες, όταν συζητούσαμε εδώ με την κυρία Μογκερίνη το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένιωσα ότι προσπαθούσε τις ομότητες του καθεστώτος του Ιράν προσπαθούσε να τις περάσει λίγο ελαφρά ενώ πρέπει να μιλήσουμε για την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή εδώ πρέπει να μεταφέρει στην κυρία Μογκερίνη αυτά τα οποία λέγονται. Τα οικονομικά μα συμφέροντα δεν υπερέχουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχω συνυπογράψει το ψήφισμα συνεισέφερα και εγώ στο κομμάτι σχετικά με την καταπίεση των θρησκευτικών μειονοτήτων και είναι σημαντικό να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα γιατί με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν δεν σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλα τα εγκλήματα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει το Ιράν. Ευχαριστώ πολύ. Αναγκόμε είναι η επόμενη ομιλήτρια. Όλο και περισσότερο υποστηρίζω ότι πρέπει με το Ιράν να συνεργαζόμαστε, αλλά και συγχρόνως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν, να στηρίζει τους άντρες και τις γυναίκες που, βασι... που αγωνίζονται για βασικά δικαιώματα εκεί, οι γυναίκες που κάθε μέρα συγκεντρώνονται με τα λευκά μαντήλια για να μην είναι υποχρεωτικό να αφορούν πια την χιτζάπ. Τον ε, Φεβρουάριο της προηγούμενης χρονιάς είδαμε ότι έχασε τη ζωή του ο Καμπούρ Σαγέντε Μάμι, ακτιβιστής. Τρομερό. Και τώρα έχουμε το δικό μας βραβείο Σαχάροφ που έχει καταδικαστεί σε 40 χρόνια φυλακή. Αλλά και πολλοί άλλοι. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοια πράγματα. Η καταδικαστική αυτή απόφαση κατά της Νασρίν Σότουντεχ βάλει και κατά του ίδιου του πολιτισμού του Ιράν. Λοιπόν, πρέπει αυτό να το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Άννα. Ο κύριος Ντεμπεσμάκερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ποιος ξέρει ακόμα και θυμάται την ε, Ναστρίν Σατουντέχ. Ήταν ε, φιναλίστη για το βραβείο Ζαχάροφ για μας. Και δυστυχώς το Ιράν παραμένει μια τεράστια φυλακή. Τότε δεν τη δόθηκε άδεια να βγει από τη χώρα. Και τώρα 43 χρόνια έχει καταδικαστική και σε 187 μαστιγώματα. Το φανταζόσαστε τι σημαίνει αυτό. Και γιατί, γιατί υποστηρίζει γυναίκες οι οποίες διαμαρτύρονται και δεν θέλουν να είναι υποχρεωτικό να φορούν την χιτζάπ. Και αυτό δείχνει και αποδεικνύει μάλλον αυτά που συχνά μου λένε οι άνθρωποι από το Ιράν, ότι το καθεστώς είναι κατασταλτικό, ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν ε, είναι μια κοροϊδία, αλλά οι ποινές που επιβάλλουν είναι πολύ σοβαρές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Τεχεράν πρέπει να ελευθερώσει όλους τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εμεί όσο δεν αποσαφηνίσουμε στο Ιράν ότι θα υπάρξουν συνέπειες, κύριε Επίτροπε, γι' αυτό θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμεσμάκερ. ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφε. Η Νεσρίνη Σουτουτέ καταδικάστηκε σε 38 ε, χρόνια φυλάκιση και 148 ραπισμούς ε, είναι πραγματικά η ενσάρκωση ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και ακριβώς καταδικάζεται επειδή έχει αφοσιώσει τη ζωή της σε αυτές τις δραστηριότητες. Η όλη διαδικασία και η δίκη τελικά ήταν ένα έσχος και απαράδεκτη. Ε, η μόνη εξήγηση που υπάρχει είναι η διαρκής και αδιάκοπη καταστολή και παρενόχληση ακτιβιστών και δημοσιογράφων που καταδικάζονται επειδή τόλμησαν να αντιταχθούν στο καθεστώς και να το πούν ανοιχτά. Είναι πολιτικοί κρατούμενοι και οι ίδια και οι υπόλοιποι και έχουν την πλήρη μας υποστήριξη. Έχουμε πολλή δουλειά σε πολιτικό επίπεδο ας πούμε, την υλοποίηση τη συμφωνίας για τα πυρηνικά. Αλλά παρά τις κατάφορες αυτές παραφιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Χρειάζεται πιο στενή πολιτική συνεργασία με την Τεχεράνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρούμε και σαφή λόγια για να καταδικάσουμε όλα αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα και διαδικασίες. Ευχαριστώ Φάμπιο, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Δρογεύσκη, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν παρακολουθώ πάρα πολύ την κατάσταση στο Ιράν, αλλά παρακολουθώ την πολιτική ασφαλείας και στην ε, αποστολή στο Πακιστάν, αλλά και στη σημερινή συζήτηση συμμετέχω. Αυτό που με λυπεί, ξέρετε ποιο είναι δεν υπάρχει συνέπεια και συνοχή σε κάποια έγγραφα και σε κάποιες δηλώσεις. Μίλησαμε για το Πακιστάν, για το Ιράν και σε προηγούμενες συζητήσεις για προβλήματα ασφαλείας, για μετανάστευση κτλ. Και σήμερα ασχολούμαστε με ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες καταχρήσεις και παραβιάσεις από πλευράς του Ιράν εις βάρος των ε, ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των γυναικών. Είναι δράμα αυτό που ζουν οι άνθρωποι αυτοί και οι πολιτικές μας πρέπει να έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Για να γίνει αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς πιο αποφασιστικοί, πιο επίμονοι και να στέλνουμε διάφορα έγγραφα σε διάφορες κυβερνήσεις, αλλά όχι μόνο τα έγγραφα αυτά, να τονίζουμε ε, τις ε, συνθήκες που επικρατούν και να είμαστε περισσότερο συνεπείς και πιο επίμονοι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Τζούλι Η κατάσταση του γραπτού τύπου επίσης είναι πολύ ανησυχητική στο Ιράν και ανησυχώ για τους δημοσιογράφους του BBC εκεί που είναι στόχος των Ιρανικών αρχών. Διώξεις ε, λοιπόν ε, ξεκίνησαν το 2009 κατά δημοσιογράφων του BBC όταν ξεκίνησε η δορυφορική τηλεόραση εκεί. Τα πρόσφατα μέτρα όμως έχουν ε, κλιμακωθεί σε βάρος δημοσιογράφων και των οικογενειών τους και οι διώξεις αυτές περιλαμβάνουν και τη διάσταση του φύλου γιατί κατευθύνονται κυρίως κατά των γυναικών και των οικογενειών τους. Τα αποτελέσματα που έχει το Ιράν μέχρι τώρα όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες είναι κάτι πολύ αρνητικό. 248 ε, μαστιγώματα και 38 χρόνια φυλακή είναι κάτι που αποδεικνύει ότι όντως τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, όπως έχουν πει και άλλοι, πρόκειται για εκφαβισμό, πρόκειται για διώξεις και για κακομεταχείριση, όπως επίσης και όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα και όλα αυτά είναι πολύ σοβαρή ευθύνη του κράτους. Ευχαριστούμε. Ιγνάσιο Φαρία τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι πολλές φορές μέχρι σήμερα έχει μιλήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι συμβαίνει με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το καθεστώς του Ιράν. Κατασταλτικό λοιπόν σύστημα. Είναι η χώρα η οποία επιβάλλει περισσότερο κατασταλτικά μέτρα με τις περισσότερες θανατικές ποινές ε, ε, κατά τον πληθυσμό στον κόσμο ολόκληρο. Δολοφονούνται ε, εκατοντάδες άνθρωποι και φυλακίζονται χιλιάδες και γυναίκες. Γιατί, γιατί ζητούν δημοκρατία και ζητούν ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το καθεστώς του Ιράν λοιπόν είναι ντροπή για τον κόσμο και για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. Μέχρι πότε θα περιμένουμε λοιπόν και θα αφήνουμε αυτό το ε, τρομακτικό καθεστώς να συνεχίζει. Έχουν περάσει 40 χρόνια με μια πάρα πολύ σκληρή δικτατορία έχουν βαρεθεί πια οι Ιρανοί, δεν θέλουν πια να συνεχίσουν έτσι. Φτάνει. Ευχαριστούμε κύριε Φαριά. Ε, Τζούντι Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Γίνονται πολλέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώ του Ιράν. Το ακούσαμε σήμερα το πρωί. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ εδώ σε κάποιου μόνο. Οι Ιρανικέ αρχέ συστηματικά στοχεύουν το προσωπικό του BBC όπως επίσης και άλλους δημοσιογράφους Ευρωπαίους. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ε, οικογένειες επίσης στο Ιράν που και αυτές διώκονται. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι με διπλή υπηκότητα. Ε, πολύ προσωπικό, αντιμετωπίζει πολύ αυστηρές, αυστηρή αντιμετώπιση και οι οικογένειές τους επίσης με αυθαίρετες συλλήψεις, με απαγορεύσεις να ταξιδέψουν, αυθαίρετες συλλήψεις κλπ. Κυρίως υπάρχει και δεσφήμιση σε βάρος γυναικών δημοσιογράφων του BBC. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην συνεχίσει να σιωπά για αυτές τις επιθέσεις σε βάρος Ευρωπαίων γυναικών και Ευρωπαίων δημοσιογράφων. Είναι χρέος μας και ευθύνη μας να στηρίξουμε τους δημοσιογράφους. Οπότε χαίρομαι για το σημερινό ψήφισμα. Και οι ίδιες ανησυχίες αναφέρονται και στον ΟΗΕ σήμερα στη Γενέβη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στάνισλαφ Πόλτσακ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, θα ήθελα κι εγώ από πλευρά μου να καταδικάσω το Ιρανικό καθεστώς όπως και οι συνάδελφοι. Είναι καθεστώς τρομοκρατίας, φυλακίζει, βασανίζει τους πολίτες του. Ο κόσμος διώκεται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ουσιαστικά είναι ανύπαρκτα στο Ιράν. Για άλλη μια φορά συζητούμε τα προβλήματα αυτά για νιωστή φορά για το Ιράν και εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε εκείνους που ε, αγωνίζονται ε, κατά αυτού του καθεστώτος. Σας παρακαλώ κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε να ενημερώσετε την κυρία Μογκερίνη για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο διαφωνεί με την ίδια για το Ιράν. Έχουμε διαφορετική άποψη και είμαστε στεναρά απέναντι σε αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς. Εδώ δεν χωράει συγκατάβαση. Και σας παρακαλώ επίσης αλλάξτε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς διαφωνούμε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Παρακαλώ κύριε Μίμητσα για να κλείσουμε τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ. Yeah. Members. Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγους μήνες, μόλις, στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η διεθνής κοινότητα γιόρτασε τη, 17η επέτειο, την 70η επέτειο από την ε, έγκριση τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επί τη ευκαιρία, είπατε εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη, δημοσίευσε μια ανακοίνωση, έκανε μια δήλωση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τονίζει ότι η επετειο την 70 η επετειο απο την εγκριση της διακηρυξη των ανθρωπινων δικαιωματων επι τη ευκαιρια ειπατε εκπρόσωπος, φεντερικα μογκερινη δημοσιευσε μια ανακοινωση εκανε μια δηλωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπου τονιζει οτι υποστήριξε για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων οι ακτιβιστέ είναι στον πυρήνα τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μια από τι ύψιστε προτεραιότητέ τη. Λίγε ημέρε αργότερα, η δέσμευση αυτή επιβεβαιώθηκε από τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με την ακτιβίστρια Νασρίν Σουντούρε, ε, την ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, που τότε, πριν από λίγες ημέρες, μόλις είχε καταδικαστεί και δεχτεί ποινή διότι απλώ ε, προσπαθούσε να προωθήσει οικουμενικώ αναγνωρισμένα δικαιώματα. Η καταδίκη τη ε, ήταν κάτι στο οποίο δηλώσαμε την αντίρρησή μα απευθεία. Η δέσμευσή μα για την ε, προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύει 365 μέρε το χρόνο και όχι μόνο στι 10 Δεκεμβρίου κάθε χρονιά μέρο τη διπλωματικής μα δράση θα πρέπει να είναι να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και μεταξύ αυτών και στο Ιράν. Ένα μέρο τη ε, αρμοδιότητας αυτή αφορά την παρακολούθηση του έργου των ε, υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να βεβαιωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο ότι δεν ε, είναι θύματα παρενόχλησης ή εκφοβισμού εκράτησης. Στο Ιράν αυτό έχει να κάνει και με τη στενή παρακολούθηση της ε, κυρίας Σουτούρε και άλλων, μεταξύ των οποίων λόγω χάρη η ομάδα των οκτώ περιβαλλοντολόγων που κρατούνται από, πέρσι, από φέτος το Γενάρη και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ε, ποινές. Στο Ιράν και σε άλλες χώρες οι προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, κάνουν τρομερή δουλειά. Ε, νομική αρρωγή σε ολόκληρε ομάδε ή κάποιου παραβάτε που μπορούν να αντιμετωπίζουν απειλέ απειλές θανατικής ποινή και ασχέτως εθνοτικής ε, καταγωγής. Πολύ συχνά όμως η δουλειά αυτή αντιμετωπίζεται από το καθεστώς με καταστολή, με καταδίκες και ασχετως εθνοτικης καταγωγης πολυ συχνα ομω η δουλεια αυτη αντιμετωπιζεται απο το καθεστω με καταστολη με καταδικες και φυλακισεις με κατηγορίες που έχουν ε, να κάνουν συνήθως με θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτό αντιφάσκει με το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα και με την Διεθνή Διακήρυξη. Το Ιράν όμως το έχει αναγνωρίσει από το 1975. Και εκεί ορίζεται ότι κανεί δεν μπορεί να είναι θύμα αυθαίρετη ε, σύλληψη ή φυλάκιση, ότι κανεί δεν μπορεί να αποστερείται τη ελευθερία του, εκτό εάν υπάρχουν αποφόντε λόγοι και έχουν τηρηθεί όλε οι ε, δέουσε διαδικασίε όπω τι ορίζει η νομοθεσία. εκτο εαν υπαρχουν αποχροντες λογοι και εχουν τηρηθει ολε οι αναφέρεται και στα πρόσφατα συμπεράσματα για το Ιράν και που ενέκρινε το Συμβούλιο στι 4 Φεβρουαρίου φέτο, ενώ έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε πλήρως τα όσα προβλέπει το συνολικό και ε, σφαιρικό πρόγραμμα δράσης, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία της με το Ιράν θα πρέπει να βασίζεται σε μια εξορροπημένη και σφαιρική προσέγγιση. Όπου υπάρχουν αποκλήσεις και παραβιάσεις θα πρέπει να υπάρχει και αντίδραση ε, και το αντίθετο όπου υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Βάσει λοιπόν αυτή τη προσέγγιση, συχνά έχουμε απευθύνει εκκλήσει στο Ιράν για να δώσει στου προασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα, ένα περιθώριο για να εκφραστούν και να κάνουν τη δουλειά τους. Συχνά έχουμε εκφραστεί επί συγκεκριμένων υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στι συνεννοήσει μα και τι συνομιλίε με τι Ιρανικέ Αρχέ σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο επίπεδο τη ομάδα για τον υψηλό διάλογο Ευρωπαϊκή Ένωση Ιράν και ο ειδικό ε, απεσταλμένο του ΟΗΕ για τα ανθρωπίνα δικαιώματα στον ΟΗΕ συμφωνεί μαζί μα και ενθαρρύνει τι Ιρανικέ αρχέ να του προσφέρουν πρόσβαση στη χώρα, πράγμα που ζητάμε και εμεί. Επίση, τα κράτη-μέλη μα έχουν αναφέρει το θέμα αυτό ε, επανειλημμένο στι διμερεί συνομιλίε του με τι Ιρανικέ αρχέ. Πιστεύουμε και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτές οι πιέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιες θετικέ εξελίξεις που ήδη τις παρατηρήσαμε να σημειώνονται τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων την απόφαση να διορθωθεί ο νόμος ε, του δικαστικού συστήματος το 2017. Έτσι υπήρξε σοβαρή μείωση των υποθέσεων, εκτελέσεων λόγω καταδικών διακίνησης ναρκωτικών. Και αυτό σχετίζεται και με το μέλλον τη υπόθεση των προασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε να ζητούμε περαιτέρω θετικέ εξελίξει σε αυτό το θέμα, με ένα άμεσο δικαιοστάσιο για την πάυση ε, τη ε, εκτέλεση ανήλικων παραβατών. Θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση όλων των ε, ε, προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε νομική αρρωγή, να έχουν το συνήγορο που προτιμούν, να μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της οικογένειάς τους, να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και όχι να είναι θύματα κακομεταχείριση ή βασανιστήριων. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, όπως ήδη κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε αμύωτε τι προσπάθειές μας για να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για τους πρασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίω και φυσικά και στο Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Έχουμε συνοχή, βλέπω, μεταξύ των ε, Ευρωβουλευτών. Έχω το ψήφισμα Γκουέ Άλντε Σοσιαλιστών ΕΛΚ. Έξι ψηφίσματα συνολικά και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε λίγο. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο στην μέση διάταξη που είναι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα. Θα οργανώσουμε με τον ίδιο τρόπο τη συζήτηση, δηλαδή πρώτα θα έχουμε τους συντάκτες του εγγράφου η κυρία μόλις κότα το λόγο. Ευχαριστώ. Μα απασχολούν πολύ οι απειλέ τη κυβέρνηση τη Γουατεμάλα σε βάρο των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίω κατά τη ΣΥΣΙΚ, τη Διεθνού Επιτροπή κατά τη Ατιμορρησία, η οποία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη Γουατεμάλα και έχει βοηθήσει του θεσμού στην Γουατεμάλα να επιβάλλουν το κράτο δικαίου και να διασφαλίσουν την προστασία των ακτιβιστών και της Λολίτα Τσάβες που ήταν μία από τους φιναλίστε του βραβείου Σαχάροφ. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εκφοβισμού σε βάρος της. Επίσης είμαστε πεπισμένοι ότι οι προτινόμενες αλληγές στην νομοθεσία περί νόμου συμφιλίωσης θα υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη ΣΥΣΙΚ. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 5 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη αποφασιστεί να τα δώσει στη ΣΥΣΙΚ. Γίνονται διαπραγματεύσεις με καλό πνεύμα συνεργασίας, οπότε πραγματικά είναι απογοητευτικό να ακούμε ότι το ΕΛΚΑ θα κρατήσει θέση αποχής για το ψήφισμα αυτό. Ελπίζουμε όμω μεγάλη πλειοψηφία να στηρίξει αυτό το ψήφισμα, καταδικάζοντα με σκληρά λόγια τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτου δικαίου στη Γουατεμάλα. Ευχαριστούμε πολύ. Ιγνάσιο Κοράουτορ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η δημοκρατία και το κράτο δικαίου δέχονται επίθεση στη Γουατεμάλα. Οι υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχονται διώξει και σωματικέ και με νόμου καταστολή. Πολύ συχνά τα συμφέροντα των πολυεθνικών ε, καθορίζουν αυτέ τι επιθέσει. Και ταυτόχρονα έχουμε, είχαμε καλύτερα, τη διεθνή κοινότητα για την Ατιμορρυσία στη Γουατεμάλα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση τη παρανομία και την επιβολή του κράτου δικαίου. Όμω πρέπει να γίνουν νέε έρευνε, γιατί ε, ήταν ε, πολλέ οι προσπάθειε παράνομων ενεργειών τη τωρινή κυβέρνηση κατά τη διάρκεια τη πρόκληση εκστατεία και πρέπει να αποκατασταθεί το κράτο δικαίου. Είναι επίκαιρο όλα αυτά, ε, γιατί έχουμε και τι εκλογέ. Το Κογκρέσο τη χώρα θα προβλέψει αμνηστία για εγκλήματα όπω τα γενοκτονία και ε, τα βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των ενόπλων σειράξεων. Εφόσον εγκριθεί αυτό ο νόμο, μπορεί ο πόλεμο να, να επιστρέψει αμέσω στη χώρα και να ε, αρχίσουν ε, οι εχθροπραξίε και τα αντίπεινα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε το Κογκρέσο από το να εγκρίνει αυτή την πράξη τη αμνηστία. Και θα πρέπει η κοινότητα κοινότητα, η Επιτροπή της Ατιμορρησίας να αρχίσει πάλι να λειτουργεί για να προσέλθουν όλοι οι αυτούργοι ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κορά. Επόμενος ομιλητής, ο Ξαβιέ Μπενίτο Θηλουάγα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για δεύτερη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει ψήφισμα για τη σοβαρή κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γουατεμάλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μεγάλε προσπάθειε στη διεθνή συνεργασία με αυτή τη χώρα τη Κεντρική Αμερική. Όμω, οπισθοχωρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότεροι στρατιωτικοί είναι στην κυβέρνηση που προωθούν μεταρρυθμίσει όπω ο νόμο συμφιλίωση που θα δώσει αμνηστία σε εγκληματίας. Όλο και περισσότερο όμω η εισαγγελία πλησιάζει υψηλά ιστάμενου τη κυβέρνηση, ακόμα και τον ίδιο τον πρόεδρο. Οι 26 ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων δολοφονήθηκαν την προηγούμενη χώρα, χρονιά στη χώρα. Και μεταξύ αυτών τέσσερι δημοσιογράφοι με τι εγκλήματα, με, ε, ενώ άλλοι κάνουν εγκλήματα μάλλον τα οποία μένουν ατιμόρυτα. Η Λολίτα Τσάβε, για παράδειγμα, εξακολουθεί να μην μπορεί να επιστρέψει στη χώρα τη ή το κάλε γιατί δεν μπορεί να έχει μια δίκαια δίκη. Γι' αυτό, όπως πολύ σωστά λέει το ψήφισμα που θα εγκρίνουμε, πρέπει να σκεφτεί πώς πρέπει η συμφωνία σύνδεσης με την Γουατεμάλα να σταματήσει όσο δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μπεατρίς Μπεσέρα Μπαστερέιτσαια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η Διεθνής Επιτροπή κατά της ατιμορρησίας στη Γουατεμάλα έχει κάνει εξαιρετικό έργο στα 11 χρόνια που λειτουργεί. Μπόρεσε να διερευνήσει πάνω από 100 περιπτώσεις και να καταδικάσει 300 άτομα και να παρουσιάσει και 34 νομικές εκθέσεις. Όλα αυτά μέχρι που έφτασε κοντά στους συγγενείς του Τζίμι Μοράλες, του Πρόεδρου. Τότε έπαψε να είναι χρήσιμη. Ο Μοράλες λοιπόν έχει μια ε, εθνικιστική ρητορική που μπορεί να μην φτάνει στο εγκληματικό επίπεδο της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, αλλά παρόλα αυτό ο αντιδραστικός του λαϊκισμός είναι καταστροφικός για τους θεσμούς της χώρας. Η περίπτωση αυτή λοιπόν της Γουατεμάλα είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, γιατί κινδυνεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαιώματο και περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει ώστε να σταματήσουν οι παραβιάσει αυτέ, να διερευνεί τη διαφθορά και να μην επιστρέψει ποτέ πια στη Γουατεμάλη η ατιμορρησία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Ραμόν Χαουρεγγί, παρακαλώ. Ατόντο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνετε να προφέρετε το όνομά μου. Μιλάμε για μια χώρα, τη Γουατεμάλα, που είναι πάμφτωχη, με τεράστιες ανισότητες και μια υποκουλτούρα βίας τεράστια και παρουσία εμπορίου ναρκωτικών πολύ επικίνδυνη. Η χώρα αυτή είναι γεμάτη διαφθορά, υπερβολική διαφθορά. Και επίσης ισχύουν αυτά που είπατε, ε, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στο κράτος δικαίου και ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά μιλούμε για μια χώρα φίλη, με την οποία συνεργαζόμαστε, την οποία αγαπάμε και θέλουμε να βοηθήσουμε, που θα έχει και εκλογές τον Ιούνιο, πάρα πολύ σημαντικές. Και έχει αποθέσει και μεγάλες ελπίδες αυτή την πολιτική αλλαγή για να χαράξει μια καλύτερη μέρα. Η Ευρώπη θέλει να βοηθήσει το λαό αυτό και τη χώρα αυτή. Και το πράττει σήμερα, μάλιστα καταδικάζοντας μια κυβέρνηση η οποία ε, πραγματικά παραβιάζει σοβαρά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ιδιαίτερα με την εκδίωξη της Διεθνούς Επιτροπής κατά της διαφθοράς τη ατιμορρησίας που είναι το σημαντικότερο από τα σημαντικότερα όργανα του ΟΗΕ και προειδοποιούμε ότι αν δεν προχωρήσει προς την ελευθερία και τη δημοκρατία θα υπάρξουν κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Ραμόν λέει ο Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Δεχόφσκι παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε. Πιστεύω Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τυχερή που είναι θεμελιωμένη σε τέτοιε αρχέ και αξίε. Η δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Και για τη Γουατεμάλα βλέπουμε να συμβαίνει εδώ κάτι ε, το ανίποτο. Γιατί εάν δεν κάνουμε τώρα κάτι για το καθεστώς της χώρας, αυτά ε, στο μέλλον ποτέ δεν θα μπορέσουν να γίνουν πράξη σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν προβλήματα με τη διαφθορά, με την οθεία ε, και που οδήγησαν στην εκλογή της σημερινής κυβέρνησης και το καθεστώς της χώρας. Ε, αλλά αυτή η διαφθορά πρέπει να καταπολεμηθεί. Μιλάμε για μια δικτατορία που έχει την κυβέρνηση. Ε, εάν δεν γίνει κάτι τώρα, θα... Θα... Δεν θα δει ποτέ ο λαό τη χώρα αυτή τη δημοκρατία εξή να γίνονται πράξη. Η χώρα λοιπόν έχει πολλά προβλήματα και δεν είναι μια χώρα ομοιόμορφη και ομοιογενή. Τα τελευταία χρόνια οι εκπρόσωποι τη κυβέρνηση έχουν βασίσει την πολιτική του σε εθνικιστικά και τοπικιστικά συμφέροντα. και έχουν υποδαβλήσει το μίσος κατά των επικριτών τους. Αυτά όλα δείχνουν ότι ο κόσμος δικαίως ε, ξεγείρεται και όσοι προσπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα κακώ δεν προστατεύονται αρκετά. Πρέπει να καλέσουμε τη διεθνή κοινότητα λοιπόν να βοηθήσει τον κόσμο τη Γουατεμάλα, του ανθρώπου τη Γουατεμάλα και να αλλάξει η πολιτική κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ε, έχουμε τους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο έχει ο κύριος ε, Χωσέ Γνάσιο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Είχα το προνόμιο να εκπροσωπήσω το κοινοβούλιο αυτό όταν υπεγράφησαν οι ρευτικές συμφωνίες στην Γουατεμάλα και όλοι ελπίζαμε ότι θα προχωρήσει προς της ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Παρόλα αυτά, δεν είμαι πεπισμένος ότι το ψήφισμα αυτό αποτυπώνει πιστά την πραγματική κατάσταση στη χώρα. Ωστόσο, Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω κάποια από τα στοιχεία του ψηφίσματος και συγκεκριμένα την ανάγκη να υπάρξει γνήσια και πραγματική αξιολόγηση ως προς τον αντίκτυπο της εργασίας της Επιτροπής αυτής για τη δικαιοσύνη, τα πολιτικά, οικονομικά και θεσμικά ζητήματα. Και κυρίως, Πρόεδρε, να διερευνήσουμε για ποιο λόγο ένα τέτοιο θεσμό που έχει γενική εκτίμηση και υποστήριξη εντό και εκτό τη χώρα, σιγά σιγά την έχει χάσει αυτή και έχει αποδυναμωθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαλαφράγκα, με ακούτε. Ωραία. Ε, ε, έχει μια μπλε κάρτα κάποιος συνάδελφος. Δέχεστε. Ε, κυρία Μιράντα, παρακαλώ. κυρία Μιράντα. Η κυρία Μιράντα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, έχω μείνει άναυδη όταν γίνεται λόγος για ε, ανθρώπινα δικαιώματα σε τόπους όπως η Βενεζουέλα, αλλάζεται ε, κριτήριο. Εδώ έχουμε κοινό ψήφισμα που έχει υπογράψει και το ΕΛΚ και ακούσαμε πάρα πολύ σημαντικά σήμερα από το ΕΛΚ και εσείς τι λέτε. Αποχή ή ότι καλά δεν είναι και τόσο βαθύ το ψήφισμα. Πραγματικά εμένα με εκπλήσει αυτή η υποκρισία. Άρα λοιπόν, θα υπερψηφίσετε αυτό το ψήφισμα. Είστε διατεθειμένοι. Ε, ε, Ο κύριος Σαλαφράγκα. Καλά τώρα υποκρισία δεν συνάδει με την κοινοβουλευτική ευγένεια και με το σεβασμό. Έχουμε ελευθερία της έκφρασης εδώ. Ε, ο άνθρωπος με το λόγο είναι ε, ανώτερος από τα ζώα, αλλά με τη σιωπή είναι ανώτερος από τον εαυτό του. Και σήμερα χάσατε μια ευκαιρία να αποδειχθείτε ανώτεροι με τη σιωπή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Σαραφράγκα, έχετε κι άλλη μία. Δέχεστε. να σας... Ε, παρακαλώ, για ερώτηση. Δεν δέχεστε την ερώτηση. Α, δεν δέχεται την ερώτηση ο κύριος Αλαφράγκα. Ωραία, ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Φρανσίσκο Ασής. Παρακαλώ. Πρόεδρε, δυστυχώς και πάλι μιλάμε εδώ για μια οπισθοδρόμηση του κράτου δικαίου σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Είχαμε χθε την ευκαιρία να συζητήσουμε το ψήφισμα για την Ικαράγουα και έγιναν δηλώσει ε, έντονες κατά δίκη τη οπισθοδρόμηση του κράτου δικαίου, του κράτου δικαίου στην Ικαράγουα. Διαφορετική ιστορία σήμερα, αλλά παρόμοιε καταστάσεις. Στην Γουατεμάλα αυτά που συμβαίνουν σταδιακά είναι πραγματικά πολύ αρνητικά σε σχέση με το σεβασμό των βασικών κανόνων κράτους δικαίου. Και μεταφράζονται και ήδη μεταφράστηκαν σε αποφάσεις που οδηγούν στην πάυση λειτουργία μια διεθνού επιτροπή ε, για την καταπολέμηση τη ατιμορρησία. Που είχε πετύχει κάποιε θετικέ εξελίξει και είχε καταφέρει κάποια πλήγματα στη διαφθορά στη χώρα. Τώρα ε, το Κογκρέσο θα ψηφίσει αμνηστία που αντίκειται στι βασικέ αρχέ του δικαίου. Εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε οπωσδήποτε και του εθαγενεί τη χώρα, ε, τους αυτόχθονες που διαρκώ διώκονταν στη Γουατεμάλα και καταπιέζονταν ω προ τα βασικά του δικαιώματα. Θα πρέπει να γίνει μια ειδική μνήμα και σε αυτού από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Άννα Μιράντα, τώρα εξ ονόματο τη ομάδα τη, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανησυχούμε πάρα πολύ από την κατάσταση στη Γουατεμάλα. Επιθέσεις υφίστανται οι αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι αυτόχθονες λαοί και οι κοινωνικοί αγωνιστές. Και αυτά δεν σταματούν. Και επίσης ε, στηρίζουμε τον Διευθυντή της Επιτροπής κατά της Ατιμορρησίας γιατί κατήγγειλε περιπτώσεις διαφθοράς ε, ε, από πλευράς του αδελφού και του γιού του Προέδρου. Και ε, ε, επίσης ε, υπάρχουν και κάποια ζητήματα με τη Σουηδική Πρεσβεία. Τι γίνεται λοιπόν με τις εκκλήσεις προς τη βία. Η ΜΚΟ τι θέλουν. Να διαδηλώνουν ελεύθερα και να συνέρχονται ελεύθερα. Ε, κάθε μέρα η κατάσταση χειροτερεύει στη Γοτεμάλα. Ανησυχούμε για του αγωνιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την αγαπημένη μα Λολίτα, για όσου ε, βρίσκονται κρατούμενοι στι φυλακέ. Και η Λολίτα θα πρέπει να μπορεί ειρηνικά να επιστρέψει στη χώρα τη και να προστατεύονται οι αγωνιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί τι θέλει η κυβέρνηση τη Γοτεμάλα να διατηρήσει τα προνόμια κάποιων πλούσιων οικογενειών, λίγων, που νομίζουν ότι η χώρα του ανήκει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Μιράντα και τώρα ο κύριος Σόσνιαρτς, μία εγγεγραμμένος. Ναι. Εδώ έχουμε χαρακτηριστικές ε, και επίμονες πράξεις ε, σεξιστικού χαρακτήρα οι οποίες καταστρέφουν ε, τις καλύτερες πρωτοβουλίες αυτού του κοινοβουλίου. Στο Ευρωκοινοβούλιο βρέπουμε έναν μια διαρκή αύξηση γυναικοκτονιών. Δεν μιλάτε όμως και για τις ανδροκτονίες, τις δολοφονίες ανθρώπων ε, που τους 5.000 που έχασαν τη ζωή τους. Λέτε ότι ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν αυξάνεται και δεν λέτε τίποτα για τους ε, υπόλοιπους άνδρες. Ε, φαίνεται ότι έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά και κάθε φορά λέτε ό,τι σας βολεύει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πιανού. Εάν διαβάσουμε το κείμενο, ιδίω για τι γυναίκε προασπίστριε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί, γιατί γίνεται ειδική μνήμα και τονίζονται οι γυναίκε, τι, τι θέλετε να πείτε με αυτό. Πραγματικά χαίρομαι που αυτή η θητεία τελειώνει και ελπίζω όλοι αυτοί οι σταχανοβιστές του φεμινισμού να μην εκλεγούν στην επόμενη θητεία. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλευτά. Η... Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γουατεμάλη η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, κυρίω εξαιτία των επιθέσεων σε βάρο ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, κυρίω εξαιτία τη βία σε βάρο των γυναικών που αυξάνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και κυρίω εξαιτία των σχεδίων του Κογκρέσου τη Γουατεμάλα για τον νέο νόμο για γενική αμνηστία. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να μνηστευτούν άτομα που ήταν εγκληματίες πολέμου κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου εκεί. Κάτι το οποίο θα πλήξει βέβαια και την ε, ασφαλεία και την προστασία των θυμάτων τους. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ, ε, πρόκειται και για ένα μήνυμα που στέλνεται γενικότερο για το ότι αμβλύνουμε έτσι τα πράγματα και δεν είμαστε τόσο αυστηροί να καταδικάζουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε σαν Κέλλη τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Κέλλη. Ε, Ευχαριστούμε. Ενώ έγιναν κάποια βήματα πρόοδου στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χάρη στη συνεργασία ε, του ΟΗΕ και τη Διεθνού Επιτροπής για την καταπολέμηση της ατιμορρυσία στη Γουατεμάλα, όλα αυτά ανεστάλησαν λόγω της απόφασης του κ. Μοράλε να μην ανανεώσει τη θητεία της Επιτροπής αυτής που εξέπνευσε εκπνέει τον Σεπτέμβριο του 2019 και δεν θα μπορέσουν όσοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες να ξαναγυρίσουν στη χώρα. Όμως η καταπολέμηση της ατιμορρησίας στη Γουατεμάλα, χάρη στη λειτουργία αυτής της Διεθνού Επιτροπής, είναι σημαντική. Θα πρέπει ο κ. Μοράλε να ανακαλέσει την απόφασή του αυτή και να επιτρέψει σε πολλούς όπως τον, στον κύριο Βελάσκες να, ε, να, ξαναγυρίσει στη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε η ατιμορρησία αυτή να ε, καταπολεμηθεί να πάψει ο εκφοβισμό και η παρενόχληση δικαστικών λειτουργών, ε, δικηγόρων, δικαστών. Δεν λειτουργεί αυτό ανεξάρτητα ο δικαστικό κλάδο και αυτό συνεχίζει να είναι ένα πρόβλημα στη χώρα. Σα ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑΕ. Ο κύριο Πόσπισιλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με του προηγούμενου ομιλητέ που ζήτησαν ε, να υπάρξει κάποια κίνηση για να γίνει μια αλλαγή στην Γουατεμάλα. Ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη ήταν ταγμένο στο σκοπό τη καταπολέμηση τη διαφθορά στη χώρα και πρέπει να πω ότι η Επιτροπή τη ε, Ατιμορρησία, καταπολέμηση τη η ΣΥΣΙΓ, έχει ουσιαστικά οδηγηθεί σε κατάργηση από την κυβέρνηση. Ε, Πρέπει λοιπόν να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι γι' αυτό. Πρέπει να πούμε ένα ηχηρό όχι και να αντισταθούμε. Υπάρχει πολλή διαφθορά ε, και έχουμε μέχρι και δολοφονίες ε, αντιφρονούντων. Χρειάζεται η χώρα λοιπόν αυτή ένα διεθνή, διεθνή φορέα που θα αντιμετωπίσει την ατιμορρησία και την παρανομία. Ε, δεν πρέπει να εφαρμοστούν οι αποφάσει τη κυβέρνηση για την κατάργηση λειτουργία τη ε, ΣΥΣΙΝ, τη Επιτροπή για την Ατιμορρησία. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε παρά να τονίσουμε την δυσαρέσκειά μα σε σχέση με την πρόσφατη δράση τη κυβέρνηση και τι αποφάσει τη. Ευχαριστούμε, κύριε Πόσπισιλ. Ο κύριο Καστάλντο. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Από την εφηβεία, η κυρία Μαρία Μανταλένα Κουκτσόκ ε, προμαχόταν, ε, ε, ε τον τόπο του Ελεστόρ, τον τόπο των Μάγια, ένα τόπο με ηθαγενείς φυλές και πλούσιους φυσικούς πόρους. Είναι πολλαπλές οι διαμάχες για την ε, αξιοποίηση των ε, φυσικών πόρων στη Γουατεμάλα και οι εχθροπραξίες επανειλημμένες. Έχουμε αύξηση των ε, επιθέσεων κατά 336% σε σχέση με την περασμένη χρονιά φέτο στη χώρα. Ε, και η χειρότερη απόφαση φέτο είναι η ανάκληση τη λειτουργία τη Διεθνού Επιτροπή για την Καταπολέμηση τη Ατιμορρησία. Παράλογη ε, απόφαση για την κατάρριξη του νόμου τη Εθνική Συμφιλίωση που προβλέπει ατιμορρησία για όλα τα εγκλήματα και τα δικήματα ε, τη κυβέρνηση και μεταξύ αυτών των εγκλημάτων κατά τη ανθρωπότητα. Το τίμημα που θα πληρωθεί θα είναι υψηλότατο, κυρίω εν ώψη των επερχόμενων εκλογών του καλοκαιριού. Θα πρέπει η κυβέρνηση τη Γουατεμάλα να κάνει κάτι και για τα δικαιώματα των ηθαγενών λαών και να δεχτεί ε, τουλάχιστον τη ρήτρα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία Συνεργασία μα. Αν εμεί δεν την προασπιστούμε, δεν θα μα ε, πιστέψουν ποτέ οι άνθρωποι τη Γουατεμάλα. Κυρία Μορβάη. Thank you very... Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Επίτροπε και αγαπητοί συνάδελφοι, ως δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Πάντα συγκινούμε πάρα πολύ με τέτοιου είδους ιστορίες, σαν αυτές που ακούμε σήμερα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι για πολιτικούς λόγους υφίστανται ε, αυθαίρετες ποινικέ δίκες, έχουμε πολιτικούς κρατημένους που ε, ε, υφίστανται και πάλι κακομεταχείριση ακόμα και βασανιστήρια. Σήμερα πήγαμε με αυτές τις ιστορίες στο Καζακστάν, στο Ιράν και τη Γουατεμάλα. Αλλά εν παρόδο, κύριε Επίτροπε, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων στη Γαλλία και την Ισπανία. Τι συμβαίνει με εκείνες τις εκατοντάδες που μπορεί να είναι και χιλιάδες που συνελήφθησαν κατά τις μαζικές διαδηλώσεις από τις αρχές ε, του κυρίου Μακρόν. Τι γίνεται, ποια είναι η νομική τους κατάσταση τώρα και τι γίνεται με τους πολιτικούς κρατουμένους που συνελήφθησαν επειδή αγωνίζονται για την αυτοδιάθεση της Καταλωνίας. Θα μπορούσατε έτσι σύντομα να μας ενημερώσετε και ε, για την κατάστασή τους ή και όχι τόσο σύντομα όσο θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Ζωζέ Ιγνάσιο Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά... Ε, την επίσκεψή μου στην Ικαράγουα πριν από δύο μήνες για να δω επιτόπου τι συμβαίνει ε, και τι γίνεται με την αντιπολίτευση στον Τανιέλ Ορτέγα. Ε, τώρα βλέπουμε ότι η ε, Γουατεμάλα κινδυνεύει να τορπιλήσει το νόμο ε, για τη συμφιλίωση που εγκρίθηκε πριν από 22 χρόνια για την καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Ξέρετε ότι ε, υπήρξε ένα θέμα αμνηστίας πριν από λίγο καιρό, αλλά ε, η κυβέρνηση εμποδίζει τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να εργαστούν και κυνηγάει και διώκει τους αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εγκριθεί κάποιοι νόμοι οι οποίοι συνιστούν ε, πραγματική οπισθοδρόμηση για τη Γοτέμαλα. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα να επανέλθουν. Ευχαριστώ ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γουατεμάλα είναι μια φτωχή χώρα με τεράστιες δυνατότητες που δυστυχώς παραμένουν μερικώς αναξιοποιητές. Η χώρα αυτή είχε μπει σε ένα σωστό δρόμο. Δυστυχώς η κατάσταση έχει αλλάξει, έχει επιδεινωθεί δραματικά όπως ακούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε πως έχει η κατάσταση γενικότερα. Επίσης γίνεται λόγος για ατιμορρησία και για καταχρήσεις και αυθαιρεσίες. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κατάσταση αυτή γιατί αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βία κατά των γεκών. Όπως είπε και ο κύριος Σόσνιερς, υπάρχει επίσης και η βία κατά των ανδρών. Ε, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι δράστες δεν είναι γυναίκες σε αυτή την περίπτωση. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και τη διεθνή πίεση αλλά και το μέσο της αναπτυξιακής βοήθειας ως μοχλό πίεσης γιατί θα πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ σκληροί απέναντι στις αρχές της χώρας αυτής. Ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα ο Επίτροπος. Παρακαλώ κύριε Μίμητσα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ στο σώμα σας όσον αφορά την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γουατεμάλα έχουν στέρες διμερείς σχέσεις που βασίζονται σε δέσμευση και από τις δύο πλευρές υπέρ αυτής και σε εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας ανησυχεί η αποδυνάμωση του κράτους δικαίου που υλοποιείται μέσω των πρόσφατων επιθέσεων ε, κατά των προσπαθειών που γίνονται για τα καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Όπω επίση ε, που φαίνεται και από τη δράση τη κυβέρνηση που θέλει να σταματήσει τη δράση τη επιτροπή ΣΥΣΙΚ, της Διεθνού Επιτροπή κατά τη Ατιμορρησία. Επίση, υπάρχουν κοινοβουλευτικέ πρωτοβουλίε που μπορεί να μειώσουν το δημοκρατικό χώρο, όπω επίση και να γενικεύσουν την ατιμορρησία για εγκλήματα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχει στηρίξει πάντα την ΣΥΣΙΚ και οικονομικά και πολιτικά. Τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 22 εκατομμύρια ευρώ στο σώμα αυτό του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς και της ατιμορρησίας. Το 2019 είναι η τελευταία χρονιά βέβαια της ε, θητείας της Επιτροπής αυτής και δίνουμε πάλι 5 εκατομμύρια. Τα επιτεύγματα στην καταπολέμηση της διαφοράς, διαφθοράς και ατιμορρησίας είναι πράγματι εντυπωσιακά και έχουν συνεισφέρει και στην μείωση της εγκληματικότητας στη Γουαταμάλα. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, η ΣΥΣΙΚ είναι δημοφιλής. Τη θαυμάζει ο κόσμος και τη σέβεται στη Γουατεμάλα, γιατί ο λαός εκεί ξέρει ότι διαφθορά υπονομεύει πάρα πολύ σοκρά το κράτος δικαίου, τους θεσμούς ε, και τελικά και την δημοκρατία στη χώρα. Οπότε επιτρέψτε μου να το επαναλάβω ενισχύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Γουατεμάλα, στηρίζει την δέσμευσή της να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη ΣΥΣΙΚ. Και βέβαια συνεχίζουμε να στηρίζουμε και όλες τις προσπάθειες που γίνονται κατά της διαφθοράς που πλήττει πολλές φορές και το δικαστικό σώμα παίζουμε σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ατιμορρησίας. Η διάκριση των εξουσιών και ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις είναι ζωτική σημασία γιατί αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους δικαίου. Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στη Γουατεμάλα έχει βελτιωθεί τελευταία. Όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε την προστασία των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων ακτιβιστών και να αποφύγουμε ε, θανάτους, επιθέσεις. Αυτό επίγει οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ήδη πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Διπλασιάστηκε ο αριθμό ε, των ε, τραυματισμών και των θανάτων τους πέρυσι. Επίσης άτομα από ευάλωτε ομάδες, οι αυτόχθονες, οι υποστηρικτέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή από την κοινότητα ΛΟΑΔ αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων. Τέλος, σεβόμενοι πλήρω τη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα, Συγχρόνω θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για δύο νομοσχέδια τα οποία συζητιώνται σήμερα στο Κοινοβούλιο της Γουατεμάλα, όπως πολύ σωστά είπε και ο Ιγνάσιο Κοράου. Το ένα νομοσχέδιο περιορίζει το χώρο στον οποίο μπορούν να δρουν οι οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών. Κάτι το οποίο υπονομεύει το δημοκρατικό ρόλο που μπορεί να παίξει μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Το δεύτερο νομοσχέδιο μεταρρυθμίζει την νομοθεσία για την συμφιλίωση μετά τον φίλιο πόλεμο και προσφέρει ατιμορρησία για εγκλήματα που έγιναν κατά της ανθρωπότητας. Χτες, η αντιπροσωπεία μας στην Γουατεμάλα μαζί με πρεσβείες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν ε, στη χώρα μαζί με τον ΟΗ και τον Καναδά ε, κάτι κατά ακριβώς τη νομοσχεδίου αυτού. Και χτες το Κογκρέσο τελικά δεν είχε απαρτία προκειμένου να συζητήσει το σχέδιο αυτό αμνηστίας. Αλλά εμείς πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί γιατί παραμένει στο τραπέζι, δεν έχει φύγει παντελώς. Η χώρα επίσης τον Ιούνιο θα έχει εκλογές. Και εμείς σεβόμαστε απόλυτα την προεκλογική περίοδο στην οποία μπαίνει η Γουατεμάλα. Οι εκλογές είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα. Ο κόσμος ενωμένο πρέπει να συζητήσει και να αποφασίσει ποιο θα εκλέξει. Πρέπει η αυτή να ενισχύσει την δημοκρατία και το κράτος δικαίου και όχι να αμφισβητήσει αυτά τα βασικά στοιχεία και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Έχω επτά σχέδια ψηφίσματος για ολοκλήρωση της συζήτησης αυτής από τους Πρασίνου, το EFTD, το ECR, την ΚΟΕ, e, την ΑΛΔΕ, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το ΕΛΚ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση για αυτό το θέμα και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σε λίγο. Ε, σταματάμε μέχρι τις 12 ακριβώς, όπου θα αρχίσει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφου για τη συνεργασία. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Der Präsident! Die Sitzung ist eröffnet. Επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση. Καταρχάς έχω δύο ανακοινώσεις να σας κάνω. έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε μια αντιπροσωπεία της Καναδικής Βουλή υπό την Προεδρία του Σκοτ Σιμς. Έχουν έρθει για να συμμετάσχουν στην 40η Επιτροπή ε, κοινοβουλευτικη Συνεργασίας ευρωπαικη ενωση Καναδά. Οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά τα περασμένα χρόνια, χάρη στην σύναψη τη Συμφωνία για μια στρατηγική εταιρική σχέση και μια ευρεία συμφωνία οικονομική και εμπορική, καθώ επίση και μετά την επίσκεψη και ομιλία του Πρωθυπουργού Τριντό το 2017 έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Αυτό είναι έκφραση όχι απλώ των κοινών αξιών Καναδά και Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε και πολλού τομεί, πολλέ κοινέ πρωτοβουλίε για την προώθηση τη πολυμερού συνεργασία, τη ειρήνη, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Η παρουσία τους στο Κοινοβούλιο συμβολίζει και την ευάθυνση των διακοινοβουλευτικών σχέσεων μεταξύ των κοινοβουλίων μας που ήδη έχει διατρανωθεί σε μία κοινή δήλωση του έτους 2017. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζουμε θερμότατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, ελπίζω να είχατε επιτυχείς συνομιλίες και σας εύχομαι καλή διαμονή και ό,τι το καλύτερο. Πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα και πάλι εξ ονόματο όλων μα να καλωσορίσω μια αντιπροσωπεία Ουκρανών βουλευτών που ήρθαν για να συμμετάσχουν στην ενάτη η ε, σύνοδο της ε, Επιτροπή σύνδεση με την Ουκρανία, που είναι και τελευταία για αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Αγαπητοί φίλοι από την Ουκρανία, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, το κοινοβούλιο μα την περασμένη πενταετία ασχολήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή με την κατάσταση στη χώρα σα. Αυτό το κάναμε για να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις όπως ζητούσε ο κόσμος στην πλατεία Μαϊντάν αλλά και για να υπερασπιστούμε την εδαφική σας ακεραιότητα και κυριαρχία. Και μάλιστα αυτό εκφράστηκε πιο πρόσφατα με την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ το 2018 στον Όλεξ Σέντσοφ. Χαιρόμαστε που είστε ανάμεσά μα και ελπίζουμε να είχατε πάρα πολύ επιτυχεί και ε, γόνιμες συναντήσεις. Ευχαριστώ. Καλώ ορίσατε και πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, την τελευταία φορά που προείδρευα στις ψηφοφορίες ε, ανακοίνωσα ότι Τώρα εδώ παραμονές εκλογών θα ε, δέχομαι να μιλούν συνάδελφοι που ε, αναφέρονται αποκλειστικά στον κανονισμό. Παρακαλώ να μας πείτε ποιο άρθρο επικαλείστε. Πραγματικά να είστε βέβαιοι ότι για τους περισσότερους έχω κάθε συμπάθεια με τα θέματα και τα μελήματά σας, ε, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο και θα τηρήσω αυτή την αρχή του κανονισμού. Με μία εξαίρεση. Για ποιο λόγο διότι σήμερα δεν συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων, οπότε θα ήθελα να δώσω την ευκαιρία στον συνάδελφο Λαμπέρτς να μας πει κάτι που ήθελα να πει στη διάσκεψη των Προέδρων. Κατά τα άλλα, κανένας εκτός κανονισμού. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, Πρόεδρε. Merci, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, βάσει του άρθρου 11, εδάφιο 1 του εσωτερικού μας κανονισμού θέλω να θυμίσω σε όλους ότι εδώ λέω ότι η συμπεριφορά των μελών πρέπει να διέπεται από αμοιβαίο σεβασμό και να βασίζεται στις αρχές που περιλαμβάνει και η συνθήκη ιδίω στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για όλα τα μέλη και συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου μας. Όλοι θα σέβονται την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και δεν θα κάνουν τίποτα που μπορεί να πλήξει το κύρος του και τη φήμη του. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ε, χθες, ε, ε ο κ. Σταγιάννη, έκανε δηλώσεις ε, στα Ιταλικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το φασιστικό καθεστώς του Μπενίτο Μουσολίνη στην Ιταλία και μάλιστα ε, πρημοδοτεί τη θέση ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και καλοί σε καθεστώτα που ισοπεδώνουν τη δημοκρατία. Τέτοιες δηλώσεις είναι απαράδεκτες και δεν αρμόζουν σε πρόεδρο κοινοβουλίου. Οι δηλώσεις αυτές, συνάδελφοι, είναι ανάρμοστες. Δεν επιτρέπονται στον πρόεδρο του πρώτου διακρατικού κοινοβουλίου της ανθρωπότητας. Τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, ε, το οποίο ακριβώς ιδρύθηκε, ώστε στην Ευρώπη να μην ξαναζήσουμε ποτέ την ε, αναβίωση τέτοιων φασιστικών καθεστώτων που οδήγησαν σε αιματοκύλισμα ολόκληρη την Ήπειρο. Ζητώ λοιπόν το Κοινοβούλιο να καταδικάσει αυτές τις δηλώσεις, να αποσυρθούν οι ή ο πρόεδρος να τις αποσύρει. Καλά, θα καταλάβετε ότι τώρα δεν θα γίνει συζήτηση γι' αυτό. Το λόγο έχει ζητήσει και η κυρία Τσίμερ. Ε, ισχύουν τα ίδια με την προηγούμενη δήλωση ότι σήμερα δεν συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων και βάσει αυτού του λόγου δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Τσίμερ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς εχθές αποφασίστηκε να ματαιωθεί η σημερινή συνεδρίαση τη διάσκεψη των Προέδρων. Εχθές το απόγευμα το έμαθα αυτό το θέμα της ραδιοφωνικής συνέντευξης το οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος Λαμπέρς και σήμερα οπωσδήποτε θα το έθετα στη διάσκεψη των Προέδρων σε περίπτωση που θα συναδρίαζε. Σήμερα το πρωί εξ ονόματος της δικής μου πολιτικής ομάδας για το λόγο αυτό έκανα και μια δήλωση και ένα δελτίο τύπου βγάλαμε ότι ως πολιτική ομάδα απαιτούμε την παρέτηση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι δεν επιτρέπεται. Δεν είναι δυνατόν στην κορυφή ε, του, το, του δημοκρατικά εκλεγμένου κοινοβουλίου ε, που έχει συγκεκριμένη εντολή να αποτρέψει να επανέλθει το μίσος, ο φασισμός και ο αντισημιτισμός και να καθορίζει την ατμόσφαιρα και τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μας. Στην κορυφή λοιπόν ενός τέτοιου κοινοβουλίου να είναι επικεφαλής ένας άνδρας ο οποίος θεωρεί ότι η εποχή του Μουσολίνη δεν είναι τίποτα το φοβερό ότι κάποια στιγμή, από κάποια στιγμή και μετά έγινε φασίστας ο Μουσολίνη, θεωρεί ο κ. Σταγιάννη. Θυμίζω ότι εδώ στο κοινοβούλιο, εδώ στο κοινοβούλιο υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι γονεί, πατεράδε πατεράδες, μητέρες, φυλακίστηκαν ήδη από τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνηση Μουσολίνη. Και εδώ στο κοινοβούλιο πάντα αναφερόμαστε στο Σπινέλη και σε άλλους. Ε, με το μανιφέστο του Βεντοτένε που έβαλαν τα θεμέλια για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη συνθήκη της Ρώμης. Κυρία Τσίμερ, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τσίμερ, όχι κυρία Τσίμερ, διακόπτει ο Πρόεδρος την κυρία Τσίμερ. Κυρία Τσίμερ, δεν έχετε πια το λόγο. Δεν έχετε πια το λόγο, κυρία Τσίμερ. Σας ανακαλώ στην τάξη. Κυρία Τσίμερ, σας ανακαλώ στην τάξη. Δεν έχετε το λόγο. Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων εκλέγονται διότι έχουν ιδιαίτερε ικανότητε, αλλά μεταξύ αυτών των ικανοτήτων είναι η τήρηση του χρόνου. Μιλήσατε περίπου δύο λεπτά. Ο κύριος Βάιντεν Χαλτσέρ εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της ομάδας του κύριο Μπούλμαν, πάλι για το ίδιο θέμα της διάσκεψης των πρόεδρων. Σας παρακαλώ να με ακούσετε. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Ταγιάννη εχθές έκανε ενοχλητικές δηλώσεις για το ρόλο του Μουσολίνη και πολλοί το θεωρούν σχετικοποίηση αυτών των σκοτεινών περιόδων της Ιταλικής ιστορίας. Ε, και δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που το κάνει ο πρόεδρος με ε, ίδιες ερμηνείες της ιστορίας δημόσια. Όλα αυτά δεν συνάδουν με τη βασική μας αντίληψη και αντιτίθεται ε, στο υπερκομματικό ε, του θόκου του Πρόεδρου. Ο Ούντο Μπούλμαν το επέκρινε και χτες. Γι' αυτό ζητούμε από τον Πρόεδρο αμέσως να λάβει θέση λεπτομερώς για τις δηλώσεις τους αυτές και επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω βήματα. E Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Κονσάλεθ Πόνς. Πρόεδρε, υπάρχει ένας νόμος που διέπει τον πολιτικό που είναι σε προεκλογική εκστρατεία και λέει μην το αφήσεις την αλήθεια να καταστρέψει μια καλή συζήτηση. Η αλήθεια λοιπόν είναι... Κοιτάξτε. Κυρία Φορέντσα, παρακαλώ να καταλήψετε αυτή τη θέση. Φύγετε παρακαλώ από μπροστά μου. Εγκαταλείψτε παρακαλώ αυτή τη θέση. Κύριε Γκονσάλε Πόντ, παρακαλώ συνεχίστε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα νόμο για τον πολιτικό που είναι σε προκλογική εκστρατεία που λέει μην αφήσει την αλήθεια να σου καταστρέψει μια καλή συζήτηση. Αλλά και ενό λαϊκιστή που λέει μην αφήσει την αλήθεια να σου κλέψει ένα καλό θέαμα. Η δικιά μου λοιπόν πολιτική ομάδα, το ΕΛΚ, καταδικάζει χωρίς καμία επιφύλαξη το φασισμό, το φραγκισμό τον ε, εθνικισμό και τον ε, κομμουνισμό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία όσον αφορά την θέση της δικιάς μου πολιτικής ομάδας. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ένας δημοκράτης και μέχρι χτες και σήμερα και θα είναι και αύριο. Όλοι γνωρίζουμε, η πλειοψηφία εδώ πέρα τον ψηφίσαμε και όλοι τον ε, θέλαμε σαν πρόεδρο και είδαμε πόσο καλά προεδρεύει των συνεδριάσεών μας. Και ο Ταγιάννη συμμερίζεται, όπως ε, είπα, με την κοινοβουλευτική μας ομάδα ολόκληρη, την καταδίκη του φρακισμού, του φασισμού, του κομμουνισμού και του εθνικισμού. Εγώ τον άκουσα που αντιτάθηκε ο συνάδελφος εδώ στη συζήτηση για τη Βενεζουέλα και προτιμά να μιλήσουμε για τα ψάρια στην υδατοκαλλιέργεια. Τον άκουσα. Κατόπιν τούτον. Όλοι μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος όταν μιλάμε στα μέσα ενημέρωσης και όλα τα μέσα μπορούν να στρεβλώσουν κάπως αυτά που λέμε. Ο κύριος Σταγιάννη εξήγησε κάτω από ποιες συνθήκες είπε τα λόγια αυτά και ότι δεν στηρίζει το φασισμό. Συνεπώς, δεν έχουμε... Ευχαριστώ, Πρόεδρος Διακόπτη, τον ομιλητή. Δεν θα φέρουμε εδώ την προεκλογική εκστρατεία. Ε, κύριε Γκονσάλης Πόνς, δεν έχετε πια το λόγο. Δεν έχετε πια το λόγο. Δεν έχετε πια το λόγο, τρίτη φορά. You do Κοιτάξτε, τρία λεπτά σχεδόν σας ακούμε. Η κυρία... Ε, ζήτησα από την κυρία Τσίμερα να σταματήσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση τώρα μακρά για αυτό το θέμα. Επέτρεψα να γίνει αυτή η μικρή συζήτηση, διότι δεν συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων. Για τους υπολείπους όλους, η κυρία Φορέντσα, δεν περιστέλνει τα δικαιώματά σας. Μην ανησυχείτε. Να μας πείτε σε ποιο άρθρο βασίζεται η ομιλία σας. Αλλιώς θα σας αφαιρέσω το λόγο. Ποιο άρθρο επικαλείστε του κανονισμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώην άρθρο 21. Ήθελα να πω ότι και εσείς αδικείτε το λειτουργήμά σας ε, ως προεδρεύοντας αυτής της ολομέλης αυτή τη στιγμή. Διότι είναι σοβαρότατο αυτό που συνέβη χθε και είναι πολύ σοβαρότερο από τον ίδιο τον ιστορικό κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου. Να θυμίσω μόνο ότι το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία ε, ξεκίνησε με την ε, φανταστική ομιλία ε, που έλεγε ότι θα μεταμορφωθεί το κοινοβούλιο σε ένα χώρο... Κυρία Φορένσα, σας αφαιρώ το λόγο. Δεν έχετε πια το λόγο. Κλείνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Και δεν θα βελτιωθούν τα πράγματα αν φωνασκείτε. Σας έχω κλείσει το μικρόφωνο. Δεν έχει νόημα να φωνασκείτε. Σα εξήγησα σαφώς ποιους κανόνες εφαρμόζω. Είναι στη διακριτική ευκαιρία του Προέδρου, του Προεδρεύοντα και σας είπα ότι σήμερα δεν έγινε η διάσκεψη στον Προέδρο, γι' αυτό δίνω λίγο χώρο στους επικεφαλείς των ομάδων. Κατά τα άλλα μόνο βάσει κανονισμού. Για να μην ε, διανυστεί η σύντομη συζήτηση που έγινε. Η κυρία Μιράντα ζήτησε το λόγο ε, ε, επί του κανονισμού. Ισχύει ακριβώς το ίδιο και για σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε απαιτώ σεβασμό και ησυχία. Τα λόγια του Προέδρου Ταγιάννη διακόπτη. Όχι κυρία Μιράντα, ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για σας. Αυτό ακριβώς δεν θα κάνουμε. Δεν είναι θέμα σεβασμού, δεν έχετε το λόγο πια, καθίστε παρακαλώ. Δεν έχετε πια το λόγο. Καθίστε παρακαλώ. Κυρία Μιράντα, δεν είναι θέμα σεβασμού αυτό. Έχω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για άλλα τα μελήματα, αλλά εδώ πρόκειται μόνο περί του κανονισμού. Άλλος, για τον κανονισμό. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Πρόεδρε, βάζει το άρθρο 1 του κανονισμού. Να πάμε στις ψηφοφορίες επιτέλους. Να περάσουμε στην κανονική μερίσια διάταξη. Κύριε Κάρβερ, αυτό ήταν για τον κανονισμό. <laughs> Παρακαλώ, ε, όλα αυτά θα πάρουν και άλλοι συνάδελφοι που το ζητούν επί του κανονισμού το λόγο. Κύριε Σόσνιερτς. Πολύ σύντομα κι εγώ. Εντάχει να πω ότι αν μιλάμε για δημοκρατία και θέλουμε να βάλουμε στην ίδια φράση και τον Αλτιέρο Σπινέλη, δεν μπορεί να ακούγεται το όνομα του Σπινέλη, διότι... κύριε συνάδελφε Σόσνιερς, τώρα δεν θα κάνουμε ερμηνείες της πολιτικής. Κανονισμός είναι το θέμα. Κύριε Φερχόφστατ, μια στιγμή, κύριε Φερχόφστατ, μη βιάζεστε. Κύριε Φερχόφστατ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Φερχόστατ. για αυτό το θέμα και δεν ήταν και διάσκεψη των Προέδρων σήμερα, όπως σας είπα. Μόλις ακούσουμε τους υπολείπους επί του κανονισμού, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φερχόφστατ. Άλλος. Κυρία Ζανή. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σοβαρά, κυρίαρχα και σύντομα. Σας ενημερώνω ότι σήμερα θα ψηφίσουμε ψήφισμα που έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος διακόπτει και κλείνει το μικρόφωνο. Τώρα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Σας αφαιρώ το ε, λόγο. Δεν ζητήσατε το λόγο βάσει κάποιο άρθρο του κανονισμού. κύριος Βιώτη. Βάσει του άρθρου 21 και μην μου κόψετε το λόγο, διότι ο πρόεδρος Ταγιάννη είναι Ιταλός και χθε προσέβαλε τον ευρωπαϊκό λαό και τον Ιταλό της μας. Ε, τον λαό της χώρας μας. Όχι κύριε Βιώτη, δεν το επιτρέπω ούτε αυτό. Δεν υπάρχει εδώ άρθρο 21 σε αυτή την περίπτωση. Δεν αρκεί να επικαλείστε το άρθρο 21. Λοιπόν, δεν είναι επί του κανονισμού αυτό το αίτημα. 5, 9, 7 στο έδρανο αυτό κάποιο συνάδελφο ζητεί το λόγο. Ε, Κυρία Ατζέα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να θυμίσω ότι το φασιστικό καθεστώς στην Ιταλία... Κλείνει το μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Δεν επιτρέπω ούτε αυτή την παρέμβαση. Δεν έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο σας έχει σβήσει. Παρακαλώ καθίστε. Αλλιώς θα πρέπει να σας ανακαλέσω στην τάξη. Κυρία Αζέα, καθίστε σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, δεν ακούγεστε. Παρακαλώ καθίστε. Από ό,τι φαίνεται τώρα δεν έχουμε πια ε, αιτήματα που να αφορούν πραγματικά τον κανονισμό. Δίνω το λόγο και πάλι, ε, πάλι μάλλον στον κύριο Φερχόφστατ. Ε, Mr. Πρόεδρε, Πρόεδρε, ο Έστεβαν Πόντς νομίζω ότι είχε δίκιο όταν είπε πριν από λίγα λεπτά ότι είναι ανόητο από κάθε πλευρά να κάνουμε εδώ αυτή τη συζήτηση και να το μπερδεύουμε με την προεκλογική εκστρατεία μέσα στην οποία φαίνεται ότι κάποιοι ήδη βρίσκονται. Πρέπει όμως να σας πω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε ο πρώτο μάλλον που πρέπει να το κάνει αυτό είναι ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Να μην αρχίζει τέτοια ιταλική προεκλογική εκστρατεία, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα εδώ σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο, και θα τελειώσω με αυτό, σα ζητώ, Εσά που προεδρεύετε εδώ σήμερα, βάσει του κανονισμού μα, να ζητήσετε από τον πρόεδρο να αποσύρει αυτά που είπε, να ζητήσει συγγνώμη για αυτά και δεύτερον να αρχίσουμε μέσω το έργο μας εδώ στην Ολομέλη. Αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, κανονικές εργασίες τώρα. Κύριε συνάδελφε, κύριε Φερχόφστατ, λαμβάνω υπόψη την πρότασή σας και φυσικά θα ενημερώσω τον Πρόεδρο για όλα όσα συμβαίνουν εδώ. Αλλά ε, προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καζακστάν. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επόμενο ψήφισμα για το Ιράν. Κοινό ψήφισμα επτά πολιτικών ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γουατεμάλα. Ένα ψήφισμα από επτά πολιτικές ομάδες. Η, ε, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Τσεκ! Ωραία, θα την ελέγξουμε. Τη 2, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Τσιέφκα. Είναι μία ονομαστική ψηφοφορία για όλη την έκθεση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Φιέλνερ. Και πάλι μία ονομαστική ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση της κυρίας Δελάνγκε και του κυρίου Γουαλτιέρη. Ε, το λόγο ζήτησε ο συνάδελφος Μακάρθη. Ματ Κάρθη. Μικρό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βάσει του άρθρου 59 παράγραφος 3 θέλω να ζητήσω να ψηφίσουμε για την ψηφοφορία των τροφολογιών. Πρέπει να πω ότι οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ ε, εμπόδισαν τις υπόλοιπες ομάδες να έχουν το δικό τους λόγο σε αυτό το πακέτο και να επηρεάσουν τον κατάλογο των ψηφοφοριών. Θα ήθελα να γίνει λοιπόν με ονομαστική κλίση η ψηφοφορία για να περάσουν αυτέ τι τροπολογίε που θα επιτρέψουν να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου ιδιοκτήτε των σπιτιών του να γλιτώσουν από τι εξώσει. Ο κύριο Κάρθη προτείνει να ψηφιστούν οι τροπολογίε. Θέλει κανεί να μιλήσει κατά ο κύριο Γκουαλτιέρη. The uh, adopted has been... Το κείμενο που έχουμε μπροστά μας εγκρίθηκε με ευρία πλειοψηφία. Το συζήτησα και με τον κύριο Γκίγκολ την περασμένη φορά. Το κείμενο αυτό είναι ιδιαίτερα ήπιο και καθόλου έντονο. Τώρα μας κατηγορείται για το αντίθετο. Είναι ένα φοβερά καλά εξισορροπημένο κείμενο που ακριβώς θα παρεμποδίσει αυτά που λέτε τις εξώσεις να γίνουν. Εγώ ενθαρρύνω να το υπερψηφίσετε όπως εγκρίθηκε και στην Επιτροπή μας. Με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε το αίτημα του κυρίου Κάρθη. Ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Προχωρούμε. Ψηφίζουμε την προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 2, αρχίζει τώρα ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ολοκληρώνεται εδώ η πρώτη ανάγνωση και περνούμε στην έκθεση του κυρίου Πίπερ. Η τροπολογία 62 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Είναι επί της προσωρινής συμφωνίας. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται ολοκληρώνεται ούτως η πρώτη ανάγνωση έκθεση Χούλμαγια. Θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθήσαμε όλες αυτές τις πολυάριθμες τροπολογίες που πρέπει να ψηφίσουμε ονομαστικά, να τις συνοψίσουμε, unblock δηλαδή. Δυστυχώς δεν συμφώνησε η ομάδα που είχε κατέθεσει τις, τροπολογίες. 16 ε, υπέρ κατά αποχές ε, Απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα έχουμε πάρα πολλές ονομαστικές ε, ψηφοφορίες. Η τροπολογία 29. Δεν θα λέω κάθε φορά ότι είναι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 30. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 31 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο αρχίζει η ψηφοφορία. Και αν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 32, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 33, η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 34, Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 35, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 36, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 37, αρχή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 38, αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία 39, αρχή ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 40 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 41, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 42, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Α, πέρασε. Απορρίπτεται. Η 43, άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισε τον όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται 47, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 48, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέρ, αυτή δεν είναι ονομαστική, κατά αποχές απορρίπτεται. Επανερχόμαστε στις ονομαστικές. Η τροπολογία 17 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, αρχή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τρία ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 21. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 22. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 23. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 11 ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 18. Το αρχικό κείμενο ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψήφισαν όλοι, λίγοι. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 13 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία εάν ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται η παράγραφος 27 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 6 υπέρ. Τι θέλετε, έλεγχο. Ε, στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου 27 αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 28, το αρχικό κείμενο ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 14, μάλλον μετά την παράγραφο 28 είναι η τροπολογία 14, ονομαστικά την ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Η 26 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 25, με ονομαστική κλίση και πάλι, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Β, το αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Να ψήφισαν όλοι. Πέρας εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στις προτάσεις ψηφίσματος για την ισορροπία των φύλων. Είναι κοινή πρόταση ψηφίσματος από πέντε πολιτικές ομάδες. Τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4, ονομαστική. Η ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 6 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τη λογική σκέψη M. Ε, το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο όπως τροποποιήθηκε, όλο το ψήφισμα δηλαδή, με ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία και αν όλοι ψήφισαν, λίγοι. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα σε άλλη, μάλλον σε ένα αίτημα για το, κανονισμό για την αναβολή ε, διορισμού ε, ε, ενός νέου μέλους του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, αναβολή της προφορίας, το λόγο έχει ο κύριος Γκίγκολτ, εξ ονόματος ομάδας των Πρασίνων. Πρόεδρε, συνάδελφοι, στο όνομα των Πρασίνων και βάσει το άρθρο 191 του ιστορικού κανονισμού, θα ήθελα να ζητήσω να αναβληθεί η ψηφοφορία των δύο εκθέσεων αυτών. Διότι τα τελευταία χρόνια και με το τελευταίο ψήφισμα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα ζητήσαμε μόλι περισσότερη ζώτα των φύλων στι ύψιστε θέσει οικονομική ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ω εξή. Στο εκτελεστικό ε, όργανο τη Κεντρική Τράπεζα έχουμε μία γυναίκα και πέντε άντρε. Στο Γενικό Συμβούλιο τη ΕΚΤ έχουμε μία γυναίκα και 22 άντρε στο, ε, ταμείο, στο μηχανισμό εξυγίανσης έχουμε μία γυναίκα, πέντε άντρες. Και το ίδιο επαναλαμβάνεται και στα υπόλοιπα όργανα και φορείς. Γι' αυτό λοιπόν το ερώτημά μου είναι το εξή. Πόσο καιρό θα περιμένουν οι γυναίκες στο Ευρωκοινοβούλιο να τους εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες και απλώς να υπόσχεται και να περνάει τον ένα διορισμό μετά τον άλλο που τον δίνει σε άντρε. Ως εκ τούτου, ως εκ τούτου Συνάδελφοι, η διάσκεψη των Προέδρων έχει συντάξει δύο επιστολές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και έλαβαν από, ε, απαντήσεις τελείως ασαφείς, με επεκφυγές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκίγκολτ. Διακόπτει τον ομιλητή ο Πρόεδρος, ο κύριος Γκουαλτιέρη, για να μιλήσει κατά το αιτήματος αυτού. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσα απλώς να πω ότι στην ψηφοφορία που μόλις έγινε και στο ψήφισμα είχαμε 407 που αποφάσισαν έναντι 104 για το θέμα της αναβολής. Και γιατί ήταν τόσο ευρία αυτή η πλειοψηφία και ήθελε να μην αναβληθεί η ψηφοφορία, διότι η αναβολή της ψηφοφορίας ε, είναι κακή απάντηση στο σωστό ερώτημα. Το θέμα που επισημαίνεται είναι απόλυτα σωστό και είναι και ο λόγος για τον οποίο στο ψήφισμα αυτό έχουμε καθορίσει ένα πρόγραμμα δράσης για να αυξηθεί ο ρυθμός των γυναικών που θα εκπροσωπούνται στις κορυφαίε οικονομικές θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό συζητούμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο και περιμένουμε και καλύτερη απάντηση στις επιστολές μας και καλύτερο σχέδιο για το μέλλον. Ε, όμως, εάν κοιτάξετε το συγκεκριμένο αίτημα του κυρίου Γκίγκολτ, ε, είναι λανθασμένο και μπορώ να σας εξηγήσω ε, γιατί με πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί να αναβάλουμε το διορισμό του κυρίου Λαβιόλα. εγκρίθηκε από 88% των μελών της Επιτροπής μας. Έχει τα προσόντα. Είναι μέλος ενός, θα γίνει μέλος ενός οργανισμού που προεδρεύει γυναίκα και ότως άλλως όλα τα μέλη προτάθηκαν είχαν και γυναίκες υποψηφίου. Ε, στον κατάλογο των ψηφίων. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη. Και τα δύο ε, αυτά ε, θέματα έπρεπε να τα εξηγήσετε μέσα σε ένα λεπτό και τα καταλάβαμε και τα δύο. Και αυτό που θέλετε να πείτε εσείς και αυτό που ήθελα να πει και ο κύριος Γκίγκολτ. Και είστε παλιέ καραβάνε εδώ, κανονικά και οι δύο θα έπρεπε να το γνωρίσατε ότι έχετε ένα λεπτό. Λοιπόν, προχωρούμε. Ονομαστική ψηφοφορία του αιτήματο του κυρίου Γκίγκολτ. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Άρα θα ψηφίσουμε για την πρώτη έκθεση του κυρίου Γουαλτιέρη, διορισμός του Σεμπαστιάνο Λαβιόλα. Είναι μυστική η ψηφοφορία και ε, με βάση το άρθρο 180 παράγραφος 2 του κανονισμού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ακολουθεί η επόμενη ε, έκθεση Γουαλτιέρη, ιδρυσμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και πάλι μυστική ψηφοφορία για τον κύριο Φίλιπ Λέιν. Αρχίζει τώρα η μυστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται επίση. Και τελευταία έκθεση, ε, Γκουαλτιέρη, διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Πρόκειται για το διορισμό του κυρίου Ζωζέ Μανουέλ Κάμπα. Ε, και εδώ είναι μυστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα, Ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 2 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 6 το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά απόχέ εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Επόμενο ψήφισμα. Το επίγον τη κατάρτιση ενωσιακή μαύρη λίστα τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο. Έξι πολιτικέ ομάδε έχουν καταθέσει ένα ψήφισμα. Όλο το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε. Κλιματική αλλαγή. Προτάσει ψηφίσματο. Από έξι πολιτικέ ομάδε έχουμε ένα ψήφισμα. Ε, Ανομαστική ψηφοφορία για την ε, τροπολογία να αρχίζει. Ε, αν ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Ε, η τροπολογία 14, ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 12 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον ονομαστικά πάντα. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας. εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 16 δύο Το πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο καταπίπτει. Η τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Είμαστε στην τροπολογία παρήθμου 12. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Παράγραφος 8 του αρχικού κειμένου ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Η παράγραφος 16, 12 ήταν η τροπολογία, 16 είναι η παράγραφος. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 9, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για την τροπολογία 9, παρακαλώ, ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει τώρα. Ψηφίσαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Παράγραφος 17. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτο είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 ερμενομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 20 το αρχικό κείμενο, παράγραφος 20, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25-26, δύο τροπολογίες ονομαστικά αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε το αρχικό κείμενο καταπίπτει. Παράγραφος 25 αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 με ονομαστική κλίση, η οποία αρχίζει τώρα. Εάν ψήφισαν όλοι. Λίξ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 27, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 27 έχουμε την ε, τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 17 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 28 σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 7 με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 31 του αρχικού κειμένου σε δύο τμήματα. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. 32 μάλλον, όχι 31. Έκανα λάθος, λέει ο πρόεδρος. Στην 32 ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. 32 πρώτο τμήμα ονομαστικά. Έκανα λάθος, είπα 31. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου 32, ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εάν ψήφισαν όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα επιστρέφουμε στην παράγραφο 31. Ψήφι κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 20. Σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον, ονομαστικά, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπέφτει. Παράγραφο 34, το αρχικό σε δύο τμήματα, το τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται, το δεύτερο υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 21 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Επόμενη. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 35 Θέλετε να ελέγξουμε την 22, ωραία, ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία παριθμών 22. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η, ε, παραγράφος 35, το αρχικό κείμενο, ονομαστικά, το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 36. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 23. Τροπολογία με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πού είμαστε τώρα. Ε, Παράγραφο 42 του αρχικού κειμένου. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφο 44. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 48. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, δέκα 10 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 55 το αρχικό τμήμα. Υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Η ε, τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 56 το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η παράγραφος 57 το αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίθηκε η τροπολογία 5 υπέ. Κατά. Αποχές. Εγκρι... Η παράγραφος 58, το αρχικό κείμενο με ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα. Ψηφίσαν όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 6 ονομαστικά ψηφίζουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. Παράγραφος 6, το αρχικό κείμενο, σε δύο τμήματα, ονομαστικά και τα δύο, ψηφίζουμε το πρώτο. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα, άρχεται ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 64 τροπολογία 8 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 65 το αρχικό κείμενο υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 66 το αρχικό κείμενο υπέρκατα αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα και τροπολογίε. τροπολογίες. Περνάμε τώρα στο ψήφισμα συστάσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΠΑ. Η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου έχει ένα ψήφισμα. Για διαδικαστικό η κυρία Ζανέ ζητεί το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βάσει του άρθρου 108 για τις εμπορικές συμφωνίες και σε σχέση με την επανάληψη των διαπραγματεύσεων αυτών με τις Ηνωμένες Πολιτείες θέλω να ενημερώσω τους συναδέρφους ότι πρόσωπος ο Αμερικανός εμπορίου είπε ότι μια τέτοια συμφωνία είναι αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς τη συμπερίληψη της Γεωργίας. Ήθελα να σας το πω αυτό. Κυρία Ζανέ, αυτό δεν ήταν διαδικαστικό τώρα το έτοιμά σας. Και αν επαναληφθεί, θα σας ανακαλέσω στην τάξη. Ψηφίζουμε. Η τροπολογία 8, ονομαστικά, αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 34, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι τροπολογίες 2, 23 και 15 ταυτίζονται. Ψήφι υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτονται. Η τροπολογία 9 ονομαστικά. Θέλετε να ελέγξουμε, ωραία, τις τρεις αυτές τροπολογίες που ταυτίζονται, 2, 23, 15, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Α, πέρασε. Mm, απορρίπτεται. Ισοψηφία. Η τροπολογία 9. Αρχίζει η ψηφοφορία νομαστική. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογίες 3, 16, 24 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Ε, μάλλον η ίδια πλειοψηφία θα είναι. Ας το ελέγξουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίζετε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 ε, ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 11 ονομαστικά. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Antrag 36 dafür. Η 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 38 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17 και 25 ταυτόσημες ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 39 ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Αποχές. Ωραία, να το ελέγξουμε. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμού 39. Die Πέρασε ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Abgelehnt. Herr Kollege, die Flieger sind nicht Απορρίπτεται. Πηγαίνουν 40 ψήφοι υπέρ, κατά. Αποχέσα. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 43 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 44 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίφθηκε. 18. Ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4, 12 και 26 ταυτόσιμε σε δύο τμήματα και ονομαστικά. Πρώτο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι Πέρασε. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέραση όλοι ψηφοφορια Απορρίπτεται. 5, 13, 27 ταυτόσημες με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στο πλαίσιο 6, 14, 22, 28, που είναι ταυτόσιμε σε δύο τμήματα με ονομαστική κλίση. Άρχεται το πρώτο, για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 ψήφι υπέρ. Κατά. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται ένα υπέρ. Να ελέγξουμε τη 32 άρχεται ψηφοφορία. 32 wird überprüft. Haben alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 33 υπέρ. Κατά εποχές απορρίπτεται. Επτά ονομαστικά άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ψηφ, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ονομαστικά το σύνολο. Ψηφίσατε όλοι. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Äh, Και πηγαίνουμε στην έκθεση Σίλβα Περέρια Μάνκα για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. 25 ονομαστικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 5 και 17 ταυτόσημες ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 15 ψήφι υπέρ. Κατά. Ποχές. 16 υπέρ. Κατά. Ποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. ποχέ. Απορρίπτεται. 6. Ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 20 πέρ; Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 21 ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22 ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 23 ψήφι πέρα κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται 14 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται 3 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται 4 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συνολικά ψηφίζουμε ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πηγαίνουμε στο ψήφισμα για την κατάσταση στην Νικαράγουα. Δι... Σε δύο τμήματα, ε, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το επόμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματο. άρχεται ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση της συναδέλφου Θεοχάρου και Γκάμπους για την ετήσια στρατηγική έκθεση για την υλοποίηση και την επίτευξη των βιώσιμων στόχων ανάπτυξη. Τροπολογία 5. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20. Παράγραφος 20. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος Θέλετε να το ελέγξουμε για την παράγραφο 20 το αρχικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Παράγραφο 22 του αρχικού κειμένου. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχέ. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά απόχέ Εγκρίνεται. Τροπολογία 23 αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά Αποχέ. Εγκρίνεται. 24 αρχικό κείμενο. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 ε, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ας, προσπα... Ας ε, ελέγξουμε την 27 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 3 είμαστε. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 29, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 32, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 49, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, Ας το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 49. Ψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 49, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56, αρχικό κείμενο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Q. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη U σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πριν φτάσουμε στην τελική ψηφοφορία, σας ευχαριστώ ε, για την τήρηση του χρόνου σας και επειδή έχουμε και τις επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλούμε να αποχωρήσουμε ε, ησύχως από την αίθουσα. Τώρα ψηφίζουμε και το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου και ζητώ από τον συνάδελφο Ντόρφαμαν, τον συνάδελφο Καρά, ε, Ιάκοψεν Φερχόφστατ, Ερτούγκ. Σας παρακαλώ όλους να αποχωρήσετε ταχαίως και ησύχως. Λοιπόν, αρχίζουμε την αιτιολόγηση ψήφου για την έκθεση ΡΕΝΤΑ για το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας Εθνικά Κέντρα Συντονισμού. Συνάδελφος Φαν Μπρέμπτ. ο συνάδελφος Κάρας και με την κυρία Γκρέσλε μαζί. Παρακαλώ ησυχία. Και εσείς συνάδελφε Γκροστέτ, παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Η κυρία Χάρκιν έχει το λόγο. Όχι, δεν είναι παρούσα. Δεν είναι εδώ η κυρία Χάρκιν. Περνάμε στην κυρία Σπυράκη. Ε, ούτε η κυρία Σπυράκη. Συνάδελφος Σόσνιετς. Αυτό που προτείνεται εδώ είναι ένα βήμα που το ώστε θα κάνει το ίντερνετ ε, να εξαρτάται τα κράτη. Ε, τελικά εδώ καλούνται οι ευρωπαϊκές αρχές να τονώσουν την έρευνα και τελικά όμως αυτή η έρευνα θα χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει την παρέμβαση των κυβερνήσεων στο διαδίκτυο. Η δωρεά εμποδομών θα οδηγήσει στην κατάσταση όπου θα υπάρχει ε, κάποια δικαιολογία να ομαδοποιούνται τα δίχτυα που, που κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά χρήματα. Οι εταιρείες που θα επιδοτούνται θα εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις, ποτέ δεν θα είναι κερδοφόρες, γιατί θα δίνονται όλες και περισσότερες επιδοτήσεις. Θέλουμε λοιπόν ανεξαρτησία, δεν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει τον, τη λειτουργία του ίντερνετ. Ευχαριστούμε. Πηγαίνουμε στην έκθεση Πύρη για την έκθεση του 2018 για την Τουρκία. Πρώτη έχει το κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χουσέν Κονακάν, Καραμάν Ντεμίρε, Μουσταφά Ερντέμ, Οσμάν Καρακρέα, Ιουσουφ Κανκάν και πολλοί άλλοι είναι δημοσιογράφοι ή καθηγητές τουρκικής καταγωγής οι οποίοι τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο πέρσι απήχθησαν από το Κωσυφοπέδιο, από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και από άλλες χώρες. Συνολικά, το 2018 είχαμε 18 ανθρώπους που απήχθησαν. Προφανώς, όλες αυτές οι απαγωγές διατάχθηκαν από τον Ερντογκάν με τη συνενοχή των αρχών αυτών των χωρών. Είδα εγώ εικόνες από τις συλλήψεις τους μπροστά σε σχολεία, ή τους πήραν από τα σπίτια τους. Απήχθησαν και μεταφέρθηκαν μέσω αεροπλάνου στην Τουρκία χωρίς έκδοση, ούτε αίτημα έκδοσης. Ήταν καθαρή απαγωγή. Ευχαριστώ όλους εκείνους που υπέγραψαν τις επιστολές για τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ κύριε Μακοβή. Κυρία Σπυράκη. Δεν βλέπω την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Κιουτσούκαρα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πόσπισιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεδομένη τη κατάσταση στην Τουρκία δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση στην κοινωνία η διακυβέρνηση της χώρας ε, που τόσο πολύ διαφέρει από την Ευρώπη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνει την Τουρκία να μην μπορεί να θεωρηθεί υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, πρέπει να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί είναι και μέλο ε, του ΝΑΤΟ. Παρ' αυτά, πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να γίνει μέλος της Ένωσης του και αυτό περιλαμβάνει το ψήμεξο και το υπερψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, κύριο Σόσνιερ, είναι επόμενο. Σε αυτή τη θητεία ε, και μάλλον σε αυτή την, ε, το μήνα έχουμε δύο ε, ολομέλειες εδώ στο Στρασβούργο γιατί είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τα νομοθετικά μας ζητήματα. Μιλάμε για το Τουρκμενιστάν, Καζακστάν, Νικαράγουα, Ρουσία, Ιράν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα ασκούμε κριτική στην Τουρκία. Ενδιαφέρεται κανείς νομίζετε. Αν έχουμε 10 ε, καταγγελίες ε, το μήνα ή τη μέρα, ποιος ενδιαφέρεται πλέον. Ακόμα και δίκιο να έχουμε. Το χάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά είναι διαστρεβλωμένο προς τα αριστερά ε, ε κατά ε, ένταξη των Ρωμά σε βάρος αφρολογουμένων, ε, το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΑΚΟΥ και όλα αυτά, μα όλα για όλα μέσα τα έχουμε στο ίδιο τσουβάλι. Δεν μπορώ να ψηφίσω. Ευχαριστώ. Για να κλείσουμε αυτή την έκθεση, ο κύριος Σκρίπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση συνοψίζει πολλά θέματα που αφορούν την Τουρκία. Αναμφισβήτητα αντιμετωπίζουμε απρόβλεπτο γείτονα. Η τουρκική η κυβέρνηση και ο στατός της συμβολίζει μιζέρια ε, και μαρτύριο για αυτούς που είναι κοντά, που είναι χριστιανοί, Τουρκμένοι, Κούρδοι και, ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει σαφή θέση ως προς της δημοκρατίας απέναντι στην Τουρκία. Γι' αυτό το χριστιανικό πολιτικό κίνημα της Ευρώπης που εκπροσωπώ έκανε ένα αίτημα για να σταματήσουν οι συνομιλίες ε, ένταξης. Αλλιώς θα αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα και θα δείξουμε στις μειονότητες που δεν μας νοιάζει στις κοινότητες της Μέσης Ανατολής, στις μειονότητες. Πρέπει να τους πούμε, το τερματισμό των συνομιλιών ένταξη είναι ισχυρή πολιτική χειρονομία και αξίζει αυτό να το κάνουμε στην Τουρκία. Δεν υπάρχει χρόνος ε, για... Πρέπει να γίνει αυτή η αναστολή όπως αναφέρεται στην έκθεση. Ευχαριστούμε κύριε Σκρίπεκ. Έληξε η επεξήγηση ψήφου για την κυρία Πύρη και τώρα για την έκθεση της κυρίας Χάρκιν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό Οικονομικής Πολιτικής. Η κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήμουν υπέρ της έκθεσης αυτής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Συντονισμό Οικονομικής Πολιτικής. Εψήφισα υπέρ κυρίω διότι το θέμα τη ανεργία είναι ένα θέμα που δεν θα πρέπει να σταματήσει να μα απασχολεί. Παρότι αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται, παρατηρείται ανάπτυξη, συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά εργασία στην Ευρώπη. Υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ στην απασχόληση και στα επίπεδα των μισθών μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Και θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι στο μέλλον θα υπάρξει κάποια κρίση, μια κρίση αυξημένης ανεργίας με προκλήσεις ε, που θα οφείλονται παραδείγματο χάρη στην αύξηση τη αυτοματοποίηση. Σε παραλληλισμό και με τον γυράσκοντα πληθυσμό αυτό μπορεί να μα οδηγήσει σε κρίση. Γι' αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσο η πολιτική μα είναι ανθεκτική και για το μέλλον. Είναι απαράδεκτο το υψηλό επίπεδο φτώχεια μεταξύ των εργαζομένων μα 9,6% αυτή τη στιγμή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι διαφορέ μεταξύ μισθών ανδρών και γυναικών επίση πρέπει να μειωθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία ε, λίγη επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Χάρκιν και περνάμε στην επεξήγηση ψήφου για, τον, για την έκθεση Φιέλνερ για την υλοποίηση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων. Η συνάδελφος κυρία Σιόντροβα. Ευχαριστώ. Ήμουνα υπέρ της εκθέσεως για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Συμφωνώ με τη σημασία που έχει το σύστημα διότι είναι εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε να μειώσουμε την φτώχεια στι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε μέσω διεθνού εμπορίου. Συμφωνώ με τη σύσταση για μελλοντική αναθεώρηση του παρόντο συστήματο και θα ήθελα να τονίσω ότι οι τομεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι η θέση των γυναικών στι χώρε που είναι δέκτε τη υποστήριξη μέσω του συστήματο. Θα ήθελα να τονίσω από τη μία πλευρά ποια είναι η κατάσταση των ανδρών και των ανθρώπων και την άλλη τα ανθρώπινα δικαιώματα τη θέση των γυναικών μάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την οικονομική θέση των γυναικών. Παρ' όλα αυτά, οι γυναίκε ακόμα είναι στόχο σε κάποιε χώρε και δεν είναι καλέ οι συνθήκε εργασία του. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική σύσταση στην έκθεση αυτή που υποστηρίζει και ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντο επίση αυτέ τι χώρε. Ευχαριστούμε κύριε Σόντροβα. Η κυρία Ward. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς βελτιώνει τις πολιτικές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εμπορικές συμφωνίες. Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για τους εμπορικούς δασμούς ε, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τονίζει τι δυνατότητες που έχει το GSP Plus να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, ε, ανάπτυξη καταπολεμώντας την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παιδική εργασία. Το πρόγραμμα αυτό έχει ε, πολλές δυνατότητες ε, και με την έκθεσή μας ε, προσπαθούμε να ζητήσουμε και βελτιώσεις. Αυτό είναι στο πλαίσιο του Δεσμευτικού Μηχανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εμπορικές συμφωνίες, όπως ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο μας τον Οκτώβριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα για να προωθήσει την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πρέπει να αποδυναμώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα στις εμπορικές συμφωνίες. Και αυτοί που είναι υπέρ του Brexit θέλουν το εμπόριο πάση θυσία. Εκατομμύρια πολιτών, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Ward. Ολοκληρώσαμε την επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Φιέλνων και περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου για τους διορισμού σε θέσεις οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ισότητα των φύλων. Κυρία Κομπούλα Νάντρη. Ευχαριστώ. 30% γυναικών έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν διορίζουμε ανθρώπους διάφορες θέσεις, οι πολίτες δεν έχουν άμεση εμπλοκή. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τους διορισμούς υψηλές θέσεις. Παράγματος χάρη, Σήμερα διορίσαμε τρεις άνδρες για σημαντικές θέσεις στην Ευρώπη. Πριν από αυτό μιλήσαμε για το πώς θα βελτιώσουμε τη θέση των γυναικών. Και όταν γίνονται αυτοί οι διορισμοί μέσω καταλόγους, θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνει στον κατάλογο ένας άνδρας και μια γυναίκα. Επί του παρόντος, η κατάσταση των την ισορροπία των φύλων δεν είναι καλή. Έχουμε 11 θεσμικά όργανα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο δύο από αυτά έχουν επικεφαλής γυναίκε. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μακριά από τον ε, στόχο. Μόνο εννέα επίτροποι είναι γυναίκες, αλλά ποτέ δεν υπήρξε πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής γυναίκα. Αυτή η κατάσταση αλλάζει πολύ αργά, με πολύ αργό ρυθμό. Θα πρέπει να ληφθούν δραστικά μέτρα τόσο ώστε να αλλάξει, να σπάσει αυτή η γυάλινη οροφή και να βελτιωθεί η ισορροπία των φίλων. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κυρία Κομπουλανάτρη και επόμενος ο κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού τελικά. Παρότι, όπως ήδη είπα κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα αυτό, όπου συζητήσαμε υποψηφίους για τρεις σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κατάλογο ε, των ε, υποψηφίων που έχουν παραμείνει, τόνισα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, η ομάδα μας υποστηρίζει την ισότητα των φύλων στην επιλογή υποψηφίων, αλλά παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε και την γεωγραφική ισορροπία. Οι υποψήφοι από την Παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση, την αποκαλούμενη Παλαιά Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να είναι η προτιμόμενη και η διαδικασία αυτή θα πρέπει να αφορά και τους υποψηφίους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε 19 άνδρες υποψηφίους και μόνο 9 γυναίκε υποψηφίου. Τελικά όμως ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιοτρόφσκι και περνάμε τώρα στι επεξηγήσεις ψήφου για ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τις κυρώσεις για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Πιοτρόφσκι και πάλι. Έχουμε λοιπόν ένα κοινό ψήφισμα για τις μελλοντικέ κυρώσεις και το σχετικό σύστημα για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να παγώσουμε τα στοιχεία εσωτερικού και να απαγορεύουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων εκείνων των φυσικών προσώπων ή φορέων που είναι υπεύθυνοι για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστηματικά να εφαρμόζουν ε, τη διαφθορά. Θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικό το νέο σύστημα, αλλά δεν είμαι πεπισμένο. Ανησυχώ με την ιδέα που για αυτό το σκοπό τα κράτη-μέλη πρέπει να ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο την χρήση των ε, κυρώσεων. Παρά αυτή την επιφύλαξη, τελικά εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα. Ευχαριστώ πολύ. Πηγαίνουμε στο επόμενο θέμα για την κλιματική αλλαγή. Κυρία Μιράντα, έχει καταρχάς το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχθηκε εδώ πολλούς ε, νέους, πολλούς εφήβους ε, οι οποίοι αγωνίζονται κατά της κλιματικής αλλαγής. Ε, μια πολύ ευπρόσδεκτη μάχη που δίνεται και η οποία και αύριο στο δρόμο θα πει ξεκάθαρο ότι πρέπει σε όλη την Ευρώπη να γίνει αυτή η μάχη για το κλίμα, για τον καθαρό αέρα, για το καθαρό έδαφος, για μια προστασία πλήρη του περιβάλλοντος. Ε, θα ήθελα εδώ να αναφέρω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Γαλλικία με τις πυρκαγιές. πυρκαγιές φυσικά υποβαθμίζουν και την ποιότητα του αέρα. Και έχουμε και ένα πρόβλημα τον ευκάλυπτο που δημιουργούνται προβλήματα με την καλλιέργεια και στον φτιάχνονται Κομποστέλα αύριο και την επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά θα συζητηθούν σε μια ε, συζήτηση που θα οργανώσουμε και για το νερό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μαρζή για δύο λεπτά θα μιλήσει εξ τις ομάδες του. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρέπει να ακούσουμε τους νέους ε, της Ευρώπης ε, και του κόσμου που είναι η ελπίδα που θα μας σώσει τώρα που όλα επιδεινώνονται για το κλίμα. Πρέπει να ακούσουμε τους νέους που έχουν επίγνωση και που λένε στους ε, ισχυρούς και στους ενήλικες ότι τώρα πρέπει να αναλάβουν δράση για το κλίμα, για τα διάφορα είδη φυτών και ζώων, για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον στον πλανήτη. Οι νέοι μας λένε ότι δεν είναι πλέον επίγον να περιμένουμε, αλλά είναι επίγον να αναλάβουμε δράση και να τα αλλάξουμε όλα άρδινα διότι αυτό που συμβαίνει ιστορικό. Βλέπουμε την νεολαία να μας καθοδηγεί και να μας δείχνει το δρόμο. Η νεολαία είναι αυτή που δεν θέλει να παρασυρθεί σε αυτό το τυφλό ε, δρόμο, σε, αυτή την, σε αυτό τον τυφλό αγώνα ταχύτητας ε, που τον οδηγούν τυφλοί και που μας οδηγούν όλους ε, στον κρεμό. Οι νέοι μας τα έχουν καταλάβει όλα. Έχει χτυπήσει το καμπανάκι για την για την οικολογική δικαιοσύνη και την κλιματική δικαιοσύνη. Ένα, δύο, τρει βαθμοί άξονα Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ουρμπάν Κρέσπο είναι ο επόμενο. Ευχαριστώ πολύ Καταγγέλουν οι νέοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στο ύψο των προκλήσεων τη κλιματική αλλαγή και είναι σαφέ το μήνυμά του. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κατεπίγουσα κατάσταση για το κλίμα. Χρειάζεται δραστική περικοπή, μείωση των αερίων θερμοκηπίου, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Με τη δική μα την ψήφο θέλουμε να δείξουμε ότι στηρίζουμε του νέου που κινητοποιούνται για να υπερασπιστούν ένα αξιοπρεπέ μέλλον και να καταγγείλουν ε, την υποκρισία και την αδράνεια, την απραξία μια Ευρωπαϊκής Ένωση, απέναντι στο, στην πρόκληση κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε κυβερνήσει και θεσμούς που θα δείξουν σθένο, ε, που θα σταματήσουν τι ε, πολιτικές που σφετερίζονται και λαιλατούν και τους φυσικούς πόρους. Πρέπει να βελτιώσουμε τα μέτρα, πρέπει να προωθήσουμε την ενεργειακή μετάβαση, την οικονομική και κοινωνική οικολογική μετάβαση γιατί δεν μπορεί κανείς να αιτιολογήσει λόγω αύξησης των κερδών την λαιλασία του μέλλοντός μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ουρμπαν Κρέσπο, συνάδελφος Κούμπου Λανάτρη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Επιτροπή έχει προτείνει δύο πιθανά σενάρια για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050 το αργότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι δεσμεύσεις μας ε, θα πρέπει να ε, επέλθουν πριν από το 2020. Έχουμε το θεματολόγιο του 2030 ε, με 55% περικοπές των εκπομπών σε σχέση με το 2019. Πολλά κράτη-μέλη και ελπίζω και η χώρα μου η Φινλανδία που θα αναλάβει την Προεδρία τον Ιούλιο, ελπίζω ότι θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν πλειοψηφία στο Συμβούλιο, ούτως ώστε να δράσουμε ταχαίως. Και η νέα Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό να εργάζεται, κάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις για να διασφαλίσει ότι θα επιτύχουμε τους στόχους μας. τα παιδιά του σχολείου στην Φιλανδία διαδηλώνουν κατά της κλιματικής αλλαγή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κουμπούλα ο κύριος Πιοτρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Στο ψήφισμά μας, το ψήφισμα του ECR, σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για λιγότερο από 10% των παγκοσμίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Δεν μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων χωρίς να ληφθούν υπόψη και δραστηριότητε άλλων οικονομιών. Δεν μιλάμε ούτε για τους δικούς μας πόρους και τη δική μας ενεργειακή ασφάλεια. Παραδείγματος χάρη, μπορούμε να υποστηρίξουμε τον τεχνολογία για καθαρό άνθρακα που θα μας επιτρέψει να, χρησιμοποιήσουμε αντιμετωπίσουμε το υδρογόνο σαν μια καθαρή πηγή ενέργειας. Γι' αυτό καταψήφισα. Ευχαριστούμε κύριε Πιοτρόφσκι. Ο κύριος Σόσνιρτς. Ευχαριστώ. Η οικονομία με μηδενικέ εκπομπέ. είναι πολιτικό φάντασμα, φαντασία. Ποτέ δεν υπήρξε, δεν θα υπάρξει. Δεν έχουμε την τεχνολογία, ανεξάρτητα από αυτά που λέτε εσείς στην αριστερά. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα, μπορείτε να γράφετε συγγράμματα, Μπορείτε να γράψετε τα πάντα επί χάρτου, αλλά δεν θα αλλάξει την πραγματικότητα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η γη θα, ότι θα στρέφεται προ την άλλη κατεύθυνση, θα περιστρέφεται την άλλη κατεύθυνση αύριο. Αυτό δεν θα αλλάξει όμως την πραγματικότητα και την περιστροφή της γης. Επίσης, για το κλίμα και τι εκπομπέ, αν είσαστε τόσο μακριά από το ρεαλισμό στους στόχους, δεν πετύχετε τίποτα. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να βλάψετε την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αυτό είναι τυπική συμπεριφορά των σοσιαλιστών. Δεν Θα υπάρξει πρόοδο όμω για το κλίμα. Είτε έχει δίκιο για την πολιτική, για το κλίμα, για το μέλλον. Είμαι εδώ για ένα χρόνο. Ψηφίσαμε χιλιάδε αλλαγέ για την αλλαγή του κλίματο. Δεν είναι κάτι προβλέψιμο, δεν είναι σταθερό. Κανεί δεν μπορεί να επενδύσει και να είναι σίγουρο ότι δεν θα αλλάξει ρότα στην πολιτική του Κοινοβουλίου αύριο. Ευχαριστούμε κύριε Σόσνιερτς. Η κυρία Ward. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν γνωρίζει σύνορα. Στην Ευρώπη έχουμε τεράστια ευθύνη έναντι του υπολείπου κόσμου. Ιδίω έναντι αυτών που ζουν σε ευάλωτε χώρε. Επίση, έχουμε μια τεράστια ευθύνη για τον πλανήτη που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Υποστηρίζουμε τους νέους, εμπνευσμένοι από την Κρέτα Thunberg που συμμετέχει στις απεργίες της Παρασκευής που κάνουν τα παιδιά του σχολείου, οι μαθητές του σχολείου. Ελπίζουμε ότι η πολυμορφία της γνώσης θα συνεχιστεί. Ελπίζω να ακούσουμε αυτά τα μηνύματα στα πλαίσια τη ε, διακοινοβουλευτική ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού λυπόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε που ε, δεν δίνουμε σε αυτού του νέου που ανησυχούν για το μέλλον τα μέσα για να προωθήσουν αυτή την πολιτική. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σα σε μια ομάδα νέων στη δική μου εκλογική περιφέρεια σε ένα σχολείο στο Άκρινγκτον που ονομάζεται Οικολογική Ομάδα και ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρουσιάσουν τι ιδέε που έχουν για το περιβάλλον. Αυτοί είναι οι ηγέτε του μέλλοντο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα το κοινό για την αλλαγή του κλίματος, διότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο εκείνο στο οποίο μόνιμα θα έχουμε τα προβλήματα, θα αλλάξουμε τη γη. Δεν πρέπει να λησμονούμε και τα προφανή σημάδια τα πρόσφατα γεγονότα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά τους σπόρους και αυτή χρειάζεται μια, μια κοινή προσπάθεια στη βιομηχανία, στη γεωργία, να υπάρξει συντονισμό και να είναι πιο υπεύθυνοι και οι καταναλωτέ και να έχουν επίγνωση των προβλημάτων. Χρειάζονται τεχνολογικά βήματα προόδου και με αυτά τα βήματα μπορούμε να βρούμε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δεν έχει νόημα να διονύζεται η χρήση των ορυκτών καυσίμων. Για αυτή τη μετάβαση χρειαζόμαστε μια μεγάλη προσπάθεια και μια πολιτική συνένεση σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνηση, σε εθνικό και ανώτερο επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια μετάβαση προ μια βιώσιμη οικονομία, να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε αυτό το στόχο. Διαφορετικά, μόνο διακοσμητική φύσεω ε, μέτρα θα λαμβάνονται που θα χρησιμοποιούνται ε, ε, προ όφελο ελαχίστων. Ελπίζω να μην είναι αργά και να μην χάνουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και για αυτό το θέμα η διαδικασία των επεξηγήσεων ψήφου και πηγαίνουμε σε επεξηγήσει ψήφου για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΑ, συστάσει. Κυρία Κέρτον Ντάρλινγκ δεν είναι εδώ, άρα ο κύριος Μορέλ θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. σε Ευρωπαϊκές Ένωσης φοβούνται περισσότερο ε, τα tweet του Ντόναλτ Τραμπ από την οργή των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι το ερώτημα. Όταν βλέπει κανείς ότι τρέχεται, η Κομισιόν τρέχει να ε, διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με τις είπα που τι κάνουν, αυξάνουν ε, τους δασμού τους και δεν μας επιτρέπουν ε, να, έχουμε συναλλαγές με το ένα. Δεν σέβονται τη Συμφωνία των Παρίσιων. Και ποια είναι τα αντίπεινα που προτείνει για την Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους ξανααναστήσει με τις ίδιες ανησυχίε για την εισαγωγή φυσικού αερίου ε, και όλα τα άλλα προβλήματα παραμένουν, αλλά την συντάφτα που την απορρίψαμε, τώρα θέλω να μας την ξαναβάλουν από το παράθυρο. Αυτή είναι η απάντηση που προσπαθούν να φέρουν και θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις. Ευχαριστώ κύριε Μορέλ. Ολοκληρώθηκαν εδώ οι επεξηγήσεις ψήφου για τις ε, εμπορικές ε, συνομιλίε με τη ΣΥΠΑ και τώρα πάμε στην κατάσταση για την Νικαράγουα. Το κύριο Ορμπάν Κρέσπο. Α, είναι αλλού. Εκεί. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάνω από 76 νεκροί, 700 τραυματίες και χιλιάδες ήταν κρατήσεις μετά τις διαδηλώσεις ε, στην Ικαράβα. Ζητούμε ανεξάρτητη έρευνα ώστε να δώσουν ε, το, ε, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη οι θύτες, οι δράστες. Θέλουμε ένα διάλογο που θα επιτρέψει να ακουστούν όλες οι φωνές και να βρεθεί μια λύση με διάλογο που θα περνάει από την ελευθερία, την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, τον αφοπλισμό των παραστατιωτικών ομάδων και την εξασφάλιση των βασικών κοινωνικών ελευθεριών όπως είναι το συνεταιρίζεσθε, η συμμετοχή η ελευθερία έκφρασης κτλ. Όπως μας έδειξε η ιστορία της Νικαράγουας ε, θα πρέπει με τη διαμαρτυρία ουσιαστικά να ε, δοθεί μια όθηση για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Το μέλλον της Νικαράγουας αυτό που πρέπει να το αποφασίσουν είναι σαφές ότι είναι οι κάτοικοι της χώρας πλήρως ε, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, χωρίς καμία καταπίεση και όλοι οι εξόριστοι επίσης πρέπει να μπορούν να γυρίσουν ελεύθερα πίσω. Ευχαριστούμε κύριε Ουρμπάν Κρέσπο. Ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώθηκαν οι επεξήγησεις ψήφου για την Ικαράγουα και τώρα για την έκθεση της κυρίας Θεοχάρους και του κυρίου Γκάμπους για την στρατηγική έκθεση για την εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρία Μάγια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια βασική αρχή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη είναι ότι είναι καθολική και ότι πρέπει όλε οι χώρε να βοηθήσουν και στη χώρα του αλλά και στο εξωτερικό ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι. Δυστυχώ νομίζω ότι πρόκειται να αποτύχουμε. Έχω μαζί μου ένα κατάλογο για ψώνια που έχει κονσέρβα, έχει σάλτσα για μακαρόνια. Ε, ε, έχουμε αυτά τα οποία ψωνίζει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ. Εξετάσαμε ε, το σύστημα το, του τι αγοράζουν οι καταναλωτές και βλέπουμε ότι η Βρετανία δεν είχε τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτό τον κατάλογο. Είναι λυπηρό ότι ε, η πείνα ε, συνεχίζει να μαστίζει τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ε, το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας. Έχει φτάσει καιρό να δράσουμε υπέρ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστούμε κυρία Μάγερ και κλείνουμε με την κυρία Βόρντ. Η στοχή βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια δέσμευση. Θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο μα για τι μελλοντικέ γενιέ, να μπορούν να ζήσουν σε αρμονία και ειρήνη. Σε ένα πιο ισότιμο κόσμο, χωρί φτώχεια και με σεβασμό για το περιβάλλον. Και 17 στόχοι που εντοπίζουν θέματα κατεπήγοντα πρέπει να λυθούν, πρέπει να προωθηθούν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει την νομιμότητα αυτών των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη σαν στόχο τη οικονομία. Οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να χέρι με χέρι και δεν θα πρέπει να ερμηνεύουμε την ανάπτυξη μόνο στα πλαίσια ΑΕΠ. Κυρίω όσον αφορά το στόχο 4, την ποιότητα τη παιδεία, καταδικάζω τη ζημιά που έχει επιβάλει λιτότητα στα συστήματα παιδεία. Ποιοτική παιδεία είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, η παιδεία είναι ένα από του τομεί που έχει πληγεί χειρότερα από τα μέτρα λιτότητα. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνονται στην ευρύτερη στρατηγική για τι χώρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, η αποχώρηση του νομού Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στην τελική κυβέρνηση να αγνοήσει τι τρέχουσε οικονομικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούν σημαντικέ επενδύσει σε δημόσιε υπηρεσίε συμπεριλαμβανομένη τη παιδεία. Ευχαριστούμε κυρία Ward. Ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση της κυρίας Θεοχάρους και του κυρίου Γκαμπούς, οπότε ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι της σημερινής συνεδρίασης. Σας εύχομαι καλή όρεξη και διακόπτουμε μέχρι τις 3.